Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα σχετικά κείμενα είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Επομένως, εγκρίνονται τα πρακτικά. Και προχωρούμε στη δήλωση Συμβουλίου και Επιτροπής με θέμα την ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες. και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες. Πολύ σημαντικό σημείο που δυστυχώς ε, μας απασχολεί όλο και πιο έντονα. Εξού και έχουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ακούσουμε καταρχάς λοιπόν την εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την κυρία Τουποράινεν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, έχουν περάσει εδώ τέσσερι μήνε από τότε που έγιναν οι ευρωεκλογέ ε, σε συνδυασμό σε αρκετά κράτη-μέλη με άλλε εκλογέ δεν εντοπίστηκε κάποια μείζων ε, εξτρατεία ξένη παρέμβαση, αλλά και έρευνε και πανεπιστημικοί μίλησαν ε, για κάποιε κακόβουλε απόπειρε παρέμβαση. Ε, και γι' αυτό πρέπει πάντοτε να είμαστε προετοιμασμένοι και να κάνουμε συνεχεί προσπάθειε για αύξηση τη ευαισθητοποίηση και τη ετοιμότητα. Πρέπει επίση να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα τη δημοκρατία μα στι κυβερνοαπειλέ μεταξύ αυτών και κατά τη παραπληροφόρηση. Αυτό είναι και μια προτεραιότητα τη ε, Φιλανδική Προεδρία, μακροπρόθεσμε προσπάθειε δηλαδή, για να είναι πιο ανθεκτικά τα συστήματα των δημοκρατικών κοινωνιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε υβριδικέ απειλέ ε, και παραπληροφόρηση που αποδυναμώνουν ε, το περιβάλλον ασφάλεια είναι ανησυχητικό ο χαρακτήρα των απειλών και αυξάνεται το επίπεδο κακόβουλων επιθέσεων. Αυτό σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνητή νοημοσύνη και, ε, και των τεχνικών συγκέντρωση δεδομένων απαιτεί τη συνεχή ευαισθητοποίηση, εγρήγορση και ε, απάντηση. Θεωρούμε ότι είναι θετικό ε, το εγχείρημα που ανέλαβε η Κομισιόν να μελετήσει δηλαδή σε βάθο την εφαρμογή των δεσμεύσεων ε, των επιγραμμικών πλατφορμών και άλλων συμβαλωμένων ε, του κώδικα καλή πρακτική. Το Συμβούλιο παρακολουθεί την εκτέλεση και το έργο των ομάδων εργασία και θα εξετάσουμε τι προτινόμενε δράσει από την Κομισιόν. Αυτό θα γίνει στα τέλη του έτου. Πριν τα τέλη του έτους αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκθεση σε σχέση με τις 29 ευρωεκλογέ με ιδιαίτερη προσοχή στην ετοιμότητα, στην αθεκτικότητα για την αντιμετώπιση παρεμβάσεων στις εκλογικές διαδικασίες και πολύ ενδιαφέρον ιδιαίτερα θα είναι να ακούσουμε τις σκέψεις της Κομισιόν για ενδεχόμενες περαιτέρω πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει. Αποδίδουμε μέγιστη σημασία στο ζήτημα αυτό, ε, όπως επανειλημμένως έχει τονίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άλλωστε, στο πλαίσιο δε και του νέου στρατηγικού θεματολογίου. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ε, το καθένα και στο πλαίσιο τη δημοκρατική διαδικασία. Σίγουρα απαιτούνται συντονισμένε προσπάθειε από την Ένωση και τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα όμω και από την κοινωνία των πολιτών και από τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να δώσουμε μια συνεκτική απάντηση, εστιάζοντας και στην εξωτερική και στην εσωτερική διάσταση των απειλών αυτών. Μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου το Μάρτιο για την εξασφάλιση δίκαιων και ελεύθερων εκλογών, έχουμε το εκλογικό πακέτο και την δάεσμη μέτρων από την Κομισιόν. Έκτοτε έχουν γίνει πολλά και από τα θεσμικά όργανα και σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών μελών. Υπήρχαν τακτικές συναντήσεις του δικτύου ε, για την παρακολούθηση των εκλογικών διαδικασιών. Εντοπίστηκαν οι απειλές, έχουμε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίηση, εθνικού συνδέσμους για την ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά την παραπληροφόρηση. Επίσης, στρατηγική ενημέρωση, ανταλλαγή πρακτικών, ενίσχυση του οικοσυστήματος των ΜΜΕ με τη διευκόλυνση δικτύων με ανεξάρτητους ε, επιτήρητες και ελεγκτές, ε, ο εγγραμματισμός των μέσων ε, μαζικής ενημέρωσης και άλλες δραστηριότητες, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία της εκαιρότητας των εκλογικών διαδικασιών, αλλά σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να αξιολογήσουμε τις υπερδικές επίσης απειλές και να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την κοινότητα των εκλογικών συστημάτων εστιάζοντα ε, και στο πώ ε, οι κοινωνικέ πλατφόρμε που ε, λειτουργούν στο δίκτυο εφαρμόζουν τον κώδικα καλή πρακτική, όπω είπα. Άρα, έχουμε μεν κάνει πολλά ήδη. Πρέπει να κάνουμε και άλλα. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, σε συνέχεια των προσπαθειών αυτών, η Ρουμανική Προεδρία είχε προετοιμάσει μια έκθεση στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση τη παραπληροφόρηση και για την άρληση διδαγμάτων από τι ευρωεκλογέ. Σε συνέχεια αυτού του έργου, μια από τι βασικέ προτεραιότητε τη δική μα Προεδρία είναι να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα της, ε, των κοινωνιών μας ε, από απειλές εξωτερικές. Αναλαμβάνοντα ολιστική δράση και προσέγγιση όλους τους τομείς για να έχουμε ε, μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλω να τονίσω πως όλο αυτό το έργο για την προστασία των ανοιχτών δημοκρατικών κοινωνιών μας θα πρέπει να γίνεται σε πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών μα. Και εδώ περιλαμβάνεται φυσικά και ελευθερία έκφραση. Σε αυτό το πλαίσιο η Προεδρία μα δίνει μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ένωσης για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και για τη μεγαλύτερη αντοχή, ανθεκτικότητα ε, των ευρωπαϊκών συστημάτων, των κρατών μελών. Των, ε, συστημάτων, ε, των κρατών μελών. Ήδη υπάρχει και η οριζόντια εντολή μιας νέας ομάδας εργασίας η οποία συγκροτήθηκε και έχει κάνει και την πρώτη τη συνάντηση. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε επίσης να αναπτύσσουμε εταιρικέ σχέσεις. Η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστεία Αντιμετώπιση των Ευρωπαϊκών Απειλών με έδρα το Ελσίνκι. Και αυτό έχει ω στόχο την ενίσχυση τη εργασία στον τομέα αυτό. Οι στρατηγικέ παραπληροφόρε από ξένα κράτη αλλά και μη κρατικού φορεί ε, υπερβαίνουν τα σύνορα τη Ένωση. Άρα απαιτείται συμπληρωματικότητα, συμπληρωματική δράση Έχουμε το σχέδιο δράση κατά τη παραπληροφόρηση, το οποίο αναφέρει πόσο σημαντικό είναι να ε, οργανώσουμε τη συνεργασία μα με του γείτονε από ε, την Ανατολική, την Νότια ε, γειτονία και τα Βαλκάνια κτλ. Θέλουμε να αναπτύξουμε επίση τι δεξιότητε σχετικέ. Από κοινού πρέπει να δράσουμε με συγκροτημένο, συντονισμένο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές προστασία των εκλογών είναι στο επίκεντρο της επέρασπισης των ευρωπαϊκών αξιών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας κυρίες και κύριοι. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα ε, έχουμε δύο προσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί μας, την κυρία Γιούροβα και τον κύριο Κίνγκ. Θα ξεκινήσει η Επίτροπος Γιούροβα. Παρακαλώ. Mr. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ο σεβασμό τη δημοκρατία, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου είναι βασικέ αξίε που ενώνουν όλου μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει όμω να θεωρούνται δεδομένε. Η πρόεδρο Φόντεν Λάιεν ανακοίνωσε ότι η προστασία των δημοκρατικών αξιών θα είναι προτεραιότητα τη Επιτροπή. Υπογράμμισε ότι τα δημοκρατικά μα συστήματα διαρκώ δέχονται ε, αυξανόμενε επιθέσει από αυτού που θέλουν να μα διαιρέσουν και να μα αποσταθεροποιήσουν. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προστατευτούμε από εξωτερικές επιρροές. Η διόγκωση της παραφληροπόρησης και η πολιτικές των σκοτεινών ε, διαδικτύων και προεκτάσεων διαστρεβλώνουν τον ε, δημόσιο διάλογο. Ε, ξένοι παράγοντες τα εκμεταλλεύονται αυτά για να επηρεάσουν την χάραξη πολιτικής σε τομείς όπως οι κλιματικές αλλαγές, η μετανάστευση, η δημόσια υγεία, τα οικονομικά. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί εφόσον δεν βασιστούμε σε επιστημονικά στοιχεία ε, αντικειμενικά και ακριβή. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση εδώ χρειάζεται και δεν μπορεί να περιοριστούμε στις ομονωμένες αντιδράσεις των κρατών μελών. Θα πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε όλες τις απειλές. Αυτό που επηρεάζει ένα κατος μπορεί να είναι πλήγμα για όλους. Γι' αυτό η δέσμη μέτρων που προτείναμε από το Σεπτέμβριο του 2018 συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένε δράσει για την υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών ώστε να διοργανώνουν ε, ένομε εκλογέ και να καταπολεμηθεί η παραπληροφόρηση. Στα πλαίσια του πακέτου αυτού έχει οργανώσει εθνικά εκλογικά δίκτυα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που μπορεί να απειλούν τη δημοκρατική διαδικασία. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών έχει υποστηριχθεί από το νέο δίκτυο συνεργασία για τι εκλογές, νέο ευρωπαϊκό δίκτυο που επιτρέπει την ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών και τη δημιουργία επιχειρησιακών ε, συνδέσμων ε, για να είναι σε επαφή τα κράτη-μέλη. Έχουν ήδη συναντηθεί εκπρόσωποι του δικτύου τέσσερις φορές πριν από εκλογές και η πρώτη συνάντηση ε, έγινε μετά από τη διεξαγωγή εκλογών με εκπροσώπους από τα εθνικά δίκτυα που είχαν επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και με συμμετοχή άλλων ε, θεσμικών οργάνων μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και τη κοινωνία των πολιτών. Αυτέ οι δραστηριότητε κάλυψαν όλε τι διαστάσει αυτού του περίπλοκου χώρου, από την ε, συνομιλία και την ενημέρωση των πολιτών, τι πλατφόρμες μέχρι τη χαρτογράφηση των νομικών εργαλείων που υπάρχουν ε, και την χρηματοδότηση από ξένες πηγέ. Επίση, υπήρχε μία προσπάθεια αναβάθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορούν να αποτιμήσουν τα κράτη-μέλη και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά του απέναντι σε κυβερνοεπιθέσει. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, εμπλακεί ε, στην λειτουργία του δικτύου και εκφράσει την επιθυμία τους και για τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά δίκτυα να συνεχίσουν με αμύωτο ρυθμό τι προσπάθειέ του εν των ευρωεκλογών αρχικά και προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να ε, έχουν καλύτερη ανθεκτικότητα στην διεξαγωγή των εκλογών και στα εκλογικά του συστήματα. Μετά τις πρόσφατες ευρωεκλογέ, τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. Ε, η συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση επέτρεψε να έχουμε καλύτερη προετοιμασία για να προλάβουμε την χειραγώγηση και τη διαστρέβλωση καθώς και την παραπληροφόρηση. Βλέπουμε μετά τις πρόσφατες εκλογές ότι η διεξοδική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των εμπειριών των ευρωεκλογών μπορεί να είναι κάτι το πολύ χρήσιμο. Έχουμε και πολύτιμού εταίρου σε διαφορετικά φόρα, όπως το G7 και το ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή και εξωευρωπαϊκών κρατών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία διάθεση συνολικά ε, στα δημοκρατικά κράτη να προστατεύσουν και να κάνουν ανθεκτικές τις δημοκρατικές τους διαδικασίες. Η διεθνής συνεργασία μας διαβεβαιώνει ότι τα εργαλεία, τα όπλα και οι δυνατότητε των μεμονωμένων εταίρων μπορούν να συνενωθούν εδώ για να προστατεύσουμε τα θεμέλια δικαιώματα, ιδίως την ελευθερία της έκφραση και του συνασπίζεστε. Εδώ λοιπόν, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος Φόντεν Λάιεν, εφόσον εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο, η Επιτροπή και η Επιτροπή, θα μπορέσουμε να εκδιπλώσουμε ένα πλήρες φάσμα εργαλείων και όπλων για την σωστή και ένομη διεξαγωγή των εκλογών σε όλες τις περιπτώσεις στην Ευρώπη. Εάν λοιπόν επιβεβαιωθεί και η δική μου θητεία, θα φροντίσω να κάνω ό,τι μπορώ για να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των δημοκρατικών μας συστημάτων, να καταπολεμήσουμε την κακή πληροφόρηση και την παραπληροφόρηση. Αυτά είναι απόλυτες ανάγκες στην κατάσταση που έχουμε περιέλθει σήμερα σήμερα. Επίσης, η, δημοκρα... ελευθερία της έκφρασης και η ελευθεροτυπία σε ένα τοπίο ε, πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης πρέπει να καλλιεργηθούν και να προστατευτούν από την επόμενη Επιτροπή. Με όλες αυτές τις προσπάθειες και εφόσον επιβεβαιωθώ στη μελλοντική μου θητεία από το σώμα θα συνεργαστώ στενά με το Ευρωκοινοβούλιο, με προσώπους των 100 μελών της κοινωνίας των πολιτών και των ενδιαφερομένων για να καλλιεργήσουμε περαιτέρω την ε, δημοκρατία όπως τη γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος Κίνγκ. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφε, εγώ θα μιλήσω περισσότερο για τις ε, προκλήσεις παραπληροφόρησης και όπως ήδη ακούσαμε, δυστυχώς στις τελευταίες ε, ευρωεκλογές δεν αντιμετωπίσαμε μεν μία μαζική επίθεση παραπληροφόρησης, αλλά δεν ήταν ελεύθερες από προσπάθειες παραπληροφόρησης αυτές οι εκλογές. Έχουμε μυριάδες εκθέσεις από όλη την Ευρώπη για τα διαφορετικά είδη της παραπληροφόρησης. Και μπορώ να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Από κάποιο άλλο κράτος μέλος, από τη Γερμανία για παράδειγμα, έχουμε εκθέσεις που δείχνουν πως online προώθησε ενός από τα γερμανικά κόμματα ήταν το 86% όλων των κομματικών δραστηριοτήτων στο Facebook. Είχαν τέσσερις φορές περισσότερα σχόλια, έξι φορές παραπάνω έκαναν share από όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα μαζί. Και πολλά από αυτά τα like και τα share προέρχεται από ένα κόμβο 80.000 ύποπτων ε, λογαριασμών με τυχαία ε, μικρά ονόματα και επίθετα δηλαδή ε, χιλιάδες ε, πληροφορίες. Μιλάμε δηλαδή για ένα κύμα αυτοματοποιημένης προπαγάνδας και παραπληροφόρησης που αποτελεί κομμάτι της καθημερινής μας πολιτικής ε, πραγματικότητας. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε αυτούς τους λογαριασμούς, τους τυχαίους, με συνδυασμό τυχαίο πρώτου με μικρού ονόματος και επιθέτου που αποτελούνται και τα δύο από δύο γράμματα, τι θα κάνουμε, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις ε, των κακόβουλων ε, ατόμων που επιτίθονται εναντίον μας με σκοπό την παραπληροφόρηση. Πώς θα αντέξουμε. Πώς θα μειώσουμε τις επιπτώσεις αυτής της παραπληροφόρησης. Μαζί με τα κράτη-μέλη λοιπόν και με έναν αριθμό από άλλους εταίρους μας έχουμε εργαστεί προς τέσσερις κατευθύνσεις. Καταρχήν, έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μπορούν και να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τις κακόβουλες επιθέσεις. Αυτό τον ε, μηχανισμό θέλουμε τον ενισχύσουμε. Περνάμε μια ε, διαδικασία διαβουλεύσεων αυτή τη στιγμή για το πώς γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και να δούμε τι μπορούν να κάνουν τα θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη και οι πλατφόρμες αυτές, όπως επίσης και η κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την προσπάθεια που γίνεται για την έρευνα και την ανάλυση των προσπαθειών παραπληροφόρηση. Τα τελευταία δύο χρόνια, και αυτό είναι το δεύτερο, έχουμε κινητοποιήσει μια κοινότητα ε, ερευνητών, Κοινωνία των πολιτών και ε, ελεγκτών αλήθειας επαληθευτές δηλαδή, που ε, ελέγχουν τις πληροφορίες για να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε τις αποκρίσεις μας και πώς θα ενισχύσουμε όσα κάνουν εκεί. Για τούτο το σκοπό θα έχουμε μια καινούρια online πλατφόρμα στην Ευρώπη, όπου αυτές οι οργανώσεις που ε, επαληθεύουν, οι 38 σε 17 κράτη-μέλη, θα συνεργαστούν πιο πολύ με χρηματοδότηση ε, από το ε, Connecting Europe, ε, το μηχανισμό Connecting Europe. Αλλά θέλουμε για να πετύχουμε να μας βοηθήσουν και οι πλατφόρμες, να έχουμε ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα για αυτούς τους ελεγχόμενους και ελεγμένους επαληθευτές έτσι ώστε μαζί να ξεκλειδώσουμε την καλύτερη απόκριση και πάντα εξασφαλίζοντας πως τα ε, διάφορα, ε, οι διάφοροι κανόνες διοντολογίας και ηθικής γίνονται σεβαστοί. Τώρα, Θέλω να σχολιάσω και το τρίτο σημείο. Εμείς τις μεγάλες πλατφόρμες τις πιέσαμε και αυτή τη στιγμή έχουν υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας για την παραπληροφόρηση. Αυτό έκλεισε πέρσι το Σεπτέμβριο και η αρχική Facebook, Google, Twitter, Mozilla και κάποια εμπορικά επιμελητήρια, διαφημιστές κτλ. έχουν ε, υπογράψει και πρόσφατα είχαμε και τη Microsoft που ε, υπέγραψε και αυτή. Είναι λοιπόν μια σειρά δεσμεύσεων, 15 δεσμεύσεις από πολύ ισχυρού παίκτες και εμείς παρακολουθούμε την απόδοσή τους να δούμε αν πετυχαίνουν αυτές τις δεσμεύσεις και σε ποιο βαθμό. Και πρέπει να σας πω πως μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου ε, ε, να Θα δούμε και την αυτοαξιολόγηση που θα κάνουν τώρα όπου να είναι γιατί έχουν αναλάβει μαζί με τρίτους ε, αξιολογητές να παραδώσουν και μία αξιολόγηση από τρίτους μέχρι μέσα Οκτωβρίου των επιδόσεών τους μέσω αυτών των δεσμεύσεων. Εμείς θα κάνουμε μία επισκόπηση του πού βρισκόμαστε και το πώς πάει η εφαρμογή του ε, κώδικα αυτού μέχρι τέλη Οκτωβρίου και πλήρη αξιολόγηση ως ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε αρχή της επόμενης χρονιάς. Αφού περάσουν και διαβολεύσεις με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, με τα κράτη-μέλη, τους ρυθμιστές ε, για τα οπτικοακουστικά στην Ευρώπη και όπως είπε και η Επίτροπος ε, Γιούρβα και η Επίτροπος Γκαμπριέλ, εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση. Ακόμα και ρυθμιστική δράση. Είχαμε μία σειρά από κανονιστικές και νομοθετικές προτάσεις από τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ε, μία ε, λευκή βίβλο για, ε, την, την online πληροφόρηση. Έχει κάτι αντίστοιχο κάνει η Γαλλία. Ζητάμε λοιπόν τα κράτη-μέλη που μπορούν να μας βοηθήσουν. Τώρα, τελευταίο σημείο. Θέλουμε να χειραφετήσουμε τους πολίτες μας κάνοντάς τους πιο εξοικειωμένους με τα μίντια για να ξέρουν ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, των δικών μας πολιτικών έτσι ώστε να ενισχυθούν οι πολίτες μας και να μην ε, πέφτουν θύματα αυτής της παραπληροφόρησης, της κακόβουλης και επιθετικής παραπληροφόρησης. Έχουμε λοιπόν καταφέρει αρκετά, πάρα πολλά μένουν ακόμα και όπως και η Επίτροπος ε, Βέρα Γιούροβα, χαίρομαι πάρα πολύ που η επόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι υπόλοιποι και οι επόμενοι επίτροποι υπογραμμίζουν τη σημασία των θεμάτων αυτών και αν επιβεβαιωθεί θα έχουμε και μια συντονισμένη ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση για τις ανθρώπινες ε, ε, διαστάσεις και επιπτώσεις της τεχνητής νοημοθένης ως νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επίσης και το θέμα της ευθύνης για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Αυτές οι προσπάθειες, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα που έχουμε συζητήσει, είναι κομβικά κομβικές, με συγχωρείτε, για να έχουμε ένα ψηφιακό μέλλον το οποίο θα είναι ασφαλές και θετικό για όλους τους πολίτες. Danke auch für die äh, Ευχαριστώ πολύ και για τις πληρέστατες ε, αυτές περιεκτικές ομιλίες. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές. Πρώτος ε, ο κύριος Τομπέ από το ΕΛΚ. Εκτός μικροφώνου. Now? Yeah. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητό Συμβούλιο, αγαπητή Επιτροπή και αξιότιμοι βουλευτές. Αυτή η συζήτηση αφορά θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, το κράτος δικαίου, την ελευθερία και δημοκρατικές εκλογές. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταθέσει μετά τη συζήτηση ένα πολύ ισχυρό ε, ψήφισμα. Εμείς ε, ως Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστούμε ε, τις δημοκρατικές ελεύθερες εκλογές χωρίς παρέμβαση ξένων κρατών. Δυστυχώς όμως σήμερα δεν έχει έτσι κατάσταση στην Ευρώπη και νομίζω ότι είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην φοβηθεί. Πρέπει να τα πει ξεκάθαρα τα πράγματα. Ιδίω η Ρωσία είναι γνωστό αυτό διεξάγει έναν πόλεμο πληροφόρησης χαμηλής έντασης κατά της Ευρώπης ε, με ολόκληρα ε, δίκτυα και άλλους φορείς ε, που συνεργάζονται με το κράτος. Αλλά αυτό το κάνουν και άλλα πολυτραχικά κράτη όπως είναι το Ιράν, η Βόρεια Κορέα, η Κίνα που προσπαθούν και αυτά τα κράτη να αποδυναμώσουν τη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρώπης και είναι σημαντικό νομίζω να υπερασπιστούμε τις αξίες ε, αν υπάρχει δε επίθεση σε βάρος ε, των δημοκρατικών μας ε, θεσμών, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν συνέπειες. Σε αυτή την ολομέλεια, αγαπητοί φίλοι, σίγουρα διαφωνούμε μεταξύ μας σε πολλά. Αυτό είναι η δημοκρατία όμως. Ε. Δεν είναι κακό να διαφωνεί κανεί με, με τον πλησίον του. Εκεί που συμφωνούμε όμως είναι, είναι στο ότι εάν αφήσουμε τη δημοκρατική δικασία λήψη αποφάσεων να ανοιχτεί στην ξένη παρέμβαση θα απολέσουμε την αυτοδιάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό από κοινού να ε, υιοθετήσουμε ένα κοινό ψήφισμα υπερασπιζόμενοι τις κοινέ μας αξίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κάτι Πύρη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμη επίτροπε, αξιότιμη πρόσωπε τη ε, Δημοτική Προεδρία. Είναι σημαντικέ οι ελεύθερε και δίκαιε εκλογέ στην Ευρώπη και γενικώ. Δυστυχώ είναι κάτι αυτονόητο και δεδομένο πρόσφατα. Κατομμύρια πολιτών ε, εκτέθηκαν σε μαζικές εκστρατείες παραπληροφόρησης ε, λόγω ξένης παρέμβασης. Ε, κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται σαν ευπροηγουμένο επίπεδα και διαστάσεις, απειλώντας στρατικές ποδομές και δεδομένα. Οι εκλογικοί νόμοι, οι νόμοι για τη χρηματοδότηση κομμάτων από τρίτα κράτη έχουν πολλές φορές είτε παρακαμφθεί είτε παραβιαστεί. Τον Ιούλιο υπήρξε το ζήτημα της χρηματοδότησης της ε, εκστρατείας του Ματέου Σαλβίνη από τη Ρωσία. Είναι τελευταία ε, περίπτωση, δεν περιορίζεται στην Ιταλία, στη Ρωσία το θέμα αυτό. Έχουμε πολλές φορές εκφράσει στην προηγούμενη θητεία ε, την αντίρρησή μας σε αυτά τα φαινόμενα παραπληροφόρησης και η Ρουμανική Προεδρία και η προηγούμενη Κομισιόν και χαίρομαι που το ίδιο κάνει και η Φιλανδική Προεδρία. Εμείς ε, καταφέραμε ως ομάδα να, σοσιαλιστών και δημοκρατών να, να βάλουμε την, ε, το θέμα αυτό στην διάταξη με μεγάλη πλειοψηφία. Και υπάρχει υποστήριξη ευρύτατη και για ένα πάρα πολύ ισχυρό ψήφισμα. Χρειαζόμαστε απαντήσεις σοβαρές πώς θα αποφύγουμε ξένη παρέμβαση ε, για, κατά των δημοκρατικών συστημάτων. Είναι μια πρόκληση. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Η ομάδα μας ζητά τη συγκρότηση ειδική κοινοβουλευτική επιτροπής ώστε η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία με πάντοτε ελεύθερες και δίκες εκλογές να παραμείνει κάτι το αυτονόητο και το δεδομένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντουρόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, ξεκινήσατε την ε, ομιλία σας λέγοντας και εκφράσατε και τη χαρά σας ότι πήγαμε καλά στις ευρωεκλογέ και ότι δεν υπήρξαν επιθέσεις τότε. Και εγώ χαίρομαι που οι ευρωεκλογέ πήγαν καλά στην διεξαγωγή τους. Όμω, οι εκλογέ εν γέννη και όλος ιδιαίτερως οι ευρωπαϊκές δεν είναι και το σύνολο των δημοκρατικών διαδικασιών. Αυτά που είπαν ο κύριος Κιν και η κυρία Γιούροβα και το εξήγησαν πολύ σωστά είναι ότι η δημοκρατία μας όπως την αντιλαμβανόμαστε στην Ευρώπη κινδυνεύει, απειλείται και απειλείται από φαινόμενα παραπληροφόρηση που σωστά σημειώσατε και σωστά εντοπίσατε κύριε Επίτροπε. Απειλείται όμως και μέσω της χρηματοδότησης και αυτό αναφέρθηκε και είναι σημαντικό να ακουστεί ξανά μέσω της χρηματοδότησης των ε, πολιτικών κομμάτων απειλείται το θεμέλιο της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι ξένες δυνάμεις που δεν θέλουν το καλό της Ένωσης και ακούστηκε η Ρωσία, αλλά δεν υπάρχει μόνο η Ρωσία, γιατί η Ρωσία το έχουμε ξεκαθαρίσει, έτσι είναι. Αλλά υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που έχουν χρηματοδοτήσει κατά ένα δις ευρώ ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάποιες φορές και κάποια από τα πολιτικά κόμματα που πολλές φορές βρίσκονται στην ε, δεξιά πτέρυγα, την ακροδεξιά πτέρυγα του ημικυκλίου μας και έρχονται από τη Γαλλία και την Ιταλία. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Το ψήφισμα είναι σημαντικό, διότι πρέπει πρώτον να εξοπλιστούμε με τα απαραίτητα μέσα. Τα μέσα με 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και το σημειώσατε κύριε Επίτροπε, ε, σωστά, 3 εκατομμύρια το χρόνο σε σύγκριση με ένα δι δεν είναι τίποτα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και τη δυνατότητα να αναλάβουμε δράση κατά των υπευθύνων τη παραπληροφόρηση. Θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα επικίνδυνα στοιχεία που απειλούν τη δική μα δημοκρατία και τα δικά μα πολιτικά κόμματα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε εργαλεία για να είμαστε τεχνολογικά ανεξάρτητοι. Διότι αν δεν το κάνουμε αυτό, συστηματικά στρεφόμαστε εκτό Ένωση και Ευρώπη για να μπορούμε να ξαναβρούμε να ξαναπάρουμε τον έλεγχο στα χέρια μα. Τα βασικά στοιχεία λοιπόν είναι η ανεξαρτησία μα και η δυνατότητα να αντιδράσουμε. Ευχαριστούμε κύριο κύριος Μπιουτικόφερ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη πρόσωπε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω συγκεκριμένα και ρητά την Φιλανδική πεδρία που παίρνει τόσο σοβαρή υπόψη αυτό το θέμα και να ευχαριστήσω επίση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εντατικά αφιερώνει την προσοχή τη στο θέμα αυτό. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να προστατεύει. Ε, στην πρώτη γραμμή, βέβαια, πρέπει να προστατεύει τι αξίε τη, που σημαίνει να προστατεύει τη δημοκρατία καθώς και την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Και περί αυτού πρόκειται. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής συζήτησης. Δεν θα πρέπει όμως ε, να ε, στρεφόμαστε προς μία μόνο κατεύθυνση και εκεί να στρέφουμε μόνο την προσοχή μας. Δεν υπάρχει μόνο η Ρωσία που αποδεδειγμένα προσπαθεί να παρέμβει, να αναμειχθεί στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Έχουμε και τον κύριο Ερντογάν ε, στην Τουρκία Έχουμε την αυταρχική κινέζικη κυβέρνηση που ε, θέλει να εκμεταλλευτεί την οικονομική εξάρτηση άλλων κρατών. Επίσης έχουμε δραστικούς κύκλους από τη ΣΥΠΑ που ήδη έχουν προσπαθήσει να έχουν επίδραση ε, αρνητική για μας στα εσωτερικά μας ε, ζητήματα. Σίγουρα ε, έχουμε αυτή την αντιπαράθεση ε, μεταξύ των ε, διαφόρων κρατών γιατί εμείς πρέπει να κερδίσουμε αυτή την αντιπαράθεση και να προστατεύσουμε τις αξίες σας. Μας πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να αναμειχθούν αλλά μόνοι μας να φροντίσουμε να μην υπάρχουν ρήγματα. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι όλοι για να, να μην μπορεί κανείς να τα αυτά τα ρήγματα γιατί και αυτό έχει να κάνει με την προστασία της δημοκρατίας και της κοινωνίας κυριαρχία μα Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος είναι ο κύριος Καμπομενόζη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση σήμερα εδώ γίνεται λίγο σουρεαλιστική και εξωπραγματική. Ακούμε στοιχεία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και σκεφτόμαστε αυτούς που ε, δεν ονομάζει κανείς όπως το ΝΑΤΟ και το Ισραήλ. Τι ρόλο μπορεί να έχουν εδώ και κάποιοι παριστάνουν ότι αυτό το παιχνίδι που έχει ήδη συνεχιστεί και ξεκινήσει μάλλον με την ψήφο εμπιστοσύνη προς την κυρία Φόντερ Λάιεν ε, να μην παρενοχληθεί από τίποτα. Υπάρχουν τόσες υποθέσεις δίθεν παραπληροφόρησης που τις διέψευσαν τα ίδια τα μέσα τελικά για να μην συζητήσω καν αυτά που έγιναν στην Ιταλία, τι κατηγορίε που είχαν ε, εκτοξευθεί και τελικά οι έρευνε έδειξαν ότι δεν είχε γίνει τίποτα. Τα δικαστήρια βέβαια θα διαλευκάνουν τι διάφορε υποθέσει, αλλά πίσω από την ανάγκη σα να γίνει αυτή η συζήτηση υπάρχει ίσω η δικαιολογία ότι θέλετε να περιορίσετε την ελευθερία στο διαδίκτυο. Το είδαμε και με τη συζήτηση για την οδηγία για το copyright, για τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. Δεν καταλαβαίνετε πλέον του πολίτε, δεν καταλαβαίνετε του ψηφοφόρου. Ε, πήγε μια πολύ σαφής απόφαση ψηφοφορία για τον Brexit. Σας ευνηδίασε. Και εδώ βλέπετε ότι στο Κοινοβούλιο διπλασιάσαμε τι δυνάμει μα και πάλι ευνηδιαστήκατε. Δεν καταλαβαίνετε τι έγινε. Ε, εδώ κλεισμένοι πίσω από αυτέ τι πόρτε, αυτέ τι αίθουσε, λαμβάνετε και αποφάσει και συζητάτε. Ενώ το 2018 το Κοινοβούλιο έδωσε 33,3 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει και να επηρεάσει ε, εκλογές στην Ευρώπη και λέτε ότι <clears throat> δεν πρέπει μόνο να αναγκάσουμε τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν αλλά να υποχρεωθούν να υποστηρίξουν και το ευρωπαϊκό εγχείρημα και μετά μιλάτε για παρέμβαση στα εσωτερικά των κρατών από άλλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Προκατσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημερίζομαι πλήρως το πνεύμα αυτού του ψηφίσματος. Όμως δεν συμμερίζομαι αυτήν την αιμονική, θα έλεγα ψυχαναγκαστική ε, διάθεση του Κοινοβουλίου να ψάχνει κάποιον εχθρό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και να εξηγηθώ. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να προασπιστούμε την ε, ασφάλεια δημοκρατική, οικονομική και κοινωνική, ε, με καλύτερες υποδομές και με καλύτερα νομοθετικά εργαλεία η επανάσταση που θα φέρει το δίκτυο 5G. Σαφώς πρέπει να τη διαχειριστούμε με ιδιαίτερη προσοχή, διαλέγοντας προσεκτικά τους οικονομικούς ε, συνεργαζομένους μας. Όμως, ε, επί της ουσίας, δεν καταλαβαίνω και δεν καταλαβαίνω και τη μέθοδο που ακολουθούμε. Είναι πιο σημαντικό να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και την προσοχή μας στο πώς οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που είναι αρμόδιοι στα θέματα αυτά θα αναλάβουν δράση, παρά να ε, παραπέουμε στην, ε, στην γεμάτη ψευδεστήσεις αναζήτηση ενός φανταστικού εχθρού. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βόλας, ο κύριος Βόλας. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι προσπαθούν να δυσκολευτούν όλοι να καταλάβουν πως ε, χάνουμε χάνουμε ψηφοφόρους προς την ακραδεξιά. Ε, και πρέπει να σας πω πως έχασε ο Μπέρνι Σάντερς τις εκλογές από τους δημοκρατικούς και όχι από την παραπληροφόρηση. Και το πρόβλημά μας στην Ευρώπη δεν είναι η παραπληροφόρηση από εκτός, αλλά η αυξανόμενη ανισότητα, η ο οικονομικός υπεριολισμός και οι μιλιταριστικοί μας πόλεμοι που δεν επιτρέπουν να ζούμε ειρηνικά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι ΙΠΑ ε, ανακατεύονται στις πολιτικές διαδικασίες ξένων χωρών με βίο τρόπο. Και αν τα συγκρίνουμε με τα όσα συνέβησαν το 2016 στις αμερικανικές εκλογές, ε, στην πραγματικότητα πολύ λίγα έγιναν τότε σε σχέση με τα οχηγούνη στο παρελθόν. Ο κύριος Μύροσλαβ Ραντακόφσκι. Ραντακόφσκι. Δεν είμαι ο Ραντακόφσκι, είμαι Ραντατσόφσκι Μυροσλάβ. Και παρακαλώ πολύ έτσι να λέτε το όνομά μου. Θα ήθελα λοιπόν κι εγώ να μιλήσω για το θέμα της παραπληροφόρωσης και να σας πω πως έχω την εντύπωση πως θέλετε όλοι να φοράμε ε, στολές, να μπούμε σε αεροπλάνα και να επιτεθούμε κατά της Μόσχας. Αυτό δεν είναι σωστό. Ποιος είναι ο εχθρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί είπαμε πως είναι η Ρωσία. Αυτός είναι ο δρόμος προς την κόλαση. Δεν είναι αποδεκτή ευρωπαϊκή ε, τακτική ο Ιάννης Παύλος ο Δεύτερος, ο Σαρλ Ντεγκόλ, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ μίλησαν ε, για την Ευρώπη από τη μάχη στα Ουράλια, ε, τον Ατλαντικό στα Ουράλια. Δεν είναι αποδεκτό να μιλάμε έτσι. Θυμηθείτε την ιστορία. Εκατομμύρια Εβραίοι σκοτώθηκαν, θανατώθηκαν στα στρατόπεδα, όπως επίσης και Σλάβοι. Αυτή ήταν η διαίρεση μεταξύ ε, Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Είναι λανθασμένα όλα αυτά. Δεν θα πρέπει να στρατικοποιούμε τον κόσμο. Πρέπει να λάβουμε τα διδάγματα της ιστορίας. Σας ευχαριστώ και Ράντα Τσόφσκι. Σας ευχαριστώ πολύ που μου μάθατε και τη σωστή προφόρα. Ίσως κάνω λάθα. Ε, τώρα στην κυρία Καρολίνα έτσι τα αντιληφθάζω ότι δεν κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η προσπάθεια επιρροή ε, των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Εκλογών δεν είναι πια κάποιο φαινόμενο το οποίο αποτελεί αντικείμενο μυθιστορημάτων και ταινιών. Είδαμε και στη Γαλλία και στην και σε άλλα σκράτη όπως και στην Αυστρία πρόσφατα που έγινε μια επίθεση στο Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα. 1,3 gigabyte, ε, εκατομμύρια gigabyte αρχεία ε, εκλάπησαν και σίγουρα επηρέασαν τις εκλογέ για το Εθνικό Συμβούλιο. Ε, χρειάζεται γρήγορα να διελευκανθεί η υπόθεση αυτή. Ε, πολιτικοί μας αντίπαλοι αντι, ε, ε, προσπαθούν να διαψεύσουν τη γνησιότητα αυτής της επίθεσης αλλά υπάρχουν ίχνη και αυτά δείχνουν ξένους σερβερ. Εδώ πρέπει να δούμε πρακτικούς και μεθοδεύσεις και υπόλογη υπολογισμούς ε, που δεν στρέφονται μόνο κατά Αυστριακού κόμματος αλλά κατά της δημοκρατίας. Ε, δημιουργεί πρόβλημα στην ελεύθερη διαμόρφωση της κοινή γνώμης, ε, πλήττει τη δημοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ αποφασιστική αυτή η συζήτηση και θεωρώ εξίσου σημαντικό το να υπάρξει και ένα εξίσου ισχυρό ψήφισμα για να δείξουμε ότι δεν θα αφήσουμε εγκληματικά στοιχεία να απειλήσουν τη δημοκρατία, τις θεμελιώδεις αξίες και τον τρόπο ζωή μα στην Ευρώπη. Θα τα προστατεύσουμε όλα αυτά με κάθε σθένος και με κάθε μέσο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες δικαστικές έρευνες και δημοσιογραφικές για την επίδραση και την επιρροή ξένων δυνάμεων, ειδικώ της Ρωσίας, αλλά όχι μόνο, για να ε, διαστρεβλώσουν πολιτικές και δημοσιογραφικές ε, εκστρατείες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Front National το 2014 ή το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία ή τα της Λίγκα στην Ιταλία. Αυτά ε, έχουν διαψευστεί ψευδώς επανειλημμένα ε, και από τον ε, Μαλτέο Σαλβίνη. Θα έπρεπε λοιπόν κάτι να κάνει και ο πρόεδρος της κυβέρνησης Κόντε είναι σαφή η προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα κάποιοι Ευρωπαίοι πολιτικοί κάνουν τους εθνικούς ε, θεματοφύλακες αυτής της ε, δημοκρατική διαδικασία που ποτέ καλούνται να προστατεύσουν, αλλά γίνονται κερκόπορτε για να περάσουν οι ξένε επιδράσει. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τη Λεπέν, το Σαλβίνι να ψεύδονται ε, απέναντι στους πολίτες και να διαστρεβλώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ξεχυλήσει πια το ποτήρι το Κοινοβούλιο, έχει αναθέσει ειδική εντολή σε υπευθύνους που πρέπει να ε, προστατεύσουν το δικαίωμα των πολιτών σε δημόσιο διάλογο, την διεξαγωγή ανεξάρτητων και ένωμων ε, εκλογών και να υπάρχει ένας διαφανής διάλογος. Θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία που έχουν προβλεφθεί στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Τουντοράκε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ λοιπόν να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες που πρέπει να απευθύνω στον Επίτροπο κύριο Κίνγκ, στην Επίτροπο κυρία Γιούροβα για το όσα μας είπαν προηγουμένως και κυρίως για να χαιρετήσω τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πατάξει αυτή την εξωτερική παρέμβαση στα εσωτερικά μας γιατί μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου ε, καταλάβαμε πως θα πρέπει να αναλάβουμε δράση για να αποφύγουμε αυτούς τους προφανείς κινδύνους και συμφωνώ με όλους τους ε, προλαλίστες και τον κύριο Ντουράν που μίλησαν για αύξηση της χρηματοδότησης για τα όσα έχουμε δημιουργήσει έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να αντιταχθούμε στις ξένες δυνάμεις οι οποίες συστηματικά προσπαθούν να υποσκάψουν την ε, εθνική και ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Συνοχή. Ο Επίτροπος κύριος Κίνγκ την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Λίμπε μας προειδοποίησε. Το Κρεμλίνο έχει διπλασιάσει τις προσπάθειες παραπληροφόρησης που έχει κάνει σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και ο αριθμός των επιθέσεων μέσω κοινωνικών δικτύων έχει αυξηθεί και έχουμε φτάσει τα 20 εκατομμύρια για παράδειγμα στο Facebook. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσω της νομοθετικής μας δράσης για να αντιμετωπίσουμε αυτή την επίθεση. Κυρία Τέρι και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ζούμε σε σταθερές, φιλελεύθερες, ε, ανθεκτικές δημοκρατίες. Πριν από 10 χρόνια θα το είχα υπογράψει και θα είχαν υπογράψει και όλοι εδώ. Και θα το πίστευα και θα έλεγα πως στη δική μου ζωή αυτό δεν θα αλλάξει. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι θα φανώ πιο προσεκτική για τέτοιου είδους δήλωση. Ναι, ακόμα ζούμε σε μια ανεκτική και σταθερή δημοκρατία όλοι μας, αλλά ειλικρινά αυτές οι δημοκρατίες βρίσκονται υπό επίθεση. Η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται ε, και σε περιθωρικές ομάδες και στους ε, ε, μετανάστες στοχεύουν, όπως επίσης και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η χρηματοδότηση μέσω σκοτεινών πηγών προσπαθώντας να καταπολεμήσουν ε, τα δικά μας ανθρώπινα δικαιώματα, να τα περιορίσουν μάλλον ε, και από τη ΣΥΠΑ και από τη Ρωσία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι σημαίνει δημοκρατική διαδικασία, πώς μπορούμε να χειραφετήσουμε την κοινωνία των πολιτών, πώς μπορούμε εμείς να υπερασπίσουμε ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε τις συζητήσεις που είναι απαραίτητες χωρίς να υποσκάπτουμε την βασική ελευθερία που είναι η ελευθερία του λόγου, παρόλα αυτά προστατεύοντας τα λεγόμενά μας. Κύριε Χουχτασάρη, έχει τώρα το λόγο. sananvapautta, jos olemme oikeasti Κύριε Πρόεδρε, εάν πραγματικά θέλουμε να προστατεύσουμε τη δημοκρατία, πρέπει όντως να λάβουμε υπόψη μας ότι η Ρωσία, η Κίνα και η ΕΠΑ θέλουν να επηρεάσουν τα ευρωπαϊκά πράγματα και τις εκλογές και τη διεξαγωγή τους. Πριν από κάποια χρόνια ο πρόεδρος Ομπάμα ήθελε να επηρεάσει τους Βρετανούς με εμπορικές συμφωνίες και ήθελε να τους τρέψει και να τους ε, οδηγήσει να ψηφίσουν σωστά. Δεν είναι καλό όμως οι ψηφοφόροι να ακούνε ότι ξένες δυνάμεις επηρεάζουν ε, τις ευρωπαϊκές εκλογές. Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν μυαλό και μπορούν να χρησιμοποιούν τον εγκέφαλό τους θεωρητικά. Τα, εθνικά, ε, τα εθνικιστικά κόμματα όμως κερδίζουν ε, δυνάμεις διότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να ανακόψουν τη μετανάστευση, θέλουν να ανακόψουν τις ισλαμιστικές δυνάμεις, θέλουν να προστατεύσουν τις χριστιανικές αξίες, τα σύνορά τους και τις ευρωπαϊκές εθνικές αξίες τους και αρχές. Θέλουν οι λαοί της Ευρώπης να είναι η προτεραιότητα και ασχέτως του τι λένε τα κόμματα που έχουν αυτή τη στιγμή την εξουσία. Ο κόσμο έχει απογοητευτεί, δυσφορεί. Θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του και γι' αυτό ψηφίζει τα εθνικιστικά κόμματα. Τώρα οι πιο φιλελεύθεροι πολιτικοί βλέπουμε να χάνουν, ε, να χάνουν δυνάμεις αλλά θα πρέπει να το αποδεχτείτε. Οι εθνικιστικές δυνάμεις κερδίζουμε έδαφος γιατί μας ψηφίζει ο κόσμος. Θέλετε να δημιουργήσετε μια πολιτικό ορθή Ευρώπη και ομάδες εργασίας που να ε, λογοκρίνουν το τι γίνεται στο διαδίκτυο. Δεν θα πείτε στον κόσμο τι να σκέφτεται. Η δημοκρατία δεν περνάει κάποια κρίση και η δημοκρατία δεν θα πεθάνει εάν δεν είναι στην εξουσία φιλελεύθερη. Κυρία Φωτίγκα τώρα. Με όλο το σεβασμό για τα μέτρα που έχουν αναλάβει η Επίτροπος Γιούροβα και ο Επίτροπος King στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου τους, θέλω να υπογραμμίσω ότι μιλάμε για μια εξωτερική διάσταση που αφορά τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως τις παρεμβάσεις ξένων δυνάμεων στις δημοκρατικές μας διαδικασίες. Ναι, βεβαίως και πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των συστημάτων μας και να εμ, θωρακίσουμε τα δημοκρατικά συστήματα. Όμως οι πολιτικές των ξένων παραγόντων και φάνηκε αυτό στην περασμένη φοιτεία ε, με τις εκθέσεις που βάλαμε σχετικά ε, παρεμβαίνουν κυρίως ε, είχαμε μιλήσει για την Ομοσπονδία της Ρωσίας αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες η Κίνα, το Ιράν, η Βόρειος Κορέα οι δικές τους οι ενέργειες με τον πόλεμο της πληροφορίας και της ε, παραπληροφόρησης πολλές φορές είναι ε, σχεδιασμένες ε, αριστοτεχνικά και στοχεύουν με μονομένα κράτη-μέλη κάθε φορά. Γι' αυτό η συνεργασία μας είναι πολύ σημαντική προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί και προκειμένου να αναπτύξουμε το ίδιο αφήγημα και να χαράξουμε κοινέ πολιτικές με υπηρεσίες που ενδεχομένως να βρίσκονται και στην ΕΕΔ. Ευχαριστούμε η κυρία Λέσλι Φίλιπς. Ξέρετε πως όλες αυτές οι εκστρατείες και τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν στους ανθρώπους που θέλουν να επιτεθούν στη δημοκρατία να το κάνουν από όλο το πολιτικό φάσμα, αλλά κάτι ακόμα συμβαίνει. Συνομωσίες που διαδίδονται για πολιτικούς λόγους, για να απονομοποιηθούν τα αποτελέσματα εκλογών γιατί ο ιτημένος δεν δέχεται, δεν δέχεται να παραιτηθεί από την ελπίδα και το είδαμε ε, και στην Αγγλία με το Brexit με ένα νεαρό άνθρωπο ε, που ε, πήγε στο δικαστήριο γιατί προπαγάνδιζε αλλαγή αποτελέσματος και είδαμε ε, και τι συνέβη με τον πικραμένο πρώην πρωθυπουργό του δικού μου κόμματος και τι έκανε στην Αγγλία. Οπορτουνισμός και συνωμοσιολογία από τους ίδιους τους πολιτικούς γιατί όταν κάποια εκστρατεία δεν τους ικανοποιεί ε, προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να την απονομοποιήσουν και αυτό τι κάνει χάνουμε την ε, αξιοπιστία μας στα μάτια των πολιτών είναι σαν την ιστορία ε, του νερού βοσκού που ζητούσε βοήθεια γιατί είχε δει δίθεν λύκο. Έχω δει πολλές ε, μπλε κάρτες να σηκώνονται. Θα δώσω στην κυρία Βόρτ ε, που σήκωσε πρώτη το χέρι το λόγο. Παρακαλώ κυρία Βόρτ. Word, συγγνώμη. Ευχαριστούμε, αλλά για την μυστική εκστρατεία που έγινε με την, και το Facebook, το Cambridge Analytica και την επίδραση στις εκλογές το 2018. Εγώ ήμουν μέλος της Φορευτικής Επιτροπής για εκ μέρους του Κοινοβουλίου και τα αποτελέσματα της έρευνας ε, οδήγησαν στο να παραδεχτεί αυτή η κυρία την ε, συμμετοχή της μέσω του Cambridge Analytica ε, στο στο, με, με, τα αποτελέσματα της έρευνας για το κέντρο αναλυτικά, είδαμε να ε, χάνει τη ζωή του και ένας άνθρωπος ε, υπεύθυνος για την παρακολούθηση των θεμάτων των... Yes. Και το δημοψήφισμα του Ηνωμένου... Με συγχωρείτε, ο χρόνος σας τελείωσε. η συνάδελφός μου πραγματικά προσωποποιεί αυτό που έλεγα προηγουμένως. Ε, εγώ ε, εργάστηκα ως freelancer για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Θα το ξέρετε πολύ καλά και εσείς ξέρετε από αμερικανικές υπηρεσίες της Cambridge Analytica το τι γινόταν και ήρθαν σε επαφή απευθείας μαζί μου για θεωρίες συνωμοσίες στο Twitter με hashtag ανθρώπων που υποτίθεται ότι... Ε, κατήγγυλαν ε, την παραπληροφόρηση. Έχω κουραστεί από όλα αυτά, έχω μπουχτίσει και ε, ενώ υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια μου και δεν μου χτυπούσατε την πόρτα του γραφείου μου να σας τα πω από πρώτο χέρι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόβατ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω και εγώ το εξή. Η δημοκρατία σημαίνει πλουραλισμός, σημαίνει πολυγνωμία. Όταν όμως η δημοκρατία υποσκάπτεται για άλλους σκοπούς. Όταν έχουμε επίθεση ενός εναντίον κυρίαρχου κράτους έθνους, τότε έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Και αυτό μας οδηγεί ε, στο να εκλείπει η ανεκτικότητα και η ανοχή. Και αν ψηφίσουμε εδώ, πείτε μου, τι σημαίνει δημοκρατία. Σημαίνει ε, ελευθερία του ψεύδομαι. Τα ψέματα προστατεύονται ως ελευθερία της έκφρασης. Ας μην είμαστε αφελείς. Είναι τεράστιες οι απειλές από τρίτες χώρες και η Βουλγαρία είναι μόνο μία από τις χώρες οι οποίες το 2015 αντιμετώπισε επίθεση σε επίπεδο κεντρικής εκλογικής επιτροπής. Και όχι μόνο. Αυτό αποτελεί παράδειγμα των όσων συμβαίνουν. Κάποιες κοινωνίες, κάποια κράτη προσπαθούν να υποσκάψουν τις δικές μας χώρες. διάφορες οργανώσεις οι οποίες έχουν ψευδούς λογαριασμούς στα ε, κοινωνικά μέσα και διοργανώνουν ε, μαζικές επιθέσεις εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήθεν υπό την κάλυψη πολιτιστικών θεμάτων κτλ. Θα έπρεπε η δημοκρατία να έχει τα εργαλεία για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Γι' αυτό ζητώ λοιπόν εμείς αυτές τις υβριδικές απειλές όλοι μαζί να τις αντιμετωπίσουμε. Δέχεστε από την κυρία Καπίνη μπλε veniți... παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κόβατσεφ, είστε από τη Βουλγαρία, εγώ είμαι από τη Ρουμανία. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό που είπατε και το θέμα είναι σίγουρα πολύ σημαντικό. Όμως, ως Ευρωβουλευτής, βλέπετε εσείς α, τρόπο να λυθεί αυτό το θέμα. Μιλήσατε για την προστασία της ελευθερίας έκφρασης, την αποτροπή παρεμβάσεων στις εκλογικές διαδικασίες. Τι λύση μπορούμε να βρούμε λοιπόν για το πρόβλημα που θίξατε εσείς. Πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Και για σήμερα μιλάω και για το μέλλον. Απάντηση. Και αυτή η ερώτηση για το τι θα κάνουμε όλοι μαζί. Ε, συντονισμένα θα προχωρήσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη για να πετύχουμε κάποιο περιορισμό σε αυτές τις επιθέσεις και εκστρατείες ε, παραπληροφόρησης και εκτός και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καλύτερο βήμα προόδου είναι να υποβάλουμε τέτοια αιτήματα στις πλατφόρμες έτσι ώστε να ακολουθούν ένα κώδικα διοντολογίας και να στηρίξουν τους σωστούς δημοσιογράφους να κάνουν ε, εκπαίδευση και επιμόρφωση στους δημοσιογραφικούς κύκλους και κυρίως να έχουμε τους πόρους. Γιατί η δημοκρατία χρειάζεται ένα ε, δίκτυ προστασίας. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κλοντ Μωράης. Thank you, President. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ζητήσαμε ισχυρότερα μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην παρεμβαίνουν σε εκλογές μας ε, από το εξωτερικό, να μην μας χειραγωγούν και να μην έχουμε παραπληροφόρηση ε, online ή offline. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Θα ήθελα όμως να πω σε όλους εδώ, και εδώ απευθύνομαι και στα νέα μέλη, πώ το κάνουμε εδώ και μήνε. Η Επίτροπος και ο Επίτροπος δήλωσαν πως έχουν αναλάβει δράση. Η Προεδρία το έχει κάνει και στη δική μας ομάδα θέλουμε να ζητήσουμε να συσταθεί μια ειδική επιτροπή για να εμβαθύνει στις δράσεις αυτές. Και το ζητάμε γιατί τα κράτη-μέλη δεν θα μπορέσουν να αντέξουν για πολύ ακόμα. Είναι πολλά τα προβλήματα και θα σας τα εξηγήσω. Οι πολίτες μας ψηφίζουν σε εκλογές όπου έχουμε ε, κόμματα της άκρας δεξιάς, όπως στη χώρα μου, που χρηματοδοτούνται και δανειοδοτούνται από ξένες χώρες. Επίσης βαθιά παρέμβαση ε, offline και θα πρέπει για παράδειγμα να μην επιτρέπεται η συλλογή προφίλ ε, ανθρώπων για εκλογικούς ε, λόγους και υπάρχει και περιεχόμενο το οποίο θα χρειαστεί να αποσυρθεί από το διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής Σιμέτσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Υπουργέ. Η παρέμβαση ξένων δυνάμεων σε δημοκρατικές εκλογές είναι μια πραγματική εκλογή. Είδαμε πολλές περιπτώσεις όπου οι προσπάθειες παραπληροφόρησης σκοπό είχαν να διαιρέσουν τους πολίτες, να τους χειραγωγήσουν και να επηρεάσουν την ψήφο τους. Βεβαίω αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Γι' αυτό η Φιλανδική Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύουν να επιληφθούν του θέματο στο προσεχέ μέλλον. αυτό πραγματικά απειλείται για τα θεμέλια τη δημοκρατία. Διότι χωρί μια διεξοδική συζήτηση για τα γενεσιουργά αίτια των προβλήματων αυτών δεν μπορούμε να προστατεύουμε τη δημοκρατία. Ταυτόχρονα έχει υποθεί ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώ οι με θεωρίε συνωμοσία ή το ρωσικό χρήμα, αλλά η πολιτική οι δικοί μα πολιτικοί που συνεργάζονται χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα, τα εργαλεία. Στην δική μου την περιοχή, στην κεντρική Ευρώπη, πολλοί πολιτικοί, κάποιοι υπουργοί διασπείρουν συνωμοσίε θεωρία στο ευρωκοινό. Ε, ή εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να δημιουργήσουν ε, συσχετισμού ε, πλειοψηφία. Αυτό είναι επικίνδυνο για την δημοκρατία. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφο Ένσλι Σκότ. Η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, οι βασικές αρχές πλήττονται εδώ και πολλά χρόνια. Ο Ψηφιακή εποφή και τα χρήματα έχουν χρηματοδοτήσει την άκρα δεξιά με προπαγάνδες οι οποίες δεν έχουν χώρο σε προοδευτικές χώρες εκλογική παρέμβαση, παραπληροφόρηση, τοξικές για τη συζήτηση σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να διαιρέσουν τις κοινότητές μας και να πάψουν οι πολίτες να εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα. Και η χώρα μου έχει πέσει σε μια περιδίνηση συνταγματικής αμφισβήτησης και ο πρόεδρος της σχετικής επιτροπής στη Βουλή των Κοινοτήτων είπε και παραπέμπω είναι η δημοκρατία μας που κινδυνεύει και οι εκλογικοί μας θεσμοί είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι απαρχιωμένοι και αυτό από τη μητέρα των κοινοβουλίων. Δεν μπορεί να είμαστε εδώ και να κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε. Είναι οι ουσιαστικές αξίες οι δικές μας και των κοινοβουλίων μας, στις πρωτεύουσμές μας από κακόφημα άτομα που προσπαθούν να υποσκάψουν δημοκρατία για τους δικούς τους στόχους. Χρειαζόμαστε στεναρία, αντίσταση και προστασία. Θα πρέπει να μπορούν οι πολίτες να αποφασίσουν μόνοι τους για την τύχη τους και όχι να είναι έρμεα αυτών που έχουν βαθιές τσέπες. Σας ευχαριστώ. Δύο πράγματα. Θα σας παρακαλέσω. Το πρώτο να προσέχουμε όλοι το χρόνο αγόρευσης. Όταν έχετε ξεπεράσει το χρόνο αγόρευσης, ε, σας αφήνω πρώτα πέντε, μετά δέκα, δευτερόλεπτα και μετά διακόπτω την ομιλία. Ένα αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της μπλε κάρτας, να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. για να μπορέσουμε να τηρήσουμε την, ε, το χρονοδιάγραμμα των συζητήσεων. Αφού το είπα αυτό, τώρα να σας ζητήσω να μου πείτε αν δέχεστε από την κυρία Ντελούτσι μία μπλε κάρτα. Ευχαριστώ, πολύ για την ευκαιρία. Το δέχεστε πρώτα απ' όλα. Δέχεστε τη γαλάζια κάρτα. Θα είναι πολύ γρήγορη η ερώτησή μου. Δεν τη δέχεται. Πάμε στον επόμενο ομιλητής ομιλητή, ο κύριος Γκαρό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ο κώδικας καλών πρακτικών κατά της παραπληροφόρησης ε, δίνει μεγάλη σημασία στην ε, ελευθερία τη έκφραση και στο ελεύθερο διαδίκτυο. Αυτά λέει το κείμενο. Αυτό όμω ο κώδικα καλή συμπεριφορά έχει εγκριθεί και γίνει αποδεκτό από το Facebook, το Twitter και το Google. Αυτοί είναι οι φορεί που είναι υπεύθυνοι για το ε, περιεχόμενο που προσφέρεται στου χρήστε του διαδικτύου. Κι όμω, πολλέ φορέ λογοκρίνουν αυτά που θεωρούνται παραπληροφόρηση. Και αυτό γίνεται διαρκώ με μέτριε λύσει. Δηλαδή, αντί να υπάρχουν ε, λογοκρισίες ή αντί να υπάρχουν λογότυπα fake news, δεν μπορούμε να θυμώνουμε τους χρήστες που απλώς έχουν ε, εκφράσει τις απόψεις τους κατά τον λόμπι και των ε, διαθέσεων ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κατακλείσει τα πάντα. Στη Γαλλία, λοιπόν, ε, έχει, για παράδειγμα, διαγραφή άρθρο το οποίο επέκρινε την ε, δημόσια γαλλική τηλεόραση και τις απόψεις που εξέφραζε για τους ε, μετανάστες. Ε, και υπήρχε ένα άρθρο που αντιδρούσε στην συμπεριφορά αυτή ο δρόμο προ την κόλαση, λέμε στα γαλλικά, είναι στρωμένο με τι καλύτερε προθέσει. Όμω εδώ έχουμε τα χέρια στα αποτελέσματα και αυτά που είχε περιγράψει και ο Τζορτζ Όρουελ στο μυθιστόρημά του 1984. Το 2019 υπάρχει σαφώ ο πειρασμό ε, να έχουμε φορεί που χειρίζονται την παγκοσμιοποίηση με μεγάλα, ε, ποσά στα, στη διάθεσή του για να ε, ανακόψουν αυτού που ονομάζουν με περιφρόνηση λαϊκιστέ. Η λογοκρισία όμως μέσω μαζικής ενημέρωσης ήταν κάτι που ε, άσκησαν από την ε, αρχή του χρόνου όλα τα πολιταρχικά καθεστώτα. Πρέπει λοιπόν εδώ να ε, δούμε την προσπάθεια των πιστών τη παγκοσμιοποίηση να μπλοκάρουν όλου του υπόλοιπου. Θέλετε, λέτε, να δημιουργήσετε έναν ε, χώρο υγειονομικά ε, παρακολουθούμενο για να προστατεύσετε τη δική σα ιδεολογία. Εμεί θα αντιδράσουμε σε όλο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει μπλε κάρτα που να τη ζητεί κάποιο βουλευτή από την ίδια πολιτική ομάδα. Άρα δεν ε, μπορώ να δεχθώ αυτή την ε, μπλε κάρτα. περνάμε στον επόμενο μιλητή που ξαντέ Βιλιάλμπα. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, το Vox, το δικό μου κόμμα, είναι ριζικά αντίθετο με οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα της δικής μας χώρας. Φυσικά και πιστεύουμε στην εθνική κυριαρχία, στην κυριαρχία των κρατών μελών. Και χαίρομαι που για πρώτη φορά ίσως και άλλες πολιτικές ε, ομάδες ε, ε, υπερασπίζονται το αναπαλωτρίο της εθνικής κυριαρχίας. Μέχρι αποδείξεως του εναντίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι λόγος για ευρωπαϊκή κυριαρχία αλλά αποκλειστικά για εθνική κυριαρχία. Και μπορεί σε πολλούς από εσά ή σε μένα να μην μας αρέσει η ανάμειξη της Ρωσίας στα εκλογικά στήματα. Δεν μας αρέσει όμως ούτε το ότι ο Μακρόν και 52 Γάλλοι βουλευτές ε, ε, επηρεάζουν ε, την κοινή γνώμη εκφράζοντας κριτική για ένα ή άλλο κόμμα της χώρας μου. Και τη διαδικασία δεν μας αρέσουν οι ξένες παρεμβάσεις. Ούτε θέλουμε όμως αυτό να είναι πρόσχημα για τη δημιουργία της Επιτροπής της Αλήθειας όπως στο βιβλίο του Άρλου του 1984 για να μας μας λένε υπερεθνικές οργανώσεις τι πρέπει ή δεν πρέπει να λένε οι υπήκοοι του καθενός κράτους μέλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το, για το κανονισμό επί της διαδικασίας θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε συζητούμε ε, τις ψευδείς ειδήσει. Είπατε πριν ε, ότι είναι στην ID ε, ουσιαστικά τα μέλη του, του κόμματος του Brexit και δεν μπορούν να ζητήσουν μπλε κάρτα. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι στην ομάδα μας οι βουλευτές αυτοί και λυπούμε εμείς που υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία να μην δίνουμε τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της μπλε κάρτας. Ο πρόεδρος αποφασίζει, κύριε συνάδελφε, την ε, διαδικασία αυτή της μπλε σε ποιον θα δώσει το λόγο. Υπάρχουν σαφεί κανόνες, τους οποίους ε, και τήρησα, γι' αυτό αρνήθηκα την μπλε κάρτα στην προκειμένη περίπτωση. επόμενο ο κύριος Λέναρς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα κύριε Πρόεδρε οι ελεύθερε εκλογέ είναι το θεμέλιο τη δημοκρατία μα. Πρέπει να τι προστατεύσουμε ε, και όποιο τολμήσει να απειλήσει το θεμέλιο αυτό θα πρέπει να μα βρει κάθετα αντίθετου. Με όλη μα τη δύναμη πρέπει να αντισταθούμε. Ε, δεν θέλουμε όμω ε, να έχουμε πρόβλημα με, τη, με τα κοινωνικά μέσα, με τι νέε τεχνολογίε που θα δυσκολεύουν και περισσότερο την διάκριση μεταξύ αλήθεια και ψεύδου. Αν δεν το κάνουμε το 2021 ο κόσμος ε, θα παίρνει πολύ πιο πολλές ψευδείς από ό,τι ειδήσει. Ε, είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό. Είναι μια πρόκληση. Το Google και άλλες ε, τέτοιε εταιρείε και πλατφόρμες παίζουν, για να μην πω κάτι, θα έπρεπε να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο γιατί α, μου δίνεται εντύπωση ότι λειτουργεί ε, κάπως καλά, αλλά όχι όσο θα έπρεπε καλά. Η συνεργασία μας με τους κολοσσούς αυτούς. Εντάξει, ε, μια μικρή ίσως τιμωρία, ε, έτσι για τα μάτια του κόσμου. Ε, όμως εδώ μιλάμε για την παραπληροφόρηση. Μπορεί για ένα μαθητή μια ε, τιμωρία έτσι ε, ελαφριά να αρκεί. Δεν αρκεί για την παραπληροφόρηση. Πρέπει να δούμε τι κυρώσεις μπορούμε να επιβάλλουμε, πώς θα πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα οι εταιρείε αυτές. Η αυτορύθμιση που προβάλλεται σήμερα ως λύση δεν μας ικανοποιεί. Κύριε Κίνγκ, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες γίνεται λόγος για νομοσχέδια, εγκρίνονται νομοσχέδια. Πώς όλα αυτά τα νομοσχέδια θα τα συντονίσετε για να μην βρεθούμε τελικά με 28 διαφορετικές νομοθέσεις, 28 διαφορετικές χώρες.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 αρμοδιότητα του Προέδρου είναι να αποφασίζει κατά πόσον θα δεχθεί μια μπλε κάρτα και το δεύτερο, το πρόσωπο στο οποίο απευθύνει την μπλε κάρτα επίσης ε, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα τη δεχθεί ή όχι. Έτσι λοιπόν έγινε και αυτή η απόφαση ελήφθη. Και τέλος, ο κύριος Σίλβα Περέιρα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η παραπληροφόρηση της κοινή γνώμης μέσω ψευδών ειδήσεων στα κοινωνικά δίκτυα που κάθε φορά είναι όλο και πιο ε, εξελιγμένα και ε, παραχαρα... καλά παραχαραγμένα είναι μια σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία μας με πολιτικές δυνάμεις και ξένους ε, που, φορείς που δρούν από το εξωτερικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά λαμβάνει μέτρα για να ελέγξει το χώρο αυτό και αυτό είναι μια καλή πρωτοβουλία διότι θα πρέπει οι εταιρείε των κοινωνικών δικτύων να αναλάβουν τις ευθύνε τους και βεβαίως όλοι να φροντίσουν να προσφέρουν πληροφορίες ελεγμένες κατά καταπολεμώντα τις ψευδείς. Θα πρέπει να βρεθούμε στο ύψο των περιστάσεων και των απαιτήσεων των καιρών μα. Το Κοινοβούλιο με μια ειδική επιτροπή που θα μα επιτρέψει να ενισχύσουμε την άμυνα των δημοκρατικών μας καθεστώτων είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό η συγκεκριμένη έκθεση είναι πολύ σημαντική και θα ψηφίσουμε υπέρ. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλερ. Κυρίες και κύριοι, Κύριε Επίτροπη, τις τελευταίες φορές τα είπατε, οι πρόσφατες εκλογές αντιμετώπισαν επιθέσεις από σταθεροποίησεις και από κράτη και από μεμονωμένους παίκτες. Το είπαν αρκετοί συνάδελφοι και ήταν άνευ προηγουμένου. Κύριε Τζούλιαν Κίνγκ, μας υπενθυμίσατε πως είχαμε τουλάχιστον ε, δεκάδες χιλιάδες ε, ψευδών λογαριασμών που στήριξαν αυτή την ε, Παραπληροφόρηση. Κυρία Γιούροβα, κύριε Κίνγκ, έχετε αναλάβει μια πρωτοβουλία το Σεπτέμβριο του 2018 μαζί με τα κράτη-μέλη για να δώσετε τα όπλα στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσει αυτή την εγκληματικότητα. Δεν ήταν όμως αρκετό. Ποιες είναι οι επόμενες πρωτοβουλίες για να ενισχύσετε τη σύγκληση των στρατηγικών σε εθνικό επίπεδο. Πώς θα ενισχύσετε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την ασφάλεια έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια σπίδα προστασίας γύρω από την Ευρώπη. Η ομάδα μας είναι υπέρ μιας τέτοιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας για να προστατεύουν τη δημοκρατία από κάθε επίθεση και θα τη στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Διδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, πόρο απέχει απ' ε, να σας ε, αμφισβητήσω τα προνόμια του προεδρεύοντος ε, Όμω αρνηθήκατε την μπλε κάρτα, λέγοντα ότι ο λόγο βουλευτέ ανήκει στη δική μα ομάδα, δηλαδή είναι στην ίδια ομάδα τα δύο άτομα. Είναι ψευδή είδηση, δεν ανήκει στην ομάδα μα και σήμερα μιλάμε για τι ψευδεί ειδήσει. Ακριβώ αυτό συζητάμε τώρα. Αυτό έλεγα. Ήδη τοποθετήθηκα σε σχέση με το θέμα αυτό. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχα. Αν υπάρχει κάποια παρανόηση θα το δούμε, αλλά τώρα πηγαίνω ε, στην επόμενη μιλήτρια σύμφωνα με τη μίσια διάταξη, κυρία Γκρεγκόροβα. Ευχαριστώ, αξιότιμη πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, οι βρεδικές απειλές, ε, ο πόλεμος των πληροφοριών. Είναι οι σύγχρονες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις που γίνονται σε νέα θέατρα επιχειρήσεων. Δημοκρατία, ελεύθερες εκλογές είναι κάτι που ξένες δυνάμεις το εναντίον μας. Μόνο και μεγαλύτερη ένταση και αποτελεσματικότητα. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό σύστημα αποτροπή στο πλαίσιο της αμυντικής μας στρατηγικής. Ωστόσο, Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφύγουμε μέτρα που κινδυνεύουν να καταστρέψουν τα θεμέλια των δημοκρατικών κοινωνιών μας. Η ελευθερία λόγου δεν ορίζεται από εμπορικά μονοπόλια. Είναι κάτι άκρο πολύτιμο για να το ορίζουν οι πλατφόρμες ε, και κάποια φίλτρα. Θα πρέπει λοιπόν να να καταπολεμήσουμε την προπαγάνδα και την ξένη παρέμβαση με τη βοήθεια των τεχνολογιών. Αλλά οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να βοηθούν και ε, σε μαζική κλίμακα παρέμβασης. Ε, πρέπει κατά αυτού να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, να υπερασπίσουμε τις δημοκρατικές μας αξίες χωρίς να τις υπονομεύσουμε. Μας κάνουμε λοιπόν έτσι το βήμα στον 21ο αιώνα. Ευχαριστούμε κυρία Κριστίνα Άντερσον. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σήμερα μιλάμε για το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της ε, εξάπλωσης της παραπληροφόρησης. Πραγματικά φαίνεται αστείο όταν ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι κατάλληλη να καταπολεμήσει τις ψευδείς ειδήσει. Είναι το κεντρικό επιτελείο της παραγωγής όλων των ψευδών ειδήσεων. Ε, και μάλιστα η πρόσφατη μπροσούρα, το φυλάδιο 60 λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπουν οι ευρωπαϊκοί λαοί σε 64 μπλεγμένα τα τα πλεονεκτήματα που τους φέρνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Ε, ε, στη σελίδα 16 έχουμε την ε, δήλωση ότι το 2016 τα κράτη-μέλη εξοικονόμησαν 50 δις ευρώ. Αυτό είναι ψευδής είδηση. Είναι μια τρελή κυβέρνηση αυτή που θέλει να συμπαρασύρει τους ευρωπαϊκούς λαούς και να θριαμβολογήσουν για τις εξοικονομήσεις που στην πραγματικότητα είναι κλοπή της περιουσίας τους. Ε, εδώ πραγματικά όταν ε, η ίδια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ατζέντα για την Ευρώπη γράφει για τη δική μου γενιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει υπόσχεση ειρήνης, ευημερίας και ενότητας ώστε να μπορέσουμε με ένα κοινό νόμισμα να προστατεύσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και την, ε, την πραγματική ευημερία. Αυτό είναι η μητέρα όλων των εκστρατιών των ψευδών ειδήσεων. Έχουμε υποσχεθεί ε, ειρήνη και ευημερία και πραγματικά έχουμε ε, ένα τρελοκομείο γραφειοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να συμπαρασύρει τους ευρωπαϊκούς λαούς με υπερβολικές ρυθμίσεις και κανόνες, ξεγελώντας τους ε, τα είδαμε να συμβαίνουν στη Γαλλία, τις κάτω χώρες και την Ελλάδα. Οι ευρωπαϊκοί λαοί ρωτούν πότε θα μπορέσουμε κι εμεί όπω οι Βρετανοί με ένα δημοψήφισμα να δείξουμε τι άποψη έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν άλλα προγράμματα δράση, ε, γιατί όλα γίνονται ήδη εδώ. Κυρία Άντερσον, μπορείτε να δεχτείτε μια γαλάζια κάρτα τον κύριο Μάντελ. Όχι. Ο κύριος Μπίτικοφερ. Κύριε Πρόεδρε, ε, για την διάταξη των εργασιών μας η κυρία Άντερσον μόλις, εκτός μικρόφωνο, η κυρία Άντερσον χαρακτήρισε το σώμα μας ένα ε, τρελοκομείο γραφειοκρατίας. Είναι προσβολή αυτή προς το Ευρωκοινοβούλιο και παρακαλώ να το διαγράψετε από τα πρακτικά και να αντιδράσετε αναλόγως. Για αυτό το χαρακτηρισμό που τόσο σωστά ε, παρατηρήσατε κι εσείς ε, θα υπάρξουν τα κατάλληλα μέτρα. Ο κύριος Βάιμερς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιε παρεμβάσει για το τι, ε, κάποια παρέμβαση για το τι συμβαίνει όταν έχουμε τέτοιε απαράδεκτε προσπάθειε παραβίαση εκλογική ε, διαδικασίας, παρέμβαση στα εσωτερικά των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ε, και παρεμβάσεις όταν ε, συναντιόνται οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Είναι απαράδεκτα, αλλά είναι απαράδεκτο επίσης να χρησιμοποιούμε τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου για να προσπαθούμε να χειραγωγήσουμε τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Να ένα έγγραφο για τα 350 εκατομμύρια κορώνα, κορώνα σουηδικής που χρησιμοποιούμε χρησιμοποιήθηκε για να χρηματοδοτηθούν εκστρατείες lobbying ε, πριν τις εκλογές. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν με ρωτήσετε εμένα, προσπαθεί να πιέσει τον κόσμο να ψηφίσει κατά τη διάρκεια των εκλογών. Και επίσης δεν επιτρέπει στον κόσμο να κάνει την επιλογή ε, υπέρ του κυρίαρχου, εθνικά, ε, κυρίαρχου κράτους και κατά της Ομοσπονδιοποίησης Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Σικόρσκι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω το λόγο στην ε, αίθουσα της Ολομέλειας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που λαμβάνω το λόγο για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Διότι έχω υπάρξει θύμα μιας κυβερνομάδας. Πήρα και τα ίδια ε, mail που πήρε ο κύριος Ποντέστα στη ΣΥΠΑ και ξέρω πως αυτό επηρέασε εκεί την εκστρατεία. Ε, υπήρχαν κάποια παραδείγματα τα ακούσαμε από προλαλήσαντες ε, παραδείγματα ξένης παρέμβασης στην Ιταλία, τη Γαλλία, τη Βρετανία αλλά και στη δική μου τη χώρα πρόσφατα όπου ο κύριος Ζετχόφσκι δημοσίευσε ένα βιβλίο, ένα σημαντικό βιβλίο και εδώ θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στην εισαγγελία να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη ε, τις πληροφορίες για παρέμβαση στην ε, πολωνική πολιτική. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, θα έλεγα καλύτερα, να κάνουμε. Η πολιτικοποίηση των μίντια η συσχέτισή τους με πολιτικά κόμματα ουσιαστικά διευκολύνει αυτούς που θέλουν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα εκλογών. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαθέσουμε μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην υπηρεσία της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, να ενισχύσουμε ε, τις δυνατότητες ε, των εθνικών ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το Creative Europe πρέπει να το περικοδοτήσουμε με περισσότερα κονδύλια, να λύσουμε δε τα ζητήματα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρακαλώ. Να μην έχουμε χειροκροτήματα από τα θεωρία. Δεν επιτρέπεται αυτό από τον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Και τώρα περνάω στον επόμενο, τον κύριο Λόπεθα Γιλάρ Ευχαριστώ πολύ την Προεδρία, τον Επίτροπο. Έχουν περάσει 10 χρόνια που η συνθήκη της Λισαβόνας ε, τέθησε εφαρμογή. Και αν μας είχαν πει τότε πως θα συζητούσαμε το θέμα αυτό ως προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συζητούσαμε για την απειλή των bot, των troll, των μη κρατικών ή κρατικών παρεμβάσεων όπως για παράδειγμα το θέμα της Ρωσίας ε, που επιτίθεται κατά των δημοκρατικών θεσμών και της τοξικής συζήτησης που γίνεται, δεν θα το είχαμε πιστέψει. Όμως είναι απειλή αληθινή και δεν είναι ούτε ουδέτερη, ούτε θα πρέπει να την υποεκτιμήσουμε. Γιατί έχουμε ακραίες και λακιστικές παρεμβάσεις που ακούγονται συνέχεια και κυρίως επιτίθεται εναντίον ευάλωτων και ε, μειονοτήτων και θα πρέπει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μαζί μια απόκριση με τους κανονισμούς και τους πόρους που χρειάζονται. Θέλουμε επενδύσεις έτσι ώστε να καταστρέψουμε αυτούς τους ψευδολογαριασμούς και για να έχουμε ε, μια ενίσχυση της ευρωπαϊκής ε, προσπάθειας ε, του να καταπολεμήσει τις προσπάθειες αυτές μέσω μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας την οποία θα στηρίξουμε όλοι μας. Ο κύριος Κέτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ελευθερία έκφρασης αποτελεί ακρογωνία ολίθιο της δημοκρατίας και ε, την σεβόμαστε. Αυτή τη στιγμή είναι η παραπληροφόρηση η οποία έχει εξαπλωθεί λόγω της διαστροφής αυτής στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μόνο την κορυφή του παγόβωνου και είναι πραγματικά επίγον το να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξεκίνησε τη μάχη, αλλά πώς θα ελέγξουμε και θα επαληθεύσουμε τις πληροφορίες χωρίς να πέσουμε στην παγίδα της λογοκρασίας. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ξέρετε πως η δημοκρατία έχει μάθει να δίνει τη μάχη κατά του ψεύδους χωρίς να καταστρατηγεί την ελευθερία έκφρασης και αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα. Θα πρέπει να βρούμε την νομοθετική απόκριση μέσω μιας ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Αυτό θα πρέπει να το κάνουν και οι δικαστές αλλά και οι δημοσιογράφοι. Εγώ είμαι. Δεν έχουμε εφεύρει τίποτα. Θα πρέπει και εμείς να δεσμευτούμε πως θα είμαστε σαφείς, αληθινοί ε, και δεν θα αφήσουμε το παραμικρό παρεθόριο σε όσους προσπαθούν να μας αποστασιοποιήσουν σταθεροποιήσουν, είτε αυτοί προέρχονται από το εξωτερικό, είτε όχι. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ταρντίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ψευδή ειδήσει και παραπληροφόρηση είναι ένα πραγματικός, ένας πραγματικός κίνδυνος που μπορεί να επηρεάζουν τους πολίτες στη διεξαγωγή των εκλογών και ε, επηρεάζει βεβαίω και τι προεκλογικέ εκστρατείε. Όπω ε, υπόθηκε εδώ, υπάρχουν βέβαια έρευνε για συγκεκριμένε περιπτώσει και υποθέσει πρόσφατα με ψευδεί ειδήσει και παραπληροφόρηση και θα κρυθούν από τα δικαστήρια. Πρέπει λοιπόν εδώ τι δημοκρατικέ μα αξίε να τι προστατεύσουμε και στο διαδίκτυο, αλλά ταυτόχρονα και την ελεύθερη κυκλοφορία των ιδεών και την ελεύθερη έκφραση για σκοπού ανεξαρτησία και ανθρώπινε αξιοπρέπεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόσχημα την καταπολέμηση τη παραπληροφόρηση δεν μπορεί να ενθαρρύνει τη λογοκρισία και την καταπίεση των ε, απόψεων που δεν συμφωνούν με τους περισσότερους. Εδώ λοιπόν πώς μια ιδιωτική εταιρεία όπως το Facebook έχει το δικαίωμα να λογοκρίνει ένα πολίτη χωρίς να παρέμβει κάποιος ανεξάρτητος φορέας ή δημόσιος έστω για να τον προστατεύσει. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε πολύ προσεκτικά τέτοιου είδους κανόνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντούρις Νικολόσνοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχει καμία σημασία σε ποια πολιτική ομάδα ανήκει ο καθένας. Έχουμε όλοι μία δουλειά, μία κοινή ευθύνη να εντοπίσουμε αυτούς που διαρκώς οργανώνουν ε, απόπειρες παραπληροφόρησης για να πλήξουν και να αποσταθεροποιήσουν τα δημοκρατικά μας ε, καθεστώτα. Ε, ήδη από τον Μάρτιο είδαμε τέτοιες υποθέσεις και πολλές φορές και σε τρίτες χώρες, Βολιβία ή Ινδία. Πρέπει λοιπόν να δούμε προσεκτικά ε, τέτοιες προσπάθειες που έγιναν να επηρεαστούν και αυτές οι χώρες από την κυβέρνηση του Πούτιν και τη Ρωσία. Έχουν μάλιστα δημοσιευτεί απειλές στο διαδίκτυο ότι πολλές από τις εκλογές μάλλον ε, ισχυρισμοί ότι πολλές από τις εκλογές του 2016 είχαν απευθείας επηρεαστεί από δυνάμεις του ε, Πούτιν ελεγχόμενες από τον Πούτιν. Μιλάμε για ένα είδος κοινωνικού μάτριξ. Εδώ είναι πολλές οι δυνάμεις που παρεσφύγουν στα εθνικά κοινοβούλια και ελέγχονται ως πιόνια από τις δυνάμεις του Πούτιν, που είναι ο πραγματικός επιτιθέμενος. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπίλτσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, η υβριδικός πόλεμος, ε, η διάδοση παραπληροφόρησης ε, ψευδών ειδήσεων απειλούν ιδίως ε, τους δημοκρατικούς θεσμούς στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, όπως χρειαζόμαστε επίσης ελεύθερα και δίκαια δημοψηφίσματα. Και επειδή η πολιτική εκστρατεία στο μεγαλύτερο μέρος τη γίνεται σε περιβάλλον μέσων κοινωνικής δικτύωση, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το διαδίκτυο μπορεί να αντιμετωπίσει εγκαίρω και αποτελεσματικά τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Στην Αυστρία είδαμε πρόσφατα hacker να επιτίθενται. Αυτό δείχνει πόσο ευάλωτε είναι οι ευρωπαϊκέ δημοκρατίε ε, στην ξένη παρέμβαση ε, σε εσωτερικέ ε, ευρωπαϊκέ διαδικασίε. Και βλέπουμε στην Αυστρία να απλώνεται η παραπληροφόρηση. Οι μικρότερε τώρα δημοκρατίε έχουν λιγότερου πόρου στη διάθεσή του και λιγότερα μέσα για να έχουν ε, επαφή με τις ε, μεγάλες πλατφόρμες, τους κολοσσούς ε, του διαδικτύου για την καλύτερη προστασία από την παραπληροφόρηση. Πώς θα προστατεύσουμε λοιπόν τη δημοκρατία στην Ευρώπη με μια ισχυρή κοινή πολιτική προσέγγιση στον τομέα της επικοινωνίας και της εργασίας με τα μέσα κοινωνικής δικαίωσης των αγώνα κατά της παραπληροφόρησης. Γι' αυτό και απευθύνω έκκληση και στην Κομισιόν αλλά και στην Φιλανδική Προεδρία του Συμβούλου να αντιμετωπίσει σοβαρά το ζήτημα. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ επίσης διότι τηρήσατε το χρόνο αγόρευσης. Επόμενος ομιλητής τώρα είναι ο κύριος Ραφέλ Γκλουξμάν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ναι, απειλείται ο δημοκρατικός τρόπος ε, διαβίωσης. Δεν απειλείται όμως από τους ε, εξόριστους που τους αφήνουν να πεθάνουν στη Μεσόγειο. Απειλείται από δυνάμεις οι οποίες αναμειγνύονται σε εκλογές και στις δημόσιες ε, συζητήσεις. Υπόθεση Στράχη στην Αυστρία. Υπόθεση χρηματοδότησης της Λέγκα στην Ιταλία. Υπόθεση Cambridge Analytica. Οι ρωσικές τράπεζες του γαλλικού μετόπου, εθνικού μετόπου. Όλα αυτά δείχνουν ε, τις σχέσεις ε, της Τη τη δεξιά με το καθεστώ του Βλαδιμίρ Πούτιν και τι χρηματοπιστωτικέ σχέσει επίση που έχουν. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν και πόσο ευάλωτα είναι τα δημοκρατικά συστήματα στην ξένη παρέμβαση. Α αφήσουμε λοιπόν του φανταστικού εχθρού, ε, όπω είναι οι μετανάστες και α δούμε ποια είναι η πραγματική απειλή. Αυτό που ζητώ αγαπητοί συνάδελφοι σήμερα είναι πραγματικά να δεχτείτε να συγκροτηθεί ειδική επιτροπή που θα ρίξει φω ε, στι ε, ξένε παρεμβάσει και θα ορίσει τον τρόπο να τι αντιμετωπίσουμε. Γιατί ουσιαστικά όταν μιλάμε για την επιβίωση τη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να αφήνουμε να μα ποδοπατούν. Πρέπει να αντιδράσουμε. Καιρό είναι. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ο κύριο Νίλ Τόρβαλτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο. Πριν έρθω έκανα μία πολύ σύντομη ανταλλαγή πληροφοριών με την Κέση Τζέσικα Ερό που ήταν η δημοσιογράφος ε, η οποία η, οποία αποκάλυψε τι γίνεται με, τα, με τις ρωσικές ε, ε, μυστικές υπηρεσίες και την παραπληροφόρηση και με την προσπάθεια απαγωγής που έγινε στην Αγία Πετροπολή. Πρέπει να σου πω πως κανείς δεν θα ήθελε να βιώσει κάτι α, αντίστοιχο γιατί προσπάθησαν να την καταστρέψουν ως προσωπικότητα. Δεν τα κατάφεραν, ήταν πολύ δυνατή. Αλλά έχω να σας ρωτήσω το εξή. Μπορείτε να δώσετε αρκετά χρήματα στην Ιντερπολ έτσι ώστε αυτές τις εγκληματικές πράξεις να μπορέσουμε να τις καταπολεμήσουμε. Herr ο κύριος Κρασνοντέψκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν και εγώ κύριε Πρόεδρε και πιστεύω πως όλοι θα συμφωνήσουμε αυτή η παρέμβαση τρίτων μερών στις ε, εσωτερικές εκλογικές μας διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της παραπληροφόρησης αποτελεί σοβαρή απειλή εναντίον της δημοκρατικής διαδικασίας και των δικαιωμάτων των πολιτών μας που ζητούν αξιόπιστες πληροφορίες και ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας και σεβασμό αυτής των κρατών μελών. Όλοι δε γνωρίζουμε πως δεν είναι τυχαίο που αναφερόμαστε μόνο σε ένα κράτος, συνέχεια τη Ρωσία και μάλιστα δεν είναι μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και οι φίλες χώρες της ανατολικής της σχέσεις ε, ανατολικής γειτονίας ε, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα και θα πρέπει να τις βοηθήσουμε να δώσουν τη μάχη κατά της παραπληροφόρησης. Και βέβαια έχουμε ψευδείς ειδήσει, τα fake news που προέρχονται και από άλλους παίκτες όχι μόνο από κρατικές πηγές. Συμβαίνει αυτό παντού. Και επίσης σήμερα μπορούμε να δούμε πως αυτοί οι οποίοι ε, κινούν ε, συνωμοσιολογικές ε, θεωρίες ακούγονται πολύ ε, και αντιμετωπίζουν τις εκλογές ως ένα παιχνίδι το οποίο προσπαθούν να επηρεάσουν. Ευχαριστούμε ο κύριος Ρανζέλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή ε, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια. Πρέπει να πω πολύ ξεκάθαρα το εξής. Η δουλειά που έχουμε μπροστά μας κατά της ε, παραπληροφόρησης, της εξαπάτησης και της φραγώγησης, ιδίως σε περίπτωση εκλογών, δεν είναι δουλειά που μπορεί να γίνεται μόνο τις παραμονές των εκλογών. Πρέπει να γίνεται ε, διαρκώς, γιατί η χειραγώγηση της κοινή γνώμης είναι κάτι που γίνεται πολλές φορές σταδιακά, βαθμιδών και στα κοινωνικά δίκτυα, στις διάφορες πλατφόρμες του ίντερνετ και με συμβατικά μέσα. Η απάντησή μας λοιπόν πρέπει να είναι διαρκείας και κατά τα άλλα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορεί να κάνει εδώ πολλά, ε, μπορεί να κοιτάξει τις πλατφόρμες Τη της τεχνολογίας και να υπάρχει ε, συνεργασία όχι μόνο έκτακτη αλλά σταθερή με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους εθνικούς φορείς και να κοιτάξουμε την προστασία των πολιτών ε, εκπαιδεύοντάς τους. Αυτό μου φαίνεται το πλέον σημαντικό. Η εκπαίδευση των πολιτών. Είτε με... Και με συγχωρείτε πρόεδρε, αλλά νομίζω ότι έχω 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Η εκπαίδευση λοιπόν των πολιτών, η εκπαίδευση των ίδιων των πολιτικών, διότι και οι πολιτικοί πολλές φορές αθελά του συμβάλλουν στις ψευδείς ειδήσει. Πρέπει να, είναι, ε, να έχουν ε, συνείδηση και συνέστηση οι πολιτικοί ηθήνοντες και οι υπεύθυνοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι όλων των υπερχόντων μέσων πρέπει να εκπαιδεύονται. Ε, είναι σημαντική λοιπόν η εκπαίδευση όλων για να αναχαιτήσουμε τις ψευδείς ειδήσει την χειραγώγηση και να αποφύγουμε τον πραγματικό κίνδυνο, τον πραγματικό κίνδυνο της λογοκρισίας που φαίνεται να αναδύεται και δεν την θέλουμε. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Καλέντα Καρλό. Ευχαριστώ. Η φιλελεύθερη δημοκρατία δέχεται επιθέσεις και θα δέχεται επιθέσεις και την ερχόμενη δεκαετία. Εκ των έσω από δυνάμεις όπως η Λέγκα του Βορρά και το κίνημα των Πενταστέρων στην Ιταλία. Η επίθεση αυτή βεβαίως οξύνεται σε ε, καιρούς εκλογών, γιατί βεβαίως η δημοκρατία μόνο από τη δημοκρατία, με τη δημοκρατία μπορεί να ε, προστατευτεί. Και δέχεται επίθεση και εξ και εδώ δεν μπορεί η δημοκρατία μόνη της να αυτοπροστατευτεί. Πρέπει να υπάρξει μια ειδική επιτροπή για να διαλευκάνει κατά ποιον συγκεκριμένο τρόπο υπήρξαν ε, παρεμβολές από συγκεκριμένα κόμματα που υποτίθεται ότι προασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα, αλλά τελικά προασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα ξένων και τρίτων χωρών. Αυτό ε, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και η Ευρώπη πρέπει να προσπιστούν τους εαυτούς τους. Η δημοκρατία, είναι ελεύθερη, δημοκρατία είναι ισχυρή, αλλά μόνο εάν την προστατεύσουμε σωστά. Διότι είναι σαφές ότι ό,τι πρόσχημα και να βρει κανείς ε, με, ψευδά, με ψευδή προσχήματα ουσιαστικά ε, εκτοξεύει μια κατηγορία στον εαυτό του. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκροσέφ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω το εξής η παρέμβαση αυτών των κρατικών ή μη κρατικών παικτών στις προεκλογικές μας διαδικασίες, αλλά και σε άλλες διαδικασίες που είναι πραγματικά στη βάση των ε, δημοκρατικών μας πολιτευμάτων στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή έχει εκτοξευθεί και υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Πρέπει λοιπόν με στοχευμένες και τους συντονισμένες δράσεις να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή με στεναρό τρόπο, με τη νέα τεχνολογία και με την πρόσβαση που έχει αυτή στη σπίτια μας, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προστατευτούμε για να έχουμε μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία με την ελευθερία της έκφρασης, η οποία όμως θα μπορεί να προστατευτεί. Υπάρχουν τεχνικές προπαγάνδες και υπάρχουν σοφιστικέ μέθοδοι έτσι ώστε να ε, διαστρέψουν την αλήθεια και να δημιουργήσουν μια ψευδή εντύπωση της πραγματικότητας και αυτό απειλεί και και που την ε, συζήτηση που γίνεται ε, στις κοινωνίες μας. Έχουμε τις βασικές μας αξίες και θα πρέπει να τις σκεφτούμε και να τις προστατεύσουμε με έναν τρόπο που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου. Και θα πρέπει η απόκριση που θα δώσουμε να είναι σωστή, ανάλογη, παληθεύσιμη και κυρίως να μην πέσει θέμα χειραγώγης από ξένους παίκτες. Ρόμπερτ Σίλε, επόμενος ομιλητής. δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την παραπληροφόρηση και πρέπει να ε, θυμόμαστε, είτε μας αρέσει είτε όχι, ε, ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλές απειλές οι οποίες ε, υπονομεύουν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς πρέπει να εστιάσουμε να συγκεντρώσουμε τα μέσα και τους πόρους, δηλαδή στη συνεργασία. Ουσιαστικά πρέπει να εστιάσουμε κάτι που ήδη το κάνουμε. Ίσως χρειάζεται μια νέα οργάνωση, δεν ξέρω. Υπάρχει το κέντρο αριστείας επίσης που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Η συνεργασία όμως πρέπει να εμβαθύνει περισσότερο για να προστατεύσουμε καλύτερα τις εκλογές στις χώρες που ε, τώρα θα τις διοργανώσουν ε, σε λίγους μήνες. Ευχαριστώ. Η Μπενθουμέα, Ιζαμπέλ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Πρέπει να σας πω πως αυτά τα ψευδί, ψευδές ειδήσει είναι βλαβερές για τις φιλελεύθερες κοινωνίες και είναι μια α, μεγάλη απειλή αλλά και στόχος. Αυτά τα fake news δημιουργούν σύγχυση στους πολίτες. Χάνουν την ε, εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς και κορυδεύουν τον κόσμο το πιο σοβαρό είναι ότι δημιουργούν και πολιτική αστάθεια. Και δεν θα πρέπει να κοροϊδευόμαστε. Είναι ένα εργαλείο των εχθρών των ανοιχτών κοινωνιών, των αυταρχικών ε, καθεστώτων και των λαϊκιστικών δυνάμεων που προσπαθούν να καθοδηγήσουν την συζήτηση σε ε, κοινωνικό επίπεδο για να πετύχουν κάποιους στόχους. Έχουμε και με τον Brexit τέτοιο παράδειγμα και με τα όσα αντιμετωπίσαμε ε, με την πρόκληση της ανεξαρτησίας το 2017 στην Ισπανία. Τότε η ανεξάρτητη Καταλάνοι χρησιμοποίησαν τις ικανότητες που έχουν ε, στην διασπορά ψευδών υγήσεων και ε, χειραγώγησης προσπαθώντας να διαδώσουν μια αρνητική εικόνα της Ισπανίας που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Αυτό δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ούτε με λογοκρισία ούτε με περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης. Θα πρέπει να έχουμε μέσα επικοινωνιών και μίντια που θα εξασφαλίζουν πως οι ειδήσει που δίνουν στους πολίτες είναι αξιόπιστες. Θα πρέπει οι πολίτες μας να είναι υπεύθυνοι και να έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν. Και θα πρέπει βέβαια να δούμε και πώς θα εκπαιδεύσουμε τους νέους μας να έχουν τις δεξιότητες αυτές έτσι ώστε να μπορούν ορθά να κρίνουν. Θα το κάνουμε για να ανταποκριθούμε στις ψευδές ειδήσει. Μόνο έτσι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίξερ. Είναι σημαντικό να γίνεται αυτή η συζήτηση, αν και δεν αρκεί, ε, διότι το μέγεθο πρόκληση είναι τεράστιο. Στηρίζω λοιπόν τη δημιουργία ειδική επιτροπή που θα έχει ω καθήκον να μελετήσει το ρόλο τη ξένη παρέμβαση σε εκλογικέ δικασίε. Η Ρωσία προσπαθεί να παρεμβεί στις εθνικέ εκλογικέ δικασίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, τεκμηρωμένε είναι και άλλε κακάβλες επιθέσει από τη χώρα αυτή. Αναφέρθηκαν κάποιε από αυτέ τι περιπτώσει και το Κρεμλίνο και άλλα ανελεύθερα καθεστώτα δεν κρύβουν το γεγονό ότι ε, Χθάνονται τι ευρωπαϊκέ αξίε, όπω η δημοκρατία, άρα δεν θα έπρεπε να μα εκπλήξει το ότι στηρίζουν οικονομικά ή με άλλου τρόπου, πολιτικέ δυνάμει σε άλλε χώρε ε, που και αυτέ ε, δεν συμμερίζονται τι δημοκρατικέ μα αξίε. Πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι θέλουν να υπονομεύσουν και την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών ε, στα δημοκρατικά εκλεμμένα θεσμικά όργανα και να απο, να αφαιρέσουν ε, την αξία αυτών των δημοκρατικών ε, θεσμών καθεστώτως αναξιόπιστου. Άρα νομίζω ότι η συγκρότηση αυτή τη επιτροπή είναι βγουν προ σωστή κατεύθυνση. Okay. Σα ευχαριστώ πολύ, Στάνισλαβ Πόλτσακ. Ευχαριστώ. Ακόμη και αν υπήρξαν προσπάθειες ε, δυνάμωσης της συζήτηση, εγώ θα μιλήσω για τη ρωσική προπαγάνδα και το ρόλο της, διότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Κρεμλίνου στη διάθεση ψευδών πληροφοριών. Έχουμε μακράν εμπειρία, ευρή εμπειρία ε, στην Τσεχία από τη ρωσική προπαγάνδα ε, με την εισβολή του 68 που ήταν ε, κάτι που το παρουσίαζαν ως ε, μια χείρα βοηθείας, μια φιλική χειρονομία και έχουμε και κάποιες ε, άλλες τέτοιες ε, περιπτώσεις τις οποίες θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Η υποχρεωτική αναφορά ε, συμβάντων από τις πλατφόρμες, το σύστημα εγκρισης προειδοποίησης είναι μερικά από τα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν την καλύτερη ανταλλαγή ε, πληροφοριών σε σχέση με αυτές τις εκστρατείες παραπληροφόρησης. Είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει στο συντονισμό. Βέβαια, σήμερα πολλά εξαρτώνται από το κατά πόσον αυτά τα μέτρα θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη. Έχω μεγάλες προσδοκίες από την κυρία Γιούροβα, η οποία θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο αυτό. Παραπληροφόρηση και ψευδής ειδήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Κύριε Πόλτσακ, δέχεστε μια μπλε κάρτα. Όχι, λέει ο κύριο Πόλτσακ. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, επόμενος ομιλητή. ο κύριος τον Πίτσουλα. Ευχαριστώ πολύ. Με την ψηφιοποίηση στις διάφορες πλατφόρμες αυξάνονται οι παραπληροφόρηση. Αυτό φυσικά είναι παράνομο. Δεν υπάρχει επαρκής προστασία των ιδιωτικών πληροφοριών, ούτε παλήθευση ε, της ε, των πληροφοριών. Έχουμε το σκάνδαλο Cambridge Analytica, που δείχνει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παραπληροφόρηση για να διαμορφώσει αποτέλεσμα εκλογών, η προεκλογική εκστρατεία. Τα δύο τρίτα των πολιτών έδειξαν στοιχεία του νεμβρίου, ανησυχούν για τη χειραγώγηση και την επηρεασμό εκλογών. Είδαμε και μετά τις ευρωεκλογέ ότι υπήρξαν ε, παρεμβάσεις τρίτων ε, χωρών για... και τελικά όλα αυτά που δυναμώνουν ε, την εγκυρότητα των... και την αγκαιρότητα των εκλογικών διαδικασιών. Πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν ε, στη καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. Πρόεδρος, έχουμε ένα μακρύ κατάλογο για τη διαδικασία Catch the Eye. Catch the Eye. Αλλά δεδομένου του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας δεν θα μπορέσω να δώσω σε όλους το λόγο. Από όσου λοιπόν έδωσαν το λόγο, ε, ζήτησαν το λόγο, θα ξεκινήσω σε αυτό, με αυτούς που δεν έχουν ακόμη μιλήσει. Κυρία Μόνικα Γκοντζάλης. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που θα προστατεύει τα άτομα. Και τι σημαίνει αυτό. Ενίσχυση και θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο ε, μήνυμα εμείς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύουμε γιατί έχουμε αυτά τα μηνύματα τα οποία βασίζονται σε εθνικιστικά και λακιστικά μηνύματα εναντίον κοινοτήτων όπως οι μετανάστες ή διαφορετικού ε, θρησκευτικού προσανατολισμού, ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Με μία προώθηση του μίσους και αυτό είναι κάτι το οποίο είδαμε στην Ισπανία και στις τελευταίες εκλογές είδαμε πως πρόκειται για μια πολιτική απολογία που βασίζεται στην έχθρα εναντίον ε, ΛΟΑΤΚΙ ε, μεταναστών, βασίζονται σε χριστιανικές ε, παρενέσεις, ψάχνοντας από δύο πομπέους τρίγου, τράγους, με συγχωρείτε, γιατί ο άλλος πια είναι ο εχθρός. Αυτός ο λαϊκισμός χρηματοδοτείται από ξένες ομάδες και γι' αυτό χρειαζόμαστε εμείς να ψηφίσουμε και με ένα ψήφισμα να δείξουμε στεναρά πώς θα υπερασπίσουμε αυτές τις ομάδες, αυτές τις κοινότητες με μια ειδική επιτροπή η οποία θα ε, αναζητήσει λεπτομέρειες για το τι συνέβη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κονσάλη. Ο κύριος Οστρεβίτσιος είναι επόμενος. Ευχαριστώ πολύ. Σκεφτείτε μια στιγμή μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ορίζει παγκόσμια ε, πρότυπα ε, για τη δημοκρατία να μην έχει ελεύθερα μέσα, να μην έχει ερευνητική δημοσιογραφία, η ε, κοινωνία μας να εκτίθεται σε ξένες απειλές, να έχουμε χρηματοδότηση από ξένους πολλών δημοσιογράφων. κάτι που βλέπουμε να γίνεται από Ρωσία, Κίνα και άλλους ακραίους. Είμαι πεπισμένος ότι κανείς δεν θεωρεί ότι είναι ε, ότι κανείς δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει να αναθεωρήσουμε τα περί όλων αυτών των ε, εκστρατιών παραπληροφόρηση. Χρειάζονται μηχανισμοί ελέγχου και για τη διαλογή των στρατηγικών επενδύσεων. Έτσι θα στηρίξουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Ευχαριστούμε κύριε Αουστρεβίτσιους. Και τώρα ο κύριος Ζερόμ Ριβιέρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα την Επιτροπή με ιδιαίτερη προσοχή και άκουσα επίση ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τον εαυτό τη για την καταπολέμηση τη παραπληροφόρηση και τη ψευτής ειδήσει και ακούω ε, ότι υπάρχουν χώρες που ε, έχουν να αντιμετωπίσουν δικές τους ε, περιπτώσεις παρεμβολών όπως η Βρετανία που φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες παρεμβολής στην λήψη εθνικών αποφάσεων χαίρεται που φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ιταλία οι δίκες που ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί και όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, φαίνεται να παρεμβαίνει η ίδια στις εθνικές υποθέσεις των μεμονωμένων κρατών και παρεμβαίνει σε θέματα εκτός της αρμοδιότητάς της. Ουσιαστικά ε, προσβάλλει τις συνθήκες μας ε, και τις παραβιάζει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν φαίνεται να είναι πολύ ψηλά τα ιδεώδη σας, αλλά δεν φαίνεται να βλέπετε τι γίνεται μπροστά στην πόρτα σας. Ευχαριστούμε κύριε Ριβιέρ. Επόμενος. Η ναι, Θα ήθελα... Είναι ηρωνικό που μιλάμε για παρεμβάσεις σε εκλογική διαδικασία όταν εδώ γνωρίζουμε πως έχουμε δημοκρατικό έλλειμμα. Αναρωτιέσαι γιατί ασχολούνται. Η πραγματικότητα είναι πως η εξωτερική παρέμβαση γίνεται από τότε που ξεκίνησαν οι εκλογές. Η ΕΠΑ παρεμβαίνει σε τεράστια κλίμακα, όχι μόνο στην Μέση Ανατολή ε, στην Λατινιακή Αμερική αλλά στην καρδιά της Ευρώπης. Και ο μοναδικός λόγος για τον οποίο μιλάμε τώρα και αναφερόμαστε στο φάντασμα της ρωσικής παρέμβησης είναι για να κατηγορήσουμε κάποιον για τις καταστροφικές επιδόσεις των καθεστωτικών ε, κομμάτων στην Ευρώπη. Οι πολιτικές άφησαν εκατομμύρια πολίτες πίσω, τους έσπασαν το ηθικό, και αυτή είναι η πραγματική λόγοι Γιατί ε, είχαμε Brexit, γιατί βγήκε ο Τραμπ, γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία της άκρας δεξιάς. Είναι εύκολο να μιλά κανείς για συνορμοσία από εξωτερικό εχθρό, αλλά οι πολίτες ξέρουν τι χρειάζεται. και αν ανησυχούμε για τις εκλογικές παρεμβάσεις, ας αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες παρεμβάσεις στις δημοκρατικές διαδικασίες από τους λομπίστες, από τους δισεκατομμυρούχους στους οποίους ανήκουν εφημερίδε από τις πολυεθνικές. Φτιάξτε αυτά και δεν θα ανησυχείτε πια για το Facebook και για το Twitter και για ψευδείς λογαριασμού που έτσι κι αλλιώς κανέναν δεν ανησυχούν. Ευχαριστούμε κυρία Ντέιλι. Ο λόγος στο κύριο, στο κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω του Επιτρόπου και τη Φιλανδική Προεδρία και να εκφράσω τι ελπίδε μου ότι θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε και να εγκρίνουμε ένα ε, ψήφισμα αποφασιστικό για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Οι παρεμβάσει στι εκλογικέ διαδικασίε και οι κυβερνοεπιθέσει, ένα τόσο ιερό δικαίωμα όπου εγγράφεται και στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις είναι απαράδεκτες. Πρέπει λοιπόν τη σημασία του συντονισμού για την προστασία των τεχνικών υποδομών που εξασφαλίζουν τη σωστή διεξαγωγή των ε, δημοκρατικών ε, διαδικασιών, προσπάθειες δηλαδή να γίνει hacking, υποκλοπή ή ε, παρεμβολή στα θεμέλια της δημοκρατίας μας είναι κάτι που δεν πρέπει να επιτρέψουμε. Πρέπει να είμαστε εμείς ο πρώτος ο πρωταγωνιστής στον αγώνα κατά των προσπαθειών αυτών και να λυθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα όσο προσπαθούν να παραβιάσουν τους κανόνες της ελεύθερης δημοκρατίας. Ευχαριστούμε. Ε, πρόφερα χάλια το όνομά σας. Είστε κυρία Κάλιουραντ. Και τώρα Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Catch the Eye, προσέλκυση τη προσοχή του Προέδρου. Δεν μπορώ να παραχωρήσω περισσότερο χρόνο, έχουμε ήδη καθυστερήσει στο πρόγραμμά μα, γι' αυτό να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον κύριο Κιν. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ για αυτή την τόσο επίκαιρη συζήτηση. Και όπως είπατε αρκετοί από εσά, οι εκστρατείε παραπληροφόρησης έχουν σκοπό να παρακολύσουν ε, τους πολίτες μας να μπορούν να κάνουν επιλογές ενημερωμένες, να διαιρέσουν τις κοινότητες και τις χώρες μας, να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα των εκλογικών μας διαδικασιών, την ακαιρεότητα των δημοκρατικών μας θεσμών. Δεν νομίζω πως μπορούμε να αποδεχθούμε ε, κάτι αντίστοιχο στη νέα συνηθισμένη πραγματικότητα. Πρέπει να αντιδράσουμε. Ένα κομμάτι του προβλήματος προέρχεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετοί από εσά αναφερθήκατε στη Ρωσία. Θέλω να είμαι σαφής. Υπάρχει μια ομάδα στους θεσμούς, στην οποία αναφερθήκαμε, και που έχει το καθήκον να παρακολουθεί τις εκστρατείες παραπληροφόρηση από το Κρεμλίνο. Οι εκθέσεις τους είναι δημόσια προσβάσιμες, αλλά στην πρόσφατη περίοδο που τσεκάρισαν, οι συντονισμένες ε, παραπληροφορίες υπέρ του Κρεμλίνου σε κάποια κράτη-μέλη το τελευταίο διάστημα είχαν διπλασιαστεί. Αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα και δεν πρέπει να το αποφεύγουμε. Αλλά είναι σαφές επίσης πως κάποιοι διδάχτηκαν από τους Ρώσους θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, περισσότερα μέτρα που να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να αντιδράσουμε για τέτοιου υποθέσεις από όπου και να προέρχονται. Και γι' αυτό ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και με την, πολιτεία των κοινων, ε, την κοινωνία των πολιτών ε, θεσπίσαμε μια σειρά μέτρα. Δεν ε, είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι και δεν είμαι εδώ για να διαφεντέψω τι δάφνε μα. Χρειάζονται παραπάνω. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας στις εκλογικές διαδικασίες. Στους επόμενους μήνες, στις επόμενες εβδομάδες θα αναθεωρήσουμε τον κώδικα διοντολογίας για την παραπληροφόρηση για να κάνουμε να τα πάμε καλύτερα στην προσπάθεια προστασίας της κοινωνίας μας που είναι δημοκρατική και μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου θα σα υποβάλουμε τη σχετική έκθεση. Να σας πω, ε, σε αντίδραση σε κάποια από τα σχόλια, αυτός ο κώδικας διοντολογίας κατά της παραπληροφόρησης που έχουμε μαζί με τις κοινωνικές πλατφόρμες δεν έχει καμία σχέση με τη λογοκρισία. Καμία σχέση με την ιδέα αυτή του Υπουργείου Αλήθειας με κεφαλαίο. Δεν έχει καμία σχέση με το αν είναι καλή ή όχι η πολιτική άποψη που εκφράζεται, αλλά με το να φωτίσει την πολιτική συζήτηση να είναι πιο διάφανη έτσι ώστε στη συζήτηση να γνωρίζουν. Βλέπουν πληροφορίες. Από πού προέρχονται. Ποιος έχει πληρώσει. Άνθρωπος ή μηχανή η οποία κυκλοφορεί τις πληροφορίες. Αυτό είναι ζωτική σημασία εάν θέλουμε να έχουμε τα εργαλεία που θα μας επιτρέπουν να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές. Επίσης, έχουμε και την έκθεση για τα εκλογικά μέτρα που πήραμε εν των ευρωεκλογών και θα σας δώσουμε την έκθεση αξιολόγησης. Ετοιμάζουμε και το σχέδιο δράσης της Ευρώπης για να είμαστε πιο ανθεκτικοί και όλα αυτά θα τα καταθέσουμε μέσω νομοθετικών ε, πρωτοβουλειών για να είμαστε πιο διάφανοι με πιο σαφείς κανόνες για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων. Και παράλληλα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αυτούς τους επαληθευτές, τους ερευνητές, την κοινωνία των πολιτών και τα κράτη-μέλη, όπως επίσης και τις online πλατφόρμες, για να κάνουμε πρόοδο και να έχουμε ένα ε, καλό και ασφαλές ε, μέλλον στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε, Επίτροπε Κίνγκ. Υπουργέ του Ποράινεν από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα είναι πραγματικά επίκαιρο και κέριο είναι προτεραιότητα για την Προεδρία μα και ευχαριστώ για την ε, τόσο εντατική σα συμμετοχή. Η ανθεκτικότητα τη Ένωσή μα εδράζεται στην ενότητα. Όσο πιο ενωμένοι, τόσο καλύτερα μπορούμε να αντισταθούμε στην διάδοση και την εξάπλωση αυτού του φαινομένου της παραπληροφόρησης. Δεν θα βυστούμε προσπαθειών να προστατεύσουμε την έννομη διεξαγωγή εκλογών και τα εκλογικά και δημοκρατικά συστήματα από την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Σεβόμενοι όλα τα βασικά δικαιώματα όμω, την ελευθεροτυπία, την ελεύθερη έκφραση, την ελευθερία του συνασπίζεστε. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε διατομιακά, πέρα από σύνορα, πέρα από στερεότυπα. Μαθαίνοντα εμένα από του ΔΕ, ανταλλάσσοντα βέλτιστε πρακτικέ και εμπειρίε. Πρόοδο έχει επιτελεστεί ήδη. Όμω, όπω είπαν η Επιτροπό Γιούροβα και η Επιτροπό Κίνγκ, πρέπει να παραμείνουμε σε επιφυλακή και σε επαγρύπνηση. Όπω είπα, οι υβριδικέ απειλέ ήδη στην ανακοίνωσή μα έχουν τύχει ιδιαίτερη έμφαση. Ετοιμάζουμε και νέε πρωτοβουλίε ε, σε συνεργασία με την Επιτροπή που τι έχει προαναγγείλει. Και να θυμίσω η γενική ευαισθητοποίηση των πολιτών μα ω προ τι νέε ευρετικέ απειλέ είναι θεμελιώδου σημασία. Οι ανοιχτέ και ελεύθερε κοινωνίε και η σωστή διαχείριση των δεδομένων να επιτρέπουν τη σωστή παραπληροφόρηση. Οπότε έτσι θα φροντίσουμε να εκκριζώσουμε αυτό το ζυζάνιο τη παραπληροφόρηση. Σα ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την τόσο επικοδομητική και πλούσια συζήτηση. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ Τουπουράινεν. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος αυτού και στην επόμενη σύνοδο θα τεθούν σε ψηφοφορία τα ψηφίσματα σε σχέση με τη συζήτηση αυτή. Θα κάνουμε τώρα μία σύντομη διακοπή και θα συνεχίσουμε με την επόμενη συζήτηση σε λίγα λεπτά. Επανερχόμαστε στη συνεδρίαση, κυρίες και We start our debate again. The next point in our agenda, the, the statement of the Commission and the Council concerning to the forest fires. του Συμβουλίου, το λόγο έχει η κυρία Τουπουράινεν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, πιστεύω ότι δεν είμαι μόνιμο όταν λέγω ότι το θέμα που έχουμε σήμερα για να συζητήσουμε, οι δασικές πυρκαγιές που καταστρέφουν την περιοχή του Αμαζονίου, είναι κάτι άκρος ανησυχητικό για όλους μας. Οι πυρκαγιές είναι τραγωδία όχι μόνο για τους ε, πληγέντες πληθυσμούς, αλλά για τον πλανήτη μας ευρύτερα και για το κλίμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε το δάσος του Αμαζονίου για να είμαστε αποτελεσματικοί στη δράση κατά της αλλαγής του κλίματος. Το δάσος του Αμαζονίου είναι μοναδικά πλούσιο και ποικιλόμορφο. Ε, ένα από τα δέκα είδη στον κόσμο έμβια ζωή ε, έμβιων όντων στην, στον πλανήτη ζουν εκεί. Λοιπόν, είναι σοβαρή απειλή για την αλλαγή του κλίματος χάνονται πολλά ήδη από τις πυρκαγιές και χάνονται και μεγάλες εκτάσεις από το δάσος. Αυτές οι πυρκαγιές σχετίζονται άμεσα με αποδάσωση εκπροθέσεως. Δυστυχώς παρατηρούμε με τα ότι ήταν πρόσφατα χειρότερα τα περιστατικά στη Βραζιλία και στη Βολιβία και στην Παραγουάη οι πυρκαγιές. Αυτές οι πυρκαγιές ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα ε, σκοτώνουν πάρα πολλά είδη φυτών της περιοχής και ζώων και διώχνουν και τους αγενείς πληθυσμούς από τις περιοχές που ζουν. Ε, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην δράση για το κλίμα και την προστασία των δασών πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα της ε, Φινλανδικής Προεδρίας. Είναι προτεραιότητα. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν καταστροφικές συνέπειες και για τα ζώα και για τους ανθρώπους Εξαρτώμεθα από τα δάση για τη διατήρηση της για να περιορίσουμε τα αποτελέσματα της αλλαγής του κλίματος και να δώσουμε και δουλειά στου ανθρώπους. Συμβάλλει το δάσο επίσης στην επίτευξη των προσδοκιών που έχουμε για ουδετερότητα όσον αφορά το κλίμα μέχρι το 2050. Συζητήθηκε η προετοιμασία για τη Σύνοδο Κορυφή για το σχέδιο δράση του ΟΗ σήμερα το πρωί, το συζητήσαμε και η απογευματινή συζήτηση ε, σχετίζεται άμεσα με αυτό το θέμα. Παρά τις δράσεις που δρομολογήθηκαν μέχρι τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποχρεώσεις που ανελήφθησαν ε, διεθνώς, η αποδάσωση και η επιδείνωση καταστάσεων των δασών συνεχώς αυξάνονται σαν προβλήματα και οι καταστροφικές πυρκαγιές στον Αμαζόνιο ε, μας οδηγούν στην ανάγκη να αυξήσουμε τις προσπάθειες και κατεπηγόντως μάλιστα. Τον Απρίλιο του 2019 το Συμβούλιο θέτησε συμπεράσματα όσον αφορά την επιτυχία πρόοδο, όσον αφορά την εφαρμογή τη στρατηγική για τα δάση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Σε αυτή την περίσταση, ε, το Συμβούλιο τόνισε τη σημασία που έχει η στρατηγική για να εξασφαλίσει συνοχή και συντονισμό των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και των 100 μελών όσον αφορά τα δάση και να προωθήσουμε περισσότερο τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Το Συμβούλιο Αλία και Γεωργία θα συζητήσει το θέμα τον επόμενο μήνα. Θα συζητήσει την ανάγκη νέα στρατηγική μετά το 2020 που θα εδράζεται από των ιδίων αρχών αλλά λαμβάνοντα υπόψη και τι νέε αλλαγέ πολιτικών στα κράτη-μέλη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα έχουν λάβει μια ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναμένει το επιμακρόν για αύξηση τη δράση Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του κόσμου. Θα εξετάσουμε λεπτομερώς τις προτεραιότητες που προτείνονται στις εκθέσεις και προσβλέπουμε στις δικές σας ιδέες επ' αυτού του ζητήματος. Το Συμβούλιο θέλει να παράσχει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά την ανακοίνωση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην μορφή συμπερασμάτων του Συμβουλίου που ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθούν το Δεκέμβριο του 2019. Τα προβλήματα ξεπερνούν τα δάση. Θέλουμε να συμμετάσχουν διάφοροι εμπειρογνώμονε από συναφεί τομεί, περιβάλλον, γεωργία και εμπόριο και άλλοι τομεί να συμμετάσχουν προσπάθεια. Προσβλέπουμε στα δράση στην ανακοίνωση αυτή και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν οι συνεισφορέ σα σε μελλοντικέ δράσεις για τα δάση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Κλείνοντα να υπογραμμίσω ότι οι δασικές πυρκαγιέ στον Αμαζόνιο είναι μια κατεπίγουσα παγκόσμια κρίση. Απαιτεί αποτελεσματική διεθνή απάντηση και ανταπόκριση. Στενή συνεργασία με τι χώρε τη περιοχή του Αμαζονίου είναι κρισίμου σημασία. Αυτέ οι χώρε, όπω είναι η Βραζιλία, έχουν κάθε δικαίωμα να ηγηθούν τι προσπάθειε, αλλά πρέπει να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει που έχουν αναλάβει. Απευθύνω θερμή έκκληση στι χώρε τη περιοχή του Αμαζονίου και στου ηγέτε των χωρών για κατεπίγουσα δράση Είμαστε εμεί έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον κύριο Μπολσονάρο και με του άλλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη, αλλά χρειάζεται τώρα δράση. Η Φιλανδία, προεδρεύουσα του Συμβουλίου, θέλει να ε, ηγηθεί του προβληματισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την αντίδραση. Κατόπιν Βουλία, οι Υπουργοί Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω συζήτησαν στην άτυπη συνεδρίασή του στο Ελσίνκι το θέμα ε, τέλο Αυγούστου. Οι Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν επί της σοβαρότητας καταστάσεως και τόνισαν την ανάγκη συντονισμού και ολοκληρωτικής προσέγγισης για τη μετώπιση της κρίσης. Ως προεδρεύοντες του Συμβουλίου θα εξακολουθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως να συμβάλλουμε στο να εξασφαλίσουμε μια ενιαία, συνεπή και αποτελεσματική δράση της Ευρωπαϊκής Ενώσης όσον αφορά το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Το λόγο εξ ονόματι της Επιτροπής έχει ο Επίτροπος κ. Βέλλα. Thank you, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Προεδρίας. Ε, συνάδελφοι, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, σήμερα αντιμετωπίζουμε μια σημαντική κρίση για το κλίμα και την βιοπικιλότητα που επηρεάζει την ζωή μας, τις οικονομίε μα και το μέλλον μα. Οι πυρκαγιές σε δάση σε όλο τον κόσμο απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, εμβαθύνοντας την κρίση όχι μόνο στον Αμαζόνιο, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως είναι η Σιβηρία. Ο Αμαζόνιος όμως ε, έχει ένα μοναδικό ε, δάσος και για το οξυγόνο που αναπνέουμε και για τη βιοπικιλότητά του και μοναδικό για την υγεία του πλανήτη. Γι' αυτό χαίρομαι που έχετε θέσει ψηλά στο θεματολόγιο σας το θέμα αυτό. Ε, είναι απαραίτητο να αναχαιτήσουμε την, την ε, αποδάσωση για τρει βασικού λόγου. Πρώτον, να σταματήσουμε την απώλεια τη βιοπικιλότητας, να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματο και για να πετύχουμε ε, τους στόχους του θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τι δεσμεύσει μα ε, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού. Η υποβάθμιση και η απώλεια των δασών έχει σημαντικέ επιπτώσει στη σταθερότητα, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κλίμα, τη βιοπικιλότητα την υγεία και το βιός ε, και των ε, τοπικών κοινοτήτων και του συνόλου του πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθάει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στις χώρες του Αμαζονίου όπου υπάρχουν επικαγές και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες αρχές συμπεριλαμβανομένων των αρχών της Βραζιλίας. Ήδη ε, έχουν τεθεί σε λειτουργία κάποια μέτρα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση κατόπιν αιτήματος της Βολιβίας. Ε, το Κέντρο ε, Άμεσης ε, Αντίδρασης έχει στείλει εμπειρογνώμονες στην πυρόσβεση προς τη χώρα αυτή και τέτοια βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί σε κάθε χώρα κατόπιν αιτήματος. Επίσης, το σύστημα χαρτογράφησης Κοπέρνικος έχει κινητοποιηθεί και ε, ε, ε, παρέχονται χάρτες και στην Βραζιλία και στο Περού και την Παραγουάη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη χρηματοδοτεί προγράμματα ανάπτυξης που σχετίζονται με τα δάση και τη χρήση γης στην Λεκάνη του Αμαζονίου, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, 128 εκατομμύρια ευρώ συνολικά αντιπροσωπεύει ε, το πρόγραμμα αυτό και έχουμε σχεδιάσει δράσεις ε, ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ. Βρισκόμαστε ε, σε επαφή με τις αρχές της Κολομβίας που συντονίζουν τις περιφερειακές προσπάθειες για αντιμετώπιση της κατάστασης. Στην πρόσφατη συνάντηση κορυφής G7 ε, προετοιμάσαμε μια συνάντηση ε, για την περιφέρεια του Αμαζονίου ε, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ενώ η άμεση προτεραιότητά μας είναι να καταπολεμήσουμε τις πυρκαγιές, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις διαθροτικές αιτίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση για την αποκατάσταση των δασών. Η ανακοίνωση αυτή περιγράφει μία σειρά μέτρων συμπεριλαμβανομένης της στήριξη για βιώσιμε πρακτικές χρήσης της γης. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τις χώρες εταίρους μας θα ε, ε, ε, ε, ασκούμε λιγότερη πίεση στα δάση και θα ενθαρρύνουμε την αποκατάσταση των δασών. Θα πρέπει επίσης να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα και να εφαρμόσουμε νομοθετικά και μη μέτρα για να περιορίσουμε την εισαγωγή προϊόντων που σχετίζονται με την αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασών. Επίσης, θέλουμε να βελτιώσουμε την πληροφόρηση για τα δάση ε, και τις ε, αλυσίδες προϊόντων. Ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασών. Οι επιστημονικέ πληροφορίε αποτελούν σημαντικό στοιχείο τη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεργασία με χώρε εταίρε ε, θα είναι το κλειδί μεταξύ άλλων για να ε, εντοπίσουμε ε, τις οικονομικές μακροπρόθεσμες συνέπειες της περαιτέρω αποδάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες τη κατά της καταστροφής των δασών και θα βοηθήσουμε όσους επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Αμαζόνιο και σε όλο τον κόσμο με κάθε δυνατό τρόπο και σε συνεργασία με τις αρχές των χωρών αυτών ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το λόγο έχει για δύο λεπτά κυρία Μαγκίνες, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Τουπουράινεν. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά από δάση και χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση στη δική σας Προεδρία και ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο για τις λεπτομέρειες. Υποθέτω ότι πολλοί επισκέπτες θα είδαν τις πυρκαγιές ε, στην Αμαζονία και χαίρομαι που οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς μπορούμε να συνεργαστούμε παγκοσμίω, γιατί δεν μπορεί καμία χώρα μόνη της να λύσει αυτά τα προβλήματα. Τη στιγμή όμως που θέλουν να είναι κυρίαρχα τα κράτη, χωράει η πολυμερή συνεργασία και η ενίσχυσή της αντί την αποδυνάμωσή της. Δεν βοηθάει να είναι οι χώρε δακτυλοδεικτούμενε. Ξέρουμε που είναι τα λάθη, αλλά αναγνωρίσαμε και την πρόοδο. Για τη Βραζιλία, α πούμε, πρόσφατα έχει αναλυφθεί η δράση ε, με 7 άλλες χώρες ε, με διάφορες ε, δράσεις για την πράσινη Βραζιλία και τον νόμο και την τάξη. Αλλά αυτά ήταν συνέπεια της διεθνούς πίεσης. Αν πεθάνει η Αμαζονία θα υποφέρουμε όλοι και ήδη απειλείται. Τα είπατε όλα αυτά σε μεγάλες λεπτομέρειες. Χάρηκα που αναφερθήκατε στην ανάγκη να κοιτάξουμε τη συνέπεια της πολιτικής κύριε Επίτροπε. γιατί αποψηλώνονται τα δάση για γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Ε, και έχουμε υπογράψει μια συμφωνία ε, για το εμπόριο και τη δημοκρατία και θα πρέπει οι ε, συνάδελφοι και οι χώρες του Μερκοσούρ να τα σέβονται αυτά. δεν μπορούμε ε, ως Ευρωπαίοι να κάνουμε μαθήματα σε άλλους, ούτε εμείς κάναμε πάντα τα σωστά για τα δάση και το περιβάλλον μας. Αν είμαστε πιο ταπεινοί, νομίζω θα μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με τους συναδέλφους μας στη Λατινική Αμερική και αλλού, στην Αρκτική, στην Ιδονησία, στη λεκάνη του ποταμού Κονγκού, σοβούν οι πυρκαγιές και απελευθερώνονται τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Είναι πάρα πολύ σημαντική συζήτηση και σα ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Το λόγο έχει η πρόεδρος της ομάδας, κυρία Γκαρθία Πέρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, οι ε, πυρκαγιές ε, του καλοκαιριού στην Αμαζονία ήταν πραγματική τραγωδία αυτό το γεγονός μας βήθησε σε θλίψη τη διεθνή κοινότητα και την κινητοποίηση, γιατί ο αντίκτυπο στο περιβάλλον, στα κοινωνικά και στα οικονομικά θέματα αυτής της τραγωδίας υπερβαίνει κατά πολύ τη λεκάνη του Αμαζονίου. Η Αμαζονία είναι ο πνεύμονας της υγιής ε, και έχει πάρα πολλά, πολλή βιοπικιλότητα από οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Παράγει 20% ε, του οξυγόνου. Πάνω από ένα εκατομμύριο αυτόχθονες ε, ζουν εκεί με τρόπο βιώσιμο και ε, υπερασπίζονται τη γη τους. Και το γνωρίζω αυτό γιατί είχα τη σπουδαία ευκαιρία ένα μήνα να ε, εργαστώ εκεί εθελοντικά με μη κυβερνητικέ οργανώσεις που στηρίζουν αυτές τις αυτόχθονες κοινότητες που χρειάζονται να έχουν ε, αηφόρες εναλλακτικές στον τρόπο ζωής τους και στον χώρο εκεί που ζουν ε, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν τολμώ να το σκεφτώ, με τέτοια τραγωδία. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι φλόγες έχουν ζώσει την Αμαζονία, είναι γεγονός. Αλλά σε σχέση με πέρσι αυξήθηκαν οι πυρκαγιές κατά 80% και πάνω και στα εθνικά πάρκα. Ε, επίσης η χρυσοθυρία ε, και η εξόριξη χρυσού χρησιμοποιεί υδράργυρο που είναι καταστροφή και θάνατος για περιβάλλον, ζώα, φυτά και ανθρώπους. Ε, ε, υπάρχουν αρνητές τη κλιματική αλλαγή που προωθούν αυτές τις δράσεις και τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Ο κύριος Μπολσονάρο προωθεί ε, μια νέα χρυσοθυρία, ένα πυρετό για το χρυσό και παραγνωρίζει την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια και για να το κάνει αυτό, για να μην ακούει την αλήθεια, απέλησε τους επιστήμονες της διαστημικής έρευνας και ε, του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ε, πρόεδρε, έχουμε φτάσει στο αμήν ε, με την αποψήλωση της Αμασονίας. Και πέρα από τα περιβαλλοντικά, εμείς οι σοσιαλδημοκράτες ανησυχούμε πάρα πολύ για τη μοίρα των αυτόχθων λαών, των πληθυσμών εκεί και της γης τους. προβλέπουμε και βλέπουμε σε όλη την Βραζιλία δολοφονίες ηγετών, ακτιβιστών όπως η Μέρα Γουάιπη, Δίγμα Φερέρα Σίλβα και Κλάουδιο Νόρ. Κωστάδα Σίλβα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθούμε πολύ ε, στενά τις προσπάθειες που κάνουν στην περιοχή για να βρουν λύσεις για την προστασία και των προσώπων και του περιβάλλοντος. Έχουν την πλήρη μας υποστήριξη και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε από την ομάδα μας. Ζητάμε από τον κύριο Μπολσονάρο να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κλιματικής Συμφωνίας του Παρισιού που έχει και περιβαλλοντικές ρήτρες επίσης η Συμφωνία Mercosur. Εάν ε, εξακολουθεί αυτή την τακτική η κυβέρνηση ε, θα απομονώσει ε, τη Βραζιλία. Και υπάρχει και μια παροιμία εκεί των Ινδιάνων. Μόνο όταν πεθάει και το τελευταίο δέντρο, όταν θα δηλητηριαστεί και το τελευταίο ποτάμι, όταν θα έχει πιαστεί και το τελευταίο ψάρι, τότε μόνο θα καταλάβουμε ότι το χρήμα δεν τρώγεται. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για την ομάδα Renew Europe το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Χόιζικ. Επαναλαμβάνω ότι στη διάρκεια του κύκλου των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων δεν θα δώσω μπλε κάρτες. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, κυρία Υπουργέ, ε, συνάδελφοι, ήταν ένα τρομερό καλοκαίρι όσον αφορά τι δασικέ πυρκαγιέ. Όλοι παρακολουθήσαμε συγκλονισμένοι να καίγεται ο Αμαζόνιο. Ακόμα περισσότερο όμω ε, συγκλονιστήκαμε όταν ε, ακούσαμε ε, τον ε, πρόεδρο Μπολσονάρο να επιτίθεται στι ε, ΜΚΟ που προσπαθούν να προστατεύσουν ε, τα δάση, ενώ οι δικέ του πολιτικέ έχουν συμβάλει στην καταστροφή που είδαμε. Αλλά δεν είχαμε πυρκαγιέ μόνο στον Αμαζόνιο. Φέτο είδαμε να, καίγε, να καίγονται δάση και στη Σιβηρία και στην Αλάσκα καταστρέφοντας ε, ε, πολύτιμα ενδιατήματα θα πρέπει να είναι σαφές ότι η καταστροφή των δασών είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ήρθε η ώρα όμως να παραδεχτούμε ότι είμαστε και εμείς μέρος του προβλήματος. Ε, όχι μόνο με, την, ε, με το θέμα των ε, εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και οι δικές μας πολιτικές ευθύνονται για την κατάσταση. Και ήρθε η ώρα να ε, το αλλάξουμε αυτό, να αναλάβουμε δράση. Θα πρέπει να ε, παραδεχτούμε ότι η συμφωνία με Ερκοσούρ είναι προβληματική ω έχει, αλλά απ' την άλλη θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε: Ωραία, α καταργήσουμε τη συμφωνία αυτή και όλα θα έχουν λυθεί. Όχι, πρέπει να προχωρήσουμε σε βάθο. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ισχυρίζεται ότι η Πράσινη Συμφωνία είναι η κύρια προτεραιότητά τη. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Πρέπει να ε, επηρεάσουμε το σύνολο του κόσμου. Εάν θέλουμε να είναι σοβαρέ οι προσπάθειά μα για να σώσουμε τον πλανήτη μα και τον πολιτισμό μα, θα πρέπει να φροντίσουμε οι γεωργικέ ε, πολιτικέ ε, να μην συμβάλλουν στην ε, καταστροφή των δασών. Διότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει αυτό και στον Αμαζόνιο. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι εμπορικέ πολιτικέ μα να μην συμβάλλουν στην καταστροφή των δασών, διότι το κάνουν αυτή τη στιγμή και το ίδιο ισχύει για τι ενεργειακέ πολιτικέ μα. Χρειάζεται λοιπόν να τα αλλάξουμε όλα αυτά για μας και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα των Πρασίνων. Το λόγο έχει η κυρία Χάουτελα, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτές οι εκπροθέσεις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο μας ξύπνησαν και ξέρουμε καλύτερα ότι συμβαίνουν και αλλού. Στην Κεντρική Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία. Αυτά είναι τα θερμασίμια, τα hot spots. Πιο σημαντικέ πυρκαγιέ συμβαίνουν εκεί. Και ξέρουμε για αντιμετωπιστή αλλαγή του κλίματο. Πρέπει το διοξείδιο του άνθρακο να το παγιδεύσουμε κάθε τρόπο. Και η μόνη βιώσιμη λύση σε μεγάλη κλίμακα είναι με τη βοήθεια των δασών. Όμω τα δάση μετατρέπονται σε αγροτικέ γέε. Και να είμαστε σαφεί, η συμφωνία του Μερκοσούρ έχει πρόθεση να εξαγάγει καφέ, σόγια ε, και ζώα που οδηγούν σε αποδάσωση και θέτουν σε κίνδυνο την περιοχή του Αμαζονίου. Η Συμφωνία Μερκοσούρ δεν έχει βιώσιμο μηχανισμό που θα εξασφαλίζει ότι η Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα και άλλες διεθνεί ε, περιβαλλοντικές υποχρεώσεις θα γίνονται σεβαστέ, Δεν έχει δόντι, δεν έχει κυρώσει όσον αφορά το κεφάλαιο τη βιώσιμη ανάπτυξη και να πω ότι η ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί αποδάσωσης και επιδείνωση καταστάσεων των δασών έχει μια υπόσχεση που μου δίνει κατά την απόψή μου. Να δούμε ποια ρυθμιστικά μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν επί τη ζήτηση. Χρειάζεται αυτή η νομοθεσία η ευρωπαϊκή που θα εξασφαλίζει για τους Ευρωπαίους καταναλωτές ότι δεν αγοράζουν μέσω ε, αποδάσωσης. Και εμεί είμαστε συνένοχοι έτσι. Και έχω μια ερώτηση προς Φιλανδική Προεδρία. Ξέρω ότι αποφασίστηκε ότι το Συμβούλιο Γεωργίας ασχολείται με την ανακοίνωση περί και επιδείνωση καταστασών. Γιατί μόνο το Συμβούλιο της Γεωργίας, γιατί όχι το Συμβούλιο Περιβάλλοντος Το Για την ομάδα ταυτότητας και δημοκρατίας το λόγο έχει ο κύριος Ρουζέ για δύο λεπτά και καλό και την κυρία Χάουτελα να με αντικαταστήσει στο Προεδρείο γιατί πρέπει και εγώ να πάρω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το δάσος του Αμαζονίου φλέγεται πέρα από την ε, ε, οικολογική καταστροφή που γνωρίζουμε. Ε, διαστόματος Προέδρου Μακρόν, η Γαλλία πραγματικά εξέφρασε τη συγκίνησή της και εμείς. Αλλά θα θέλαμε να συγκινηθεί το ίδιο ο κύριος Μακρόν με τις εξίσου καταστροφικές πυρκαγιές στην υποσαχάρια Αφρική. η έκτη και η ένατη μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη ε, τσακώνονται σαν παιδάκια. Ξέρουμε για ποιο λόγο καίγονται τα δάση. Από τη ΣΕΤΑ εκεί καλλιεργούν και γεές ε, ε, και έχουν ξενοτροφική δράση Καναδοί. Η Μαρίν Λεπέν και το κόμμα μα αντιτίθενται στην ΣΕΤΑ όπω και στο Μερκοσούρ γιατί είναι καταστροφική συμφωνία για του Γάλλου αγρότε. Ο πρόεδρο Μακρόν τελικά κατέληξε στην ίδια διαπίστωση και με πολύ κοινικό τρόπο άδραξε την ευκαιρία τη καταστροφή στο Αμαζόνιο για να απειλήσει ότι δεν θα υπογράψει το Μερκοσούρ. Δεν θα διαφωνήσει κανεί εδώ ότι η οικολογία και το περιβάλλον είναι πολύ σοβαρά θέματα και πολύ σημαντικά για το μέλλον ε, του κόσματος, ώστε να είναι παιχνιδάκια για εσωτερική κατανάλωση. Και στο κάτω-κάτω ας αρχίσουμε από την αυλή μας. Εμείς θα περιμέναμε από τον πρόεδρο Μακρόν να ε, σταματήσει ε, να διαλύει τον οργανισμό δασών, να κοιτάξει τι γίνεται στην νήσο Ρένιον στις πλημμύρες στη Μαγιότ, στο κίνδυνο ραδιοενέργειας της νήσους Μάρσαλ, γιατί κινδυνεύουν οι Γάλλοι συμπατριώτες στην Πολυνησία, να σκεφτεί τους Γάλλους επίσης στη Γουιάννα για να ε, συντηρήσει καλύτερα τον Αμαζόνιο, το γαλλικό Αμαζόνιο και στη θάλασσα των Σαργασών και στη Μαρτινίκα και στη Γοδελούπη. Δυστυχώς μετά από ε, όλες αυτές ε, τις φασαρίες που έχει κάνει και τους εντυπωσιασμούς δεν θα κάνει τίποτα και τελικά θα υπογράψει και το Μερκοσούρ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας η Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ κύριε Ρούζε. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Τέρτς από το κόμμα, την ομάδα μάλλον ECR. Ε, καλησπέρα σας, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά ακούω εδώ για τον Βολσονάρο να γίνεται λόγος, τον κατηγορούν για όλη την τραγωδία. Ξέρετε ότι λησμονούμε κάτι εδώ. εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε τα στραβά μάτια ε, σε σχέση με το ότι γίνεται. Ήδη εστρεβλώνουμε την αλήθεια. Ακούσαμε τώρα τους Ισπανούς σοσιαλιστές να μιλούν για χρυσοθυρία και για την καταστροφή της. Μα αυτά γίνονται κυρίως στη Βενεζουέλα, σε αυτή την περιοχή της Αμαζονίας, εκεί όπου ελέγχει τα πράγματα ο κύριος Μαδούρο και ε, οι Κολομβιανοί αντάρτες που είναι εκεί παρόντες χάρη στο κομμουνιστικό καθεστώς του κυρίου Μαδούρο και τον τζαβισμό. Αυτή τη στιγμή στην Βολιβία και έχονται 2,5 εκατομμύρια εκτάρια. Στη Βολιβία. Ποια Βραζιλία. Στη Βολιβία. Κανείς δεν μιλάει για τη Βολιβία. Διότι ο κύριος Μοράλες, ο οποίος ε, αύξησε ε, την καλλιέργεια κόκας για την κοκαίνη, η οποία έχει εκτοξευτεί η καλλιέργεια, άρχισε να καίει τα δάση γι' αυτό το λόγο. Και από εκεί ξεκίνησε μέγα τμήμα της καταστροφής. Γιατί μόνο τον Μπορσονάρο σκεφτόμαστε. Σας ευχαριστώ και τώρα ο κ. Παπαδημούλης εξ ονόματος της ομάδας του όσα μας είπε το Συμβούλιο και η Κομισιόν, αλλά και όσα μας λένε οι επιστήμονες και η πραγματικότητα, επιβάλλουν σε μας όχι μόνο λόγια, αλλά και δράση. Δεν αρκεί μια συζήτηση. Χρειάζεται να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, να πάρουμε μέτρα, να ασκήσουμε μια πίεση για να σταματήσει η αποψήλωση του Αμαζονίου και η καταστροφή του μεγαλύτερου πνεύμανα του πλανήτη και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πιστεύω όταν οι αριθμοί δείχνουν ότι επί της θητείας του μπολσονάρου έχει αυξηθεί κατά 80% μέσα σε ένα χρόνο η αποψήλωση του αμαζονίου όταν μέσα σε λίγους μήνες ο αμαζόνιος έχει αποψηλωθεί περισσότερο από ό,τι τα τελευταία τρία χρόνια πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και είναι ντροπή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η συζήτηση αυτή δεν θα καταλήξει σε ψήφισμα με ευθύνη μιας συμμαχίας των πολιτικών ομάδων της δεξιάς και της ακροδεξιάς. πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μέτρα και να αξιοποιήσουμε και το εργαλείο της μερκοσούρ για να ασκήσουμε πίεση στον ακροδεξιό μπολσονάρο. σας ευχαριστώ. Παπαδημολίου, ο κύριος Παπαδάκης ε, τώρα, μη εγγεγραμμένος. Παρακαλώ. Περιβαλλοντική καταστροφή στο δάσος παγκόσμιο πνεύμονα του Αμαζονίου είναι αποτέλεσμα της επιδρομής μεγάλων καπιταλιστικών αγροτοβιομηχανικών επιχειρήσεων, εξορυκτικών δραστηριοτήτων ομίλων ξυλίας καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που τις χρηματοδοτούν. η αντιδραστική κυβέρνηση μπολσονάρο κλιμακώνει την αντιπεριβαλλοντική πολιτική προηγούμενων κυβερνήσεων έχοντας παραδώσει την περιοχή στην επιχειρηματική εκμετάλλευση για παραγωγή βιοκαυσίμων αγροτοβιομηχανικών προϊόντων αλυσίδας εξορίξεις και ανεξέλεκτη λοτομία η αποψήλωση του αμαζονίου φέρει και τη σφραγίδα ευρωνοσιακών μονοπωλίων. γι' αυτό είναι υποκριτική ανησυχία τη ευρωπαϊκή ένωση και των κυβερνήσεών τη που έχει να κάνει και με αντιθέσει σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ευρωπαϊκή ένωση μερκοσουρ. είναι ενδεικτικό ότι παρά τα παχιά του λόγια για την κατάσταση του κλίματο το ευρωκοινοβούλιο και με την ψήφο του λαϊκού κόμματο αρνήθηκε ακόμα και να εκδώσει ψήφισμα για τον αμαζόνιο. στηρίζουμε την πάλη για να διατεθούν όλα τα αναγκαία μέσα υποδομέ και πόροι για την κατάσβεση των πυρκαγιών στον αμαζόνιο την αποκατάσταση των καταστροφών την αναδάση των καμένων εκτάσεων. να σταματήσει άμεσα στην περιοχή κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη. Τώρα έχουν το λόγο οι άλλοι ευρωβουλευτές. Ο κύριος Πέτερ Λίζα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο αποτελούν τεράστια καταστροφή. Ένα παράδειγμα να σας δώσω στην ε, Συμφωνία του Παρισιού. Ε, η Βραζιλία δεν δεσμεύτηκε να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές από ε, τη βιομηχανία ή άλλους τομείς. Η βασική οι βασικέ της δεσμεύσεις είχαν να κάνουν με τα δάση, ε, προστασία των δασών και αναδάσωση. Και αυτό δεν έχει γίνει και αυτό αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για το ε, κλίμα όλου του κόσμου. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα. Έχουμε τις πυρκαγιές στη Σιβηρία και στην Αλάσκα που είναι τεράστιο πρόβλημα για το κλίμα διότι απελευθερώνονται τεράστιες ποσότητες μεθανίου που επιβαρύνουν το κλίμα ακόμα περισσότερο και από το διοξίδιο του άνθρακα. Μερικοί ζητάνε να ε, ε, σταματήσει η συμφωνία με Ερκοσούρ. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε το εμπόριο, αλλά ε, έτσι θα έχουμε προχωρήσει, θα έχουμε μέσο πίεση, θα έχουμε τρόπο να ελέγξουμε τι κάνουν οι Κίνα και άλλοι. Φυσικά πρέπει να ε, ασκήσουμε πίεση και όχι ε, να αφήσουμε να περάσει η συμφωνία Μερκοσούρ χωρίς καμία ε, κριτική, αλλά θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μα. Χθε συζητήσαμε για τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ μπορούμε να προστατεύσουμε τα δάση μα στην Ευρώπη, πώ μπορούμε να αναδασώσουμε την Ευρώπη. Και στα δύο αυτά θέματα όμω πρέπει να δοθεί συνέπεια. Ε, είναι θετικό. Μάλλον ούτε για το ένα θέμα ούτε για το άλλο έχουμε ψήφισμα, αλλά θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Θα πρέπει μέσα στις επόμενες εβδομάδες να το κάνουμε αυτό από κοινού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λίζε. Ε, η Μίρια Μντάλη για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό που συζητούμε, μιλάμε για το μεγαλύτερο δάσος στον κόσμο το οποίο φτάνει στην καταστροφή, καταστρέφεται και φτάνουμε στο σημείο μη επιστροφή. Μα πειράζει το θέμα του Αμαζονίου γιατί πειράζει το παγκόσμιο κλίμα. Απορροφά τον άνθρακα και αυτό είναι κάτι που μπορεί μειώσει τα αποτέλεσμα τη αλλαγή του κλίματο. Αν τα δάση του Αμαζονίου πεθάνουν, πολλά αέρια του θερμοκηπίου θα απελευθερωθούν και αυτό θα επιταχύνει την αλλαγή του κλίματο. Άλλη ανησυχία. Έχουμε εκατοντάδε πυρκαγιέ που έχουν καταγραφεί φέτο στην Αρκτική και την Υπαρκτική περιοχή. Αυτέ οι πυρκαγιέ μόνο του έχουν παράγει 100 εκατομμύρια τόνου διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι ένα φαύλο κύκλο. Αν η διεθνή κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αυξήσει την προσπάθεια για περικοπή των αερίων, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δεν θα μειωθεί ο ρυθμό αλλαγή του κλίματο και θα διαδίδονται περισσότεροι φωτιέ. Μέτρα για την προστασία των δασών του Αμαζονίου είναι ένα κομμάτι τη συμφωνία που επετέθη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών Μερκοσούρ. Και είναι προ όφελο πάντων αυτέ οι διατάξει να εφαρμόζονται. Στο ίδιο πνεύμα, αυτοί που έχουν προγράψει Συμφωνία των Παρισίων και που υποσχέθηκαν να πληρώσουν οι πλούσιοι τι αναπτυσσόμενε χώρε για να φυτέψουν δέντρα που απορροφούν τον άνθρακα, πρέπει να το κάνουν αυτό. Όλοι που έχουμε ευθύνη. Πρέπει να βοηθήσουμε να αλλάξει η μορφή κατανάλωση τώρα που είναι επιβλαβή. Χρειάζεται συλλογική δράση ευρωπαϊκή και παγκόσμια που απαιτείται για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Ντάλη. Επόμενη ομιλήτρια. Ε, κύριε Στεφανούτα για 1,5 λεπτό. Ο κύριος Στεφανούτα συγγνώμη. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, όπως βλέπετε έχουμε νέους εδώ που μας ακούνε στα θεωρία και ανησυχούν περισσότερο οι νέοι από όλου μα για την αλλαγή του κλίματο. Οι δασικέ πυρκαγιέ και φυσικέ καταστροφέ δεν είναι μόνο θέμα για μεμονωμένε χώρε προ αντιμετώπιση σε απομόνωση. Ε, Δυστυχώ οι πυρκαγιέ του Αμαζονίου είναι ένα κομμάτι μεγαλύτερη τάση παγκόσμια. Ο αριθμός των πυρκαγιών στον κόσμο αυξήθηκε εν συγκρίση με πέρσι και αυτό συνέβη με εκδετικό ρυθμό. ρυθμό. Τον Αύγουστο 2018 είχαμε 16.000 πυρκαγιές. Αύγουστο 2019 79.000 πυρκαγιές. Αύξηση πάνω από 400% με άλλα λόγια. Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι στο περιθώριο όταν άλλε χώρε υποφέρουν από καταστροφέ και χρειάζεται βοήθεια. Καμία χώρα στον κόσμο ε, δεν μπορεί να γλιτώσει τι καταστροφέ. Καμία δεν ασφαλεί από αυτέ και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτέ τι καταστροφέ μόνη τη. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε συντονισμένη δράση για να σταματήσουμε αυτέ τι καταστροφέ και να ανακάμψουμε. Η επιτάχυνση αλλαγή του κλίματο και η αύξηση γενική θερμοκρασία του κλίμα του πλανήτη είναι ένα φαινόμενο. Χρειάζεται να έχουμε ανταπόκριση στα πλαίσια πολιτική προστασία και να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε με καλύτερο τρόπο φυσικέ καταστροφέ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συμπληρώνουμε τι εθνικέ προσπάθειε όταν τελικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Τα λέω αυτά διότι τώρα το Συμβούλιο έχει περικόψει αυτούς τους πόρους, κυρία Πρόεδρε, και θα πρέπει να αποκατασταθούν οι πόροι αυτοί δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τι δασικέ πυρκαγιέ. Είναι κάτι που αφορά του λαού και το μέλλον των νέων, αυτών των νέων εκεί πάνω μα ακούνε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στεφανούτσα. Επόμενος ομιλητής ο Γιάννη Ζαντζό για να 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, υπάρχουν δύο τρόποι να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ο πρώτος είναι η συγκίνηση και η καταγγελία. Πώς να μην ε, θρυνήσουμε αυτό το καταπληκτικό δάσος που καταστρέφεται. Θα χαθούν οι λαοί που ζουν εκεί. Πώς να μην καταγγείλουμε τον Πολσονάρο που είναι κλίματοσκεπτικιστής και θέλει να πουλήσει τη χώρα του και την Αμαζονία στις agro-business. Ε, και ε, το GPS, παγκοσμίω ηγέτης του Βόλου Κρέατος, τον έχει αγοράσει και αυτόν και την προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι ξενοφοβικό, ομοφοβικός, σεξιστής. Υπάρχει όμω και άλλο τρόπο να αντιδράσει που δεν καταργεί τον προηγούμενο. Να δούμε τι ευθύνη έχουμε εμεί σε αυτέ τι δαξικέ πυρκαγιέ που δεν είναι καθόλου συγκυριακέ. Κύριε Επίτροπε, καταφέρατε να μην αναφέρετε ούτε την ΚΑΠ ούτε το Μερκοσούρ. Επίτευγμα. Άκουσα εκπροσώπου του ΕΛΚ, του ΡΕΝΙΟΥ, ακόμα και σοσιαλδημοκράτε που μα είπαν ε, να σεβαστούμε τη συμφωνία του Μερκοσούρ. Καλό θα ήταν. Μα δεν βλέπετε ότι η συμφωνία συμφωνία Μερκοσούρ που υπέγραψε η Βραζιλία γιατί θα εξάγει σόγια και βόλιο κρέας, ότι αυτό διαρθρωτικά καταστρέφει τον Αμαζόνιο και την Αμαζονία και ε, είναι και κλίμα τοκτόνο συστηματικά. Αν δεν βλέπετε μια κοινή γεωργική πολιτική ε, που την υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η και Κομισιόν και θα έχει αύξηση της αγωγής βραζιλιάνικης σόγιας, ε, τότε δεν βλέπετε τις ίδιες σας τις ευθύνες και δεν συμμετέχετε στο να ε, σταματήσουν οι πυρκαγιές. Ας σοβαρευτούμε λίγο εδώ πέρα μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαντό. Η Μόλιν Πιόρκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αμαζόνιος καίγεται. Οι πνεύμονες του κόσμου που θα αποφασίσουν εάν τα καταφέρουμε ή όχι να πετύξουμε τους στόχους μας όσον αφορά το κλίμα. Ε, οι πυρκαγιέ αυτέ θα οδηγήσουν σε υπερθέρμανση του πλανήτη, κάτι που θα καταστρέψει και την βιοπικιλότητα. Ο πρόεδρος ε, της Βραζιλίας, ο Μπολσονάρο, ε, είναι συνένοχος. Όχι μόνο η πολιτική του είναι επικίνδυνη για τις γυναίκες, τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, τους αυτόχθονες λαούς και τους στοχούς Βραζιλιάνους. Η πολιτική του θέτει σε κίνδυνο το σύνολο του κόσμου η πολιτική ε, ε, καταστροφή των δασών του. Και γι' αυτό έχουν αντιδράσει πάρα πολύ και ε, απαιτούν να δράσουν. Και συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτό. Ένα προφανή τρόπο όμω είναι να παγώσουν οι συμφωνίε για τη συμφωνία Mercosur. Να την παγώσουν και να πούμε ότι είναι δεσμευτική η στόχη του παρουσιού και θα πρέπει να σταματήσει η καταστροφή των δασών του Αμαζονίου. Οι νέοι άνθρωποι περιμένουν από εμά να κάνουμε ό,τι ε, μπορούμε και εγώ πιστεύω ότι ε, θα το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πιόρκ. Η Ελεονόρα Εύη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν και για τις δασικές πυρκαγιές στον Αμαζόνιο γιατί καταναλώνουμε αυτό το κρέας, ε, ε, το φινικέλαιο, παίρνουμε ζωοτροφές, ε, σόγια, λιπάσματα Όλα αυτά οξύνουν την πίεση ε, προς τις χώρες αυτές και τα δάση τους. Εξού και η αποψήλωση. Άρα η παριθμόν ένα προτεραιότητα θα πρέπει είναι να μειωθεί το αποτύπωμα των Ευρωπαίων καταναλωτών που επηρεάζει άμεσα τα δάση και προκαλεί την αποψήλωσή τους. Ας μην είμαστε υποκριτές. Εδώ Έχουμε ένα δισεκατομμύριο κόσμο που δεν μπορεί να φάει και ένα δισεκατομμύριο που είναι παχύσαρκοι. Και τώρα ακούμε και παράγει πάρα πολύ, πάρα πολλά βιώσιμα, λίγα τρόφιμα μα, πολύ τρόφιμα και πολύ σπατάλη των τροφίμων. Και τελικά τίθεται σε κίνδυνο ο πλανήτη. Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα στη ρίζα του, στην κοινή αγροτική πολιτική και την εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αν θέλουμε πραγματικά σοβαρά να κάνουμε προσπάθεια για να πετύχουμε του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη και το πρόγραμμα του 2030 και αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη φτώχεια, την πείνα, τι ανισότητε και την εκμετάλλευση, την αδιάκριτη των διαφόρων πόρων στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Εύη. Στη συνέχεια ο κύριος Γιαρούμπας για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι ο Αμαζόνιος, η περιοχή του Αμαζόνιου είναι μια ε, φυσική σημαντική ε, περιοχή και καίγεται. Κάποιες πυρκαγιές είναι εμπρισμοί για να καθαριστεί το έδαφος για καλλιέργειες, για βοσκή. Ε, προφανώς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις απόψεις που εκφράζουμε. Έχουμε μια εμπορική συμφωνία, τη συμφωνία Μερκοσούρ και πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή για να εφαρμοστούν κάποιες διατάξεις οι οποίες εξασφαλίζουν ότι αυτές οι χώρες ε, συμμορφώνονται με τη Συμφωνία ε, των Παρισίων την προστασία του Αμαζονίου. Πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι οι διατάξεις γίνονται σεβαστές. Θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε και εφαρμογή των ευρωπαϊκών κριτηρίων όσον αφορά την κτηνοτροφία. Ναι, όπως ισχύουν στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία, να ισχύουν και εκεί. Οι ευρωπαϊκές ε, τράπεζες επενδύουν εκατομμύρια ευρώ στη Νότια Αμερική σε, για, σε περιοχές που δεν στηρίζουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Προφανώ οι διατάξει τη συμφωνία Μερκοσούρ δεν θα είναι αποτελεσματικέ αν δεν εφαρμόζονται. Πρέπει να κάνουμε κάτι για τι δασικέ πυρκαγιέ του Αμαζονίου. Πρέπει όμω να εξασφαλίσουμε ότι δεν προωθούμε αθέμητο ανταγωνισμό μέσω γεωργικών προϊόντων που έρχονται από αυτές τις ε, χώρες και δεν σέβονται τα ίδια κριτήρια τα ποιοτικά. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Γιαρούμπας. Η κυρία Κάτι Πύρη, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, οι τρομερές αυτές ε, δασικές πυρκαγιές ε, μας ε, βάζουν στο επίκεντρο ε, τις 350 εθνοτικές ε, ομάδες στον Αμαζόνιο, εκ των οποίων πέντε παραμένουν απομονωμένες. Οι συνθήκες διαβίωσής τους όμως επιδεινώνονται. Ε, και υπάρχουν ε, άνθρωποι που στηρίζονται από την κυβέρνηση που θέλουν να ε, πλουτίσουν από την καταστροφή των δασών και γι' αυτό οι πυρκαγιές αυτές δεν ήταν ατύχημα. Ε, έγιναν πυρκαγιές ε, για να ε, επιτρέψουν γεωργία και άλλη ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ έχουν αυξηθεί οι πυρκαγιές αυτές από τότε που ανέλαβε την εξουσία ο κύριος Μπολσονάρο. Στόχο έχει να οδηγήσει τους αυτόχθονε να εγκαταλείψουν την γη τους. Οι διακριτικές αυτές πολιτικές δεν έχουν δεν έχουν αντιδράσει αυτόχθονε στι πολιτικέ αυτέ. Γι' αυτό πρέπει εμεί να ενισχύσουμε τη φωνή του και να χρησιμοποιήσουμε την ισχύ μα και τα εργαλεία στην εξωτερική πολιτική για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη βιοπικιλότητα και τον πλανήτη μα. Και ε, να τελειώσω με τα λόγια του Μάρκο Μαγιουρούνα ε, που λέει ότι το δάσος δεν είναι μόνο ε, δικό μας, εμάς των αυτόχθονων λαών, είναι όλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πύρη. Ο Αντσονι Χουκ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο ουρανό επάνω από το Σαν Πάολο έχει μαυρίσει από τον καπνό των πυρκαγιών του Αμαζονίου. Τα δάση αυτά είναι οι πνεύμονε του κόσμου ε, χρειάζεται να αναπνέει η ατμόσφαιρα και οι αυτόχθονες που ζουν εκεί ε, θέλουν μόνο ε, το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να ε, τους αφήσουν στην ησυχία τους και οι πυρκαγιές αυτές καταστρέφουν τα, καταστρέφουν τα σπίτια τους. Πολλοί άνθρωποι στην Αγγλία έχουν αντιδράσει. Το, Ευρω... το Βρετανικό Κοινοβούλιο έχει κλείσει, αλλά το Κοινοβούλιο μα εδώ μας δίνει φωνή. Το ΑΕΠ αυξάνεται, έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια κατά ένα τέταρτο και ε, το θέμα είναι αν θα μπορέσουν να επιβιώσουν οι άνθρωποι εκεί. Κύριε Μπολσονάρε, αν καταστρέψετε τα δάση θα καταστρέψετε και τις δυνατότητές σας για καλή συνεργασία με την Ευρώπη. Είναι απαραίτητο να σβήσουμε τις φωτιές αυτές για να σώσουμε τον πλανήτη. Thank you very much. Ε, ε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χουκ. Σκοτ ε, Κέιτο έχει παρουσιάσει ε, μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Ναι, φυσικά. Ωραία, παρακαλώ, συνάδελφε. Ε, μισό λεπτό έχετε. Κομματική επιστολή επεστάλει στην κυρία Μάλστρομ και πολλοί στο κοινοβούλιο την υπέγραψαν και την προσοχή στην πολιτική του Μπολσονάρου κατά του περιβάλλοντο και είπαν ότι δεν πρέπει να υπογράψουμε την εμπορική συμφωνία εκτό αν υπήρχαν νομικές, νομικά δεσμευτικέ προδιαγραφέ εκεί. Εκεί οι φιλελεύθεροι δεν υπέγραψαν αυτή την επιστολή. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χουκ, είναι έτοιμο τώρα να υποσχεθεί να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ όταν δεν συμπεριλαμβάνει νομικά δεσμευτικέ διατάξει για την περιβαλλοντική προστασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κυρία Πρόεδρε, δεν γνωρίζω την επιστολή που ανέφερε η συνάδελφό μου. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που είναι πολύ περίπλοκο, ούτω ώστε να καταλήξει σε μια απάντηση να ναι, όχι, μια επιστολή. Πρέπει να εξεταστεί λεπτομερώ. Αλλά σίγουρα εγώ Πιστεύω ότι οι εμπορικέ συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, φιλελεύθερε αξίε, να προωθούν τη δικαιοσύνη και πράγματι την προστασία του περιβάλλοντο. Uh, Ευχαριστώ, συνάδελφε Χουκ. Και τώρα, η συνάδελφο Άννα Καβατσίνη έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η Αμαζονία φλέγεται Κάθε ε, λεπτό ε, πεθαίνει ένα κομμάτι από τον πνεύμονα της ε, Υφηλίου. Και ο Μπορσονάρο με την ακροδεξιά του πολιτική βάζει τα θεμέλια και ανάβει το φυτίλι για αυτές τις πυρκαγιές. Ωστόσο, ευθύνη έχει και η τη κοινότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρσι εισάγαμε 60.000 τόνους εθανόλης, 70.000 ε, ε, τόνους βόλιο κρέας και περίπου 5,5 εκατομμύρια τόνους σόγια. Ε, να μην αποψηλώνουν τα δάση εκεί η Φίλιος φλέγεται και εμείς συνεχίζουμε τον εμπρισμό γιατί η συμφωνία με το Μερκοσούρ είναι επιταχυντής σαν να ρίχνουμε βενζίνη και άλλη εθανόλη και άλλο βοιοκρέας, και άλλη αποψήλωση και άλλες φωτιές και μας ευχαριστούν ο Μπολσονάρο και το αγροτικό λόμπι. Τώρα θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας εμείς για τον πλανήτη και για το κλίμα. Οι διαμαρτυρίες στο δρόμο, α πούμε αυτή την εβδομάδα, η παγκόσμια κλιματική απεργία ε, δείχνει ότι θα πρέπει και εμείς ως Κοινοβούλιο να αναλάβουμε ευθύνες, να σταματήσουμε τη συμφωνία με το Μερκοσούρ και οι αλυσίδες διανομής να είναι ελεύθερες ε, εκμετάλλευσης ανθρώπων θα πρέπει, έχουμε το δικαίωμα και την ευθύνη να διαμορφώσουμε όλη αυτή την αλυσίδα δίκαια και σωστά. Και έχει έρθει η ώρα να το κάνουμε. Ευχαριστώ κυρία Καβατσίνη. Και τώρα το λόγο έχει κύριος Μπούσμαν από την ΚΟΕ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, εδώ και εβδομάδες σοβούν οι πυρκαγιές ε, στον Αμαζόνιο, στο Παρθένο δάσος. Πρωτοφανής, για ποιο λόγο, γιατί ε, ε, τρώμε κρέας χωρίς μέτρο. Αυτή η εμπρισμή και η αποψήλωση εγκληματική κρατάει χρόνια. Καταστρέφει φυτικά είδη και χώρο επιβίωσης των αυτοχθών. Τα ζώα καίγονται με φρικρό τρόπο, τα φυτά καταστρέφονται ε, διοξίδιο του άνθρακος απελευθερώνονται. Αυτά είναι λίγες από τις βλαβερές συνέπειες. Καταστρέφονται τα οικοσυστήματα και αυτό έχει όνομα, οικοκτονία. Και όπως τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ε, τα εγκλήματα πολέμου και οι γενοκτονίες ορίζονται από τον ΟΗΕ ως έγκλημα. Ωστόσο, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, Αγγλία, Γαλλία και Ολλανδία ζήτησε να διαγραφεί από τον κατάλογο ε, αυτό το ε, έγκλημα της οικολογικής δολοφονίας, της οικοκτονίας. Μόνο κάτι πρόστιμα τους βάζουν. Αλλά τα μονοπόλια δεν τους πειράζει το πρόστιμο γιατί είναι πολλαπλάσιο το κέρδος που έχουν από την αποψήλωση. Θα πρέπει λοιπόν να έχει ένα τίμημα σοβαρό αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μπούσμαν. Ο κύριος Χρήστοφ ε, Χάνσεν παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτό το καλοκαίρι και εγώ ήταν ο πλανήτη μας. Ε, είχαμε πυρκαγιέ στον Αμαζόνιο, στην Ασία και στην Αφρική. Ε, είχαμε περισσότερες φωτιές ε, στην Ευρώπη από ό,τι είχαν ανάμεσα στο 2008-2018 ε, και οι φωτιές στην Αρκτική σημαίνουν ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντί να κατηγορούμε τις εμπορικέ συμφωνίες όπως έκανε ο κύριος Ζαντό που ε, μετά την παράστασή του έφυγε, θα πρέπει να φροντίσουμε να εξάγουμε τα περιβαλλοντικά μας πρότυπα και να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο επίπεδο. Η Συμφωνία Μερκοσούρη είναι ε, μια μοναδική ευκαιρία να φροντίσουμε η Βραζιλία να τηρήσει τις ε, δεσμεύσεις της σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού. Θα πρέπει ε, να μηδενιστεί η παράνομη καταστροφή των δασών μέχρι το 2030, όπως είπε ο συνάδελφος Πέτερ Λίζε. Κυρίες και κύριοι, η εμπορική πολιτική δεν αποτελεί τη μαγική λύση για τα προβλήματα αυτά, σίγουρα όμως μπορεί να βοηθήσει. Μεταξύ άλλων με πολυμερεί συμφωνίε για το εμπόριο και τα περιβαλλοντικά αγαθά στα χέρια μας ε, βρίσκεται η λύση για να έχουμε ε, χρήσιμα ε, συνοδευτικά μέτρα. Η συνεργασία είναι ο τρόπος που θα πρέπει να προχωρήσουμε. Η καταστροφή αυτή που έχει προκληθεί από άνθρωπο μπορεί να βρει και λύσεις από τους ανθρώπους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Χάνσεν. Mm. Η Ιούτα Γκούτελαντ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε. Τα δάση είναι οι πράσινοι πνεύμονές μας. Τα ε, δάση του κόσμου παίζουν αποφασιστικό ρόλο για το μέλλον μας, για το κλίμα, για τη δυνατότητά μας να προσαρμοστούμε, να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον το δάσος ε, με τα, δέντρα του απορροφάει διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και γι' αυτό παίζει αποφασιστικό ρόλο ε, στην επίτευξη των ε, στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Γνωρίζουμε όμως ότι τα δάση μπορούν να συμβάλλουν με νέες τεχνικές που θα είναι αποφασιστική σημασία για την προσαρμογή μας. αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρουν τα δάση του Αμαζονίου που είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Δεν είναι τυχαίο ότι ε, ονομάζονται οι ε, πνεύμονα του πλανήτη. Δύο δισεκατομμύρια διοξίδιο του άνθρακα απορροφούν τα δάση αυτά το χρόνο, δηλαδή το 5% των συνολικών εκπομπών του κόσμου. Είναι η βασικότερη η βασικότερη πηγή για να μπορέσουμε να ε, πετύχουμε τους στόχους του Παρισιού και οι πυρκαγιές στον Αμαζονίο αποτελούν απειλή για το μέλλον μας. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, θα πρέπει να αναλάβουμε τα ηνία στην προστασία του, ε, του δάσους του Αμαζονίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκούτελαντ. Στεφάν Μπιζού, ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Προέρχομαι από τα, ήρθα από την δάφη της, της Γαλλίας και ακούγονται εκεί κραυγές ανησυχίας από το λαό της Αμαζονίας που απειλούνται από τις πυρκαγιές των δασών που είναι καταστροφικές. Όλη η ανθρωπότητα προβληματίζεται, το είπαμε, αλλά εν πρώτης περίπου 300.000 Ευρωπαίοι που ζουν στην Γαλλική Γουιάννα στο δάσος του Αμαζονιού η Γαλλία και η Ευρώπη συνεπώς έχει ένα κοινό σύνορο με τη Βραζιλία που καίει και αυτό μας δίνει μια νομιμότητα και θα έλεγα μια ευθύνη αυξημένη για να δράσουμε και για να προστατεύσουμε τον Αμαζόνιο. Βέβαια προφανώς υπάρχει ο τρόπος και ο τύπος της ταχείας δράσεως. Είναι ένα θέμα κατεπήγων, αλλά να δράσει κανείς μέσα διαδικασίας κοινοβουλευτικής που διαθρώνεται και συντονίζεται σωστά είναι ένα θέμα συνοχής και αποτελεσματικότητας. Λοιπόν, Μα ζητείτε να χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι μοχλοί, ώστε στον Αμαζόνιο να έχουμε στατηγική και απέτηση για το σεβασμό των στόχων της ανάπτυξη βιώσιμη, το σεβασμό του έφταυστου χαρακτήρα τη βιοπικιλότητας, να γίνει σεβαστή η ισχύ των τοπικών, των τόπιων πληθυσμών και το σεβασμό τη πολιτιστική του κληρονομία και να γίνουν σεβαστέ οι δεσμεύσει που ανελήθησαν στη Συμφωνία των Παρισίων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπιζού και τώρα επόμενος ομιλητής είναι ο Μπάς Άικχαουτ ε, που έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συγκλονίστηκαν όταν είδαν αυτά που είδαμε αυτό το καλοκαίρι στι πυρκαγιέ του Αμαζονίου και σωστά συζητούσαμε την εμπορική συμφωνία του Μερκοσούρ, η οποία έχει στόχο τη βελτίωση και τη βελτίωση του εμπορίου μεταξύ Βραζιλία και Ευρώπη, Φερρυπίν. Αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι κατηγοριών. Το λέω αυτό προ τα μέλη του ΕΛΚ. Διαβάστε τι λέει η συμφωνία. Αν δείτε τι γίνεται για την πρόληψη τη αποδάσωση στην εμπορική συμφωνία του Μερκοσούρ, θα βρείτε κάπου, κάπου στο κεφάλαιο για εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη μια αναφορά και το μόνο που αναφέρεται είναι να ενθαρρύνουμε εμπόριο και προϊόντα από δάσος που βιώσιμα το διαχειρίζονται και να προωθήσουμε τη συμπερίληψη, τον, ε, την κάλυψη των τόπιων πληθυσμών και των ενθαγενών. Μιλάμε για ενθάρρυνση και προώθηση. Η υπόλοιπη συμφωνία είναι πολύ δεσμευτική. Αυτό δείχνει ότι αυτή η εμπορική συμφωνία έχει πολύ παράδοξο καθορισμό προτεραιοτήτων. Περισσότερο εμπορίο και όταν μιλάει για βιωσιμότητα, προώθηση και ενθάρρυνση. Αυτή είναι η διατύπωση που χρησιμοποιούμε. Και αυτό είναι το ερώτημα που ευθύνω και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θέλετε να αλλάξει η διατύπωση του ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε θεσμευτικού κανόνε που ισχύουν αντί αυτή, αυτά τα πολύ ισχνά κεφάλαια που έχουμε στην παρούσα συμφωνία την εμπορική του Μερκοσούρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάουτ και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Εμμανουέλ Μογέλ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προφανώς όλες και όλοι μας έχουμε μείνει άναυδοι με την κατάσταση στην Αμαζονία, αλλά δεν μπορούμε να ε, αναλωθούμε στις καταγγελίες, στις καταδίκες. Θα πρέπει να βγάλουμε και πολιτικές συνέπειες και συμπεράσματα γνωρίζοντας τα αίτια. Και το πρώτο αίτιο είναι η εγκληματική πολιτική του κυρίου Μπολσονάρο που διαλύει τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, καταστρέφει τους αυτόχθονες και χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τοξικά φυτοφάρμακα με τις agro εκεί στη Βραζιλία που βασίζονται στις εξαγωγές και χρειάζονται όλο και περισσότερες γέες, επιφάνειες για να καλλιεργούν σόγια. Ποια είναι η δική μας ευθύνη, ας σταματήσουμε τις ε, ε, υποκρισίες. Άκουσα έναν δεξιό συνάδελφο που είπε ότι το μέρκοσουρ θα αναγκάσει τον κύριο Μπολσονάρο να είναι ενάρετος. Πλάκα μας κάνετε. Περισσότερη εθανόλη, περισσότερη ζάχαρη, περισσότερο κρέας. Τα γράφει αυτά η συμφωνία. Άρα είναι τεράστιο κίνητρο για την αποψήλυψη. Ε, αποψήλωση των δασών. Α είστε λογικοί και συνεπεί συνάδελφοι από το Ρινιού και τη δεξιά. Απορρίψτε το Μερκοσούρ. Ευχαριστώ τον κύριο Μορέλ. Τότ. The mic is working. Okay. Δουλεύει το μικρόφωνο. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει κυρία Τότ. Ε, κοιτάξτε, είδαμε τις καταστροφικές περκαγιές ε, των δασών ε, και συζητούμε για τον Αμαζόνιο και τα όσα συμβαίνουν εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η καταστροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει βοήθεια και οικονομική και τεχνική ε, σε όποιον τη χρειάζεται. Η αποψήλωση των δασών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλοι από κοινού. Αλλά να ξέρουμε και τι κρύβεται από πίσω και τους εμπορικούς λόγους και τους υπόλοιπους. Χάρηκα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί προτεραιότητα την προστασία των δασών. Και στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τονίσει ότι όλα αυτά που, κάνει, που εξαγγέλει μάλλον τα υλοποιεί. θα πρέπει να αναλάβει σημαντική δράση για να προληφθούν τέτοια φαινομένα στο μέλλον. Το ζήτημα είναι παγκόσμιο να αναχαιτιστεί η αποψήλωση των δασών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της θα πρέπει ε, να προχωρούν σε αναδάσωση. Στην Ουγγαρία αυτό θεωρείται προτεραιότητα και φέτος η αναδάσωση ήταν ε, διπλάσια από ό,τι στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Τότ. Μπουρκάρτ, ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο αποτελούν καταστροφή όχι μόνο για, για τη φύση, ε, είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δράσης, ε, διότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι λιγότερο κερδοφόρα. Η κατανάλωσή μας ε, είναι υπεύθυνη, συνυπεύθυνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει αναγνωρίσει αυτό στην ανακοίνωσή τη. Ε, τώρα όμως θα πρέπει να δούμε δράση. Δεν θα πρέπει να συμφωνήσουμε με καμία συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Μερκοσούρ εάν δεν έχουμε προστασία των δασών, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίτευξη των στόχων του Παρισιού. Τα, μέχρι στιγμής ε, δεν είδαμε αποτελέσματα. Τα δάση θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο ε, εάν θέλουμε να, να εμποδίσουμε την ε, αλλαγή του κλίματος και την καταστροφή της βιοπικιλότητας. Ε, θα πρέπει ε, να επιμείνουμε στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθούν στον δρόμο, διότι ε, προς το παρόν μόνο λόγια έχουμε να τους προσφέρουμε, αλλά θα πρέπει να μην τους απογοητεύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπόρχαρτ και τώρα η κυρία από το Ρήνιο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω να προεδρεύετε σε αυτή τη συζήτηση ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ και τον Επίτροπο Βέρα, Βέλα, συγγνώμη, θα είναι από τις τελευταίες συζητήσεις του μάλλον. Ο Αμαζόνιος φλέγεται, καταστρέφεται το μεγαλύτερο δάσος του κόσμου, ε, φλέγεται και η κοινή γνώμη και δυναμητίζονται οι διπλωματικές σχέσεις. Η Αμαζονία που φλέγεται σημαίνει ότι ε, ε, κινδυνεύει από ασφυξία μια ολόκληρη περιοχή. Οι πρόεδροι Μοράλες και Βολσονάρο φέρουν τεράστια ευθύνη. Είναι φαύλος ε, κύκλος. Αντί να απορροφούν άνθρακα, τα δάση αυτά ε, ε, απελευθερώνουν στο περιβάλλον διοξίδιο του άνθρακα που έχουν αποθηκεύσει και δεσμεύσει εδώ και αιώνε. Όλα αυτά τα προϊόντα, το φινικέλαιο, το, η ξυλία, το βόιο κρέα και φυσικά η σόγια, ένα στα δέκα προϊόντα συνδέεται με την αποψήλωση και καταναλώνεται στην Ευρώπη. Τελειώνω. Η απάντησή μα θα πρέπει να είναι στο ύψο των περιστάσεων και εγκάρσια. Δεν φτάνει ε, να πω όλα τα μέτρα, ένα μέτρο, ένα σήμα, ένα σήμα πιστοποίησης να δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ταυτοποιούνται και να προωθούνται τα προϊόντα που συνδέονται με μηδενική αποψήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρίς. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Τουσά, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι καίγεται η περιοχή του Αμαζονίου και οι πυρκαγιέ και είναι και το τελευταίο φράγμα κατά τη αλλαγή του κλίματο. Ο πολλαπλασιασμό των πυρκαγιών δεν συνδέεται μόνο με την ξηρασία, συνδέεται με τα οικονομικά συμφέροντα που θυσιάζουν τα δικαιώματα τη φύση. Στην Αμαζονία, λοιπόν, απο, απαλωτιώνουν εδάφη, αποδασώνουν, προσπαθώντα να πετύχουν κέρδη. Να μην κοιτάμε αλλού. Ε, σαν να είμαστε αδιάφοροι. Αυτέ οι επιχειρήσει, οι αγροτροφημικέ ή αυτέ οι εξορυκτικές είναι και ευρωπαϊκέ. Αυτέ οι επιχειρήσει σήμερα από κανέναν κανόνα δεν δεσμεύονται, κανένα καθήκον επαγρύπνηση και ελέγχου. Και ανάμαστε στου βασικού ρηπαντέ του κόσμου, πώ μπορούμε να ανεχθούμε ότι το ΤΑΛ και η ΣΕΛ αυτέ οι δύο εταιρείε πετρελαίου ευρωπαϊκέ δεν πρέπει να, συμφωνούν, να συμμορφωθούν με τη Συμφωνία των Παρισίων. Πρέπει να δράσουμε. Όταν Ευρώπη θα, πότε θα αναγνωρίσει το δικαίωμα τη φύση Ευρώπη πλέον τη, τη δολοφονία του κλίματος, τα δικαιώματα του πλανήτη. Μιλάτε για την προάσπιση του τρόπου ζωής μας. Σας ρωτάω, πώς θα, μπορέσετε να επεσταστείτε έναν τρόπο διαβίωσης που θα συνάδει με το μέλλον μας. Θα πρέπει να σεβαστούμε ε, τα όρια του πλανήτη και τα περιθώρια που μας δίνει ο πλανήτης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τωσά. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Ρέγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε φλέγεται ο Αμαζόνιος και ο πλανήτης ε, χάνει χρόνο, τελειώνει ο χρόνος. Αυτή τη στιγμή με και με τη σοβαρή οικολογική κρίση θα πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά. Ακούσαμε τον αντίκτυπο αυτών των περικαγιών. Χάνεται η βιοποικιλότητα, καταστρέφεται το δάσος για να προωθηθούν ε, τα συμφέροντα της κρεοπαραγωγής. Χάνουν τα εδάφη του οι αυτόχθονε κοινότητε και βλέπουμε και την ανικανότητα του Μπολσονάρο και τη ακροδεξιά κυβέρνησή του. Δεν μπορούν με σοβαρότητα και ευθύνη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Το μόνο που του νοιάζει είναι να μοιράσουν την πίτα ανάμεσα στου ολιγάρχε. βεβαίω με τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη εμπορική πολιτική. Δεν αρκεί να στέλνουμε ευρωπαϊκά κονδύλια και πολύ λιγότερο να τα διαχειρίζεται αυτό ο φασίστα. Θα πρέπει να ε, δούμε ποιε είναι οι συνέπειε του οικονομικού μοντέλου. Προηγουμένω ζήτησε προτάσει εκπρόπως του Συμβουλίου. Σα δίνω προτάσει. Να παραλύσει η Συμφωνία Μερκοσούρ, γιατί είναι τμήμα του προβλήματο. Να σταματήσουμε τι μαζικέ εισαγωγέ κρέατο και να μην έχουμε τέτοια παραγωγή και τέτοια κατανάλωση που πιέζουν τόσο το πλανήτη και να σταματήσουμε να είμαστε συνένοχοι αυτών που σπαίνουν το θάνατο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ρεύο και τώρα να πω το εξής. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι έχουμε 20 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο και δεν έχουν λάβει το λόγο και είναι πολύ σημαντική και έχουμε τόσα πολλά αιτήματα, 12 αιτήματα εκτός του καταλόγου των ομιλητών. Και θα ήθελα να διαβάσω τα ονόματα εκείνων στους οποίους θα επιτραπεί να έχουν χρόνο αγόρευσης εκτός του καταλόγου των ομιλητών. Η εξής. Agius Saliba, Auram, anteeksi, Joveva, Keleger, Chowns ja Kanjesna. Ja valitettavasti te tulette... Και δυστυχώς πρέπει οι υπόλοιποι από εσά να απογοητευτείτε. Δεν μπορώ να σα δώσω το λόγο. Επόμενη παρέμβαση από την κυρία Μπέντελε. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό, κυρία Μπέντελε. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, οι ειδήσει και οι εικόνε από τον Αμαζόνιο ήταν τρομερέ. Ε, το τόνισαν αυτό αρκετοί από του προλαλήσαντες. Ε, και ε, αν σκεφτούμε ότι οι δάση καίγονται όχι μόνο στη Νότια Αμερική, αλλά ότι έχουμε καταστροφή δασών και στη Σιβηρία, την Αλάσκα και στην Αφρική, θα πρέπει να αναρωτηθούμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε αυτήν την απαραίτητη καταβόθρα διοξιδίου του άνθρακα. Και ε, ε, ε, κατά την εκπόνηση εμπορικών συμφωνιών η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον θα πρέπει να φροντίσει να εκμεταλλεύεται το βάρος και των 28 κρατών μελών για να πετύχει αυτά που θέλει. Η προστασία του κλίματος θα πρέπει να αποτελεί μόνιμο συστατικό της ε, αναπτυξιακής πολιτικής μας. Βρισκόμαστε τώρα στην αρχή μιας νέας θητείας, μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει τα καθήκοντά της και ειλικρινά εμένα μου λείπουν από τις δηλώσεις ε, Μπορέλ και ε, ε το κλίμα και το περιβάλλον. Θα πρέπει μάλιστα να προωθήσουμε τις πολιτικές αυτές όχι μόνο εσωτερικά αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν στην αναπτυξιακή συνεργασία μας ε, να φροντίσουμε να παρέχουμε πόρους ε, για το περιβάλλον. Η Πρόεδρος Διακόπτη έχετε υπερβεί το χρόνο σας. Θα πρέπει λοιπόν να διαμορφώσουμε ανάλογα το νέο μέσο μας για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Σάντος. Σας παρακαλώ ε, να περιορίζεστε στο χρόνο ομιλία σας, ε, διότι αρκετοί ομιλητές δεν θα μπορέσουν καθόλου να πάρουν το λόγο. Σάντος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Οι δασικές πυρκαγιές στην περιοχή του Αμαζονίου ε, επιζητούν την προσοχή μας, όχι μόνο λόγω της καταστροφής που προκαλούν, που καταστρέφουν τους πνεύμονες του πλανήτη, αλλά και λόγω της παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αυξάνονται με αστρονομικό ρυθμό. Είδαμε ανεξέλεγκτες βιοπραγίες κατά των Ιθαγενών και είδαμε ότι δύο ηγέτες των Ιθαγενών δολοφονήθηκαν, που ήταν ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των Ιθαγενών. Δύο λοιπόν αρχηγοί δολοφονήθηκαν το μήνα Ιούνιο των πληθυσμών αυτών. Υπάρχει μακρύ κατάλογο τέτοιων ακτιβιστών και θα πρέπει αυτό να χτυπήσει το κουδούνι του συναγερμού περί των τεκτενομένων. Υπήρξαν απειλέ, υπήρξαν παρενοχλήσει, βιοπραγίε. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε μια στεναρή απάντηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ηγέτες, οι πολιτικοί τη Βραζιλία είπαν ότι θα κάνουν περισσότερα, ε, θα κάνουν περισσότερες διερευνήσεις για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εξορίξεις στον Αμαζόνιο. Βλέπουμε ποια θα είναι η πολιτική εκμετάλλευση στον Αμαζόνιο. Θα πρέπει να ανησυχούμε για τα δικαιώματα των ηθαγενών πληθυσμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αγνοεί τις υποχρεώσεις που έχει σαν ηγέτης στο παγκόσμιο προσκήνιο και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να μπορέσει να υπερασπίσει και να προστατεύσει τα δάση του Αμαζονίου και το περιβάλλον και να εξασφαλίσει το ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης θα τύχουν προστασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Σάντος. Και τώρα, επόμενος συνάδελφος είναι η κυρία Κάλσμπρο. Κυρία Πρόεδρε, ο Αμαζόνιος καίγεται. Είναι μια ε, οξία κρίση για το σύνολο του κόσμου. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο έχει δείξει ότι δεν ε, θα ασχοληθεί με την ε, πρόκληση ε, για το κλίμα και τη διατήρηση των δασών. Μάλιστα είπε ότι θέλει να αποσυρθεί από την Συμφωνία του Περισιού μαζί με τον Ντόναλτ Τραμπ. Ακούστηκαν ε, διαμαρτυρίε ε, από το υπόλοιπο του κόσμου, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, οι οποίες όμως είχαν και κάποιο αποτέλεσμα. Θέλουμε να φροντίσουμε να τηρηθεί η Συμφωνία του Παρισιού. Αν θέλουμε να σώσουμε τον Αμαζόνιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μα. Η Συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μερκοσούρ είναι σημαντική και για εμά και για την Βραζιλία. Είναι όμω και μια μοναδική ευκαιρία να ασκήσουμε πίεση και να δημιουργήσουμε κίνητρα για την κυβέρνηση ε, της Βραζιλίας ε, για να αναλάβει δράση. Είναι λοιπόν ε, ένα από τα καλύτερα και πιο αποτελεσματικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ας το χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Κάρλσπρο. Γκερέιρο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, Επίτροπε, τα γεγονότα είναι σαφή, τα στοιχεία είναι σαφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη ευθύνη για την καταστροφή των δασών, δασών του Αμαζονίου λόγω γεωργικής παραγωγής και ως εισαγωγέας ε, σόγιας από τη Βραζιλία. Αυτά που τρώμε καταστρέφουν τελικά εν μέρη τον Αμαζόνιο και έχουν αντίκτυπο και για τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Γι' αυτό κυρία Υπουργέ και Επίτροπε θα θέλαμε να δούμε η συμφωνία του Μερκοσούρ να μπλοκάρεται και να σταματήσουμε εισαγωγέ κρέατος και σόγιας από αυτή την περιοχή του κόσμου. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά είναι υψή τη σημασία να γίνει αυτό για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον Αμαζόνιο και τη βιοπικιλότητα εκεί και του διάφορου αυτόχθονε πληθυσμού που ζουν εκεί. Σα ευχαριστώ, κύριε Γκερέιρο. Επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Βάλλα που έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η παραγωγή βοηού κρέατος αμφισβήτηταν η μεγαλύτερη αιτία για τη αποδάσωση στον Αμαζόνιο. Και είναι λογικό ο ταχύτερο τρόπο να σταματήσει η αποδάσωση του Αμαζονίου θα είναι να μειώσουμε τη ζήτηση για το βραζιλιανό κρέα, το βραζιλιάνικο κρέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πλημμυρίσει την ευρωπαϊκή αγορά με περισσότερο κρέα από τη Νότια ε, Αμερική μέσω τη Μέρκοσουρ. Λοιπόν, 80% από τη σόγια που καταναλώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τη Βραζιλία. Υπάρχουν περιορισμοί για την παραγωγή ε, τη ε, σόγια αλλά αυτό ε, τελικά αυξάνει τελικά την πίεση από την κτηνοτροφία. Λοιπόν, αντικαταστήθηκε η κτηνοτροφία τελικά από καλλιέργεια σόγιας και γι' αυτό τελικά από μια περιοχή πήγανε αυτοί οι καλλιεργητές οι σόγιας από εκεί που αφήσαν τις περιοχές τους πήγαν στην περιοχή του Αμαζονίου. Έχει γίνει λοιπόν εκτοπισμός και μετακίνηση των κτηνοτρόφων. Τον Μάρτιο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς στα κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα, πώς κατέληξε στη συμπέρασμα ότι η παραγωγή σόγιας δεν δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά την αλλαγή της χρήσης των γεών. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατέληξε αυτό το συμπέρασμα λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα και αυτά που πραγματικά συμβαίνουν εκεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στη συνέχεια το λόγο έχει η κυρία Κολέα Έστερλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε με τις εμπορικές συναλλαγές φέρουμε και εμείς το τμήμα της ευθύνης για τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο διότι εισάγουμε τα προϊόντα από την αποψήλωση και την καταστροφή των δασών, βόλιο κρέας και σόγια συγκεκριμένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ένα στεναρό μήνυμα, αλλά να επιβάλλει και βιώσιμη διαχείριση του δάσους με δεσμευτικές ρήτρε που να σέβονται το, τη Συμφωνία για το Κλίμα, γιατί σήμερα δεν προβλέπεται καμία κύρωση. Στις διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ είναι εκ των όνων κάνευ αυτό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε και τους οικολογικούς φραγμούς που ήταν προεκλογική μας ε, εξαγγελία και δεσμεύτηκε η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν και χαιρόμαστε. Πώς θα γίνει αυτό όμως προχωρώντας στις διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές μας, να ε, στηρίξουμε τους παραγωγούς και τις βιομηχανίες απέναντι στους ρηπαίνοντες από τις τρίτες χώρες. Σήμερα αυτό δεν γίνεται με τη Συμφωνία Μερκοσούρ και θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ε, για την κατάσταση στην Αμαζονία. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ και εγώ κυρία Κολάνστερλε. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Φαμπρέμπτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Γεια σας αγαπητέ Επίτροπε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω σε αυτή τη ε, σημαντική συζήτηση. Διαπιστώνω πάρα πολύ ότι υπάρχει εδώ διακομματική συμφωνία. Είμαστε ομόφωνοι για το τι συμβαίνει στον Αμαζόνιο. Και άρα συμπεραίνω ότι μπορούμε να αναζητήσουμε και να βρούμε ομοφωνία ε, στη λύση που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αλλά ένας κρίσιμος τρόπος να το αντιμετωπίσεις είναι η εμπορική πολιτική. Να την ε, ξανασκεφτούμε εκ βάθρων με τους βιώσιμους στόχους, τις στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, να τους παίρνουμε σοβαρά και να φροντίσουμε να σταματήσει η αποψήλωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν ε, το TST κεφάλαιο βιωσιμότητας που θα πρέπει να είναι πραγματικά δεσμευτικό ε, στις συμφωνίε. Αλλά εμεί ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να φροντίσουμε να έχει και δόντια αυτή η συμφωνία. Δηλαδή να λέμε από την αρχή τη συζήτηση ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η αποψήλωση και ε, να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βραζιλία. Και από εκεί και πέρα συζητάμε την οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία. Ε, ας το κάνουμε αυτό τα επόμενα χρόνια και να τους τρίξουμε και τα δόντια λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μπιλμπάο Μπαραντίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κύμα των πυρκαγιών που είδαμε φέτος στον Αμαζόνιο και τους αυτόχθονες λαούς έχει επιπτώσει σε όλους μας και μας επηρεάζει και επίσης από οικονομικής απόψεως είναι τρομακτικό γιατί υποτίθεται ότι είναι αναπτυξιακή αυτή η προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, υπάρχει και ένα σύμφωνο στις 6 Σεπτεμβρίου ε, από διάφορες χώρες εκεί της περιοχής για τον Αμαζόνιο και δεσμεύονται χώρες αυτές ε, με τις διεθνείς συνθήκες να προστατεύουν το περιβάλλον και ιδιαίτερα τη Συμφωνία των Παρισίων. Θα πρέπει εμείς να ενθαρρύνουμε αυτή την κίνηση, γιατί οι πολιτικές πρόληψης, κατάσβεσης και ε, αναδάσωσες θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές. Εμείς θα πρέπει να εισάγουμε προϊόντα ε, που έχουν παραχθεί με σωστό τρόπο και τα υπόλοιπα να απαγορεύονται, να μην πολλούνται πουθενά, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό, ε, να είναι πρώτα οι αξίες και μετά τα συμφέροντα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πιλιπάο. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Οσάλιβαν. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Πρόεδρε. Με τρόμο παρακολουθήσαμε τις καταστροφικές ε, πυρκαγιές στον Αμαζόνιο αυτό το καλοκαίρι, ε, που μάλιστα ενθάρρυνε το καθεστώς Μπολσονάρο. Η η παγκόσμια κατανάλωση, η ζήτηση για ε, φτηνό βόλιο κρέας ε, βρίσκονται στην καρδιά της καταστροφής αυτής. Θα πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε στην κατάσταση αυτή και ε, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται και με το θέμα του εμπορίου και τις πολιτικές που έχουν οδηγήσει στην καταστροφή των δασών ε, καθεστώς ο Μπολσονάρο τιμωρεί τις ε, ε, αλλά αυτό δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί όπως και η παραβίαση διεθνών ε, συμφωνιών. οι ε, τάσεις ανάπτυξης ε, ε, συγκρούονται με την ανάγκη προστασίας του Αμαζονίου. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θα υπάρχουν θέσεις απασχόλησης σε ένα νεκρό πλανήτη. ελάχιστε θέσεις απασχόλησης όμως υπάρχουν και σε τεράστιες φοιτίες που στόχο έχουν το μέγιστο βραχυπρόθεσμο κέρδος. Ελπίζω λοιπόν το Κοινοβούλιο να απορρίψει τα μέτρα αυτά και να εγκρίνει το ψήφισμα που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Οσάλιβαν. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Φερνάντης, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να πολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος και αυτό χρειάζεται μια παγκόσμια συντονισμένη δράση. Τα δάση θα είναι πολύ σημαντικά στην προσπάθεια αυτή. Η βιωσιμότητα θα πρέπει να είναι η λέξη κλειδί. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και αλληλεγγύη. Πρέπει να σεβαστούμε τα δάση του Αμαζονίου. Είναι μια τεράστια έκταση. Εννέα χώρες καλύπτονται, όχι μόνο η Βραζιλία. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και εμείς πυρκαγιές. Έχουμε αυτή την εμπειρία. Θα μπορούσαμε να είμαστε παράδειγμα και για τον υπόλοιπο κόσμο. Στη χώρα μου, το 2017, είχαμε εμπειρία πυρκαγιών και χάσαμε και πάρα πολλέ ζωέ κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εστιάσει προσπάθειε επί επιπρόληψης και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να συνεργαστεί ε, και να χρηματοδοτήσει προγράμματα, να διαθέσει κατάλληλους πόρους, ούτω ώστε στην περιοχή του Αμαζονίου, αλλά και σε άλλα δάση, να υπάρχει προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να εστιαστούμε επί της βιωσιμότητας και αυτό είναι ένα απόσπαστο κομμάτι των ευθυνών που έχουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Φερνάντες. Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος Λουένα που έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ναι, καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, ε, η συζήτηση αυτή που κάνουμε έχει να κάνει με την εκμετάλλευση των δασών και την ε, καταστροφή τους. Και το είπε και η ε, Προεδρεύουσα. Θα πρέπει να ε, δείξουμε ηγετικό πνεύμα. Το θέμα είναι εάν μπορούν με βιώσιμο τρόπο να ε, συγκεραστούν τα συμφέροντα. Έχουμε δασική στρατηγική όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι τα προϊόντα αυτά που καταστρέφουν τα δάση δεν τα εισάγουμε, τα περιορίζουμε. Δίνουμε μάχη αγαπητοί συνάδελφοι απόψε απέναντι ε, σε πραγματικούς αρνητές της κατάστασης. Αλλά μπορούμε να το κερδίσουμε αυτό δείχνοντας ηγετική στάση, συνέπεια ε, και χωρίς να παρετούμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κατάινα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι δασικές πυρκαγιές μας θυμίζουν ε, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, για παράδειγμα στη Συμφωνία Μερκοσούρ, ε, καθώς και τη Συμφωνία της Συμφωνίας του Παρισιού. Θα πρέπει να φροντίσουμε η Συμφωνία Μερκοσούρ να εφαρμοστεί σύντομα, σύμφωνα με τις αρχές ε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί θα πρέπει να γίνουν σεβαστά και θα πρέπει να φροντίσουμε το εμπόριο να βασίζεται σε διατάξεις ωφέλιμες και τις δύο πλευρές. Η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δείχνει ότι η αποψήλωση των δασών είναι όλο και λιγότερο πρόβλημα στην Ευρώπη. Τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, ε, κάνουν αναδάσωση, αλλά δεν υπάρχει αρκετά καλός συντονισμός. Η επικαιροποίηση της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση είναι πιο σημαντική σήμερα από ποτέ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, επόμενος ομιλητής, ο κύριος Χόλμγκρέν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα τη δυνατότητα να συναντηθώ με δύο εκπροσώπους ε, της ε, ε, ε του Αμαζονίου, ε, των οποίων η ε, πόλη κάηκε και θα πρέπει ο αγώνας τους να είναι ο δικός μας κοινός αγώνας. Καίγεται ο Αμαζόνιος. Ταυτόχρονα ο πρόεδρος Μπολσονάρο απειλεί ότι θα εγκαταλείψει τη Συμφωνία του Παρισιού ε, και θα ε, διευρύνει την αποδάσωση του Αμαζονίου, κάτι όμως που πρέπει να σταματήσει τώρα αμέσως, διότι ε, είναι το πιο ευαίσθητο ε, μέρος ε, του πλανήτη μας. Και επίσης θα πρέπει να υποτιμήσουμε τις συνέπειες ε, για τους αυτόχθονες λαούς. Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στις χώρες Μερκοσούρ και θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορεί να φροντίσει οι χώρες αυτές τώρα αμέσω να επιλέξουν να προστατεύσουν ε, τα δάση για να μην χάσουν το εμπόριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Χόλμκρεν. Ο κύριος Πέρν Χούμπερ, ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, από τις αρχές του έτους 6.000 ε, ε, ε, έχει, έχει καεί μια έκταση που αντιστοιχεί στο 80% της χώρας μου, της Αυστρίας. και ε, στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν οι εκτάσεις αυτές για τη γεωργική παραγωγή. Έτσι θα δημιουργηθούν τεράστιες εφητείες που δεν μπορούν να συγκριθούν με τις δικές μας. Ε, η σχέση με τη Συμφωνία Μερκοσούρ ε, είναι άμεση και είναι ντροπιαστική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την καταστροφή ε, των δασών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη να τηρήσουμε τους στόχους ε, ε, για το κλίμα και ταυτόχρονα να εισάγουμε προϊόντα από τις χώρες Μερκοσούρ τη στιγμή που ήδη έχουμε αρκετά περιφερειακά προϊόντα σε επαρκείς ποσότητες. Εάν ε, η ε, βραζιλιάνικη κυβέρνηση συνεχίσει προ την ίδια κατεύθυνση, προτείνω την απαγόρευση τη εισαγωγή βόλιου κρέατος από τι ε, χώρε Μερκοσούρ, όπω ήδη έχει προτείνει η Φιλανδική Προεδρία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόγια έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε καίγεται η περιοχή του Αμαζονίου και, και αν καίγεται η γη που παράγει το 20% του οξυγόνου που αναπνέμε και διάφοροι και κληρονομιά, πολιτισμοί, πληθυσμοί, βιοπικιλότητα καίγονται. Οι άνθρωποι δημιουργούν τις πυρκαγιές, οι ηγέτες που εκμεταλλεύονται τους πηγές και τους ανθρώπους βάσει του παλιού καπιταλισμού χωρίς βιωσιμότητα που προωθεί την ευημερία όλων. Υπάρχει μια έκφραση στην ντόπια γνωσή που, που λέει πάνω κάτω ότι πώς είναι η καλή ζωή, πώς μπορεί να ζει καλά. Αυτό τον τρόπο του εφζίν θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε και στην πολιτική μας και στις πολιτικές της Ένωσης. Γιατί δεν μπορούμε το θάρρος να επανεξετάσουμε και τη συμφωνία του Μερκοσούρ να έχουμε πιο αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας περιβαλλοντικής. Δεν έχουμε το θάρρος να πούμε ότι δεν μπορούμε να, να κάνουμε τους περιβαλλοντολόγους με τα δάση άλλων των χωρών των αναπτυσσοπμένων. Είναι ένα πρόβλημα δικό μας. Θα πρέπει να συμβάλλει η Ευρώπη σε ένα σχέδιο για την αναδάσωση της περιοχής αυτής. Σας ευχαριστώ κυρία Τόγια. Επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Μέτς που έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από το 1990 μέχρι το 2016 χάσαμε 1,3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα δασών. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 800 γήπεδα ε, ποδοσφαίρου την ώρα. Αυτή η καταστροφή αφήνεται στη ζήτηση τροφίμων και ε, ζωοτροφών στον κόσμο. Εισάγουμε σόγια γενετικά τροποποιημένη ενθαρρύνοντα τη χρήση την τεράστια παρασιτοκτόνων για να θρέψουμε τα ζώα μας. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πουθεν, πουθενά δεν προτείνει μια στατική προστασία στον δασών. Από τη μία πλευρά θέλει προστασία των δασών και προτείνει τα άλλα. Από την άλλη πλευρά η ΚΑΠ ενθαρρύνει την εντατική καλλιέργεια και την μαζική εισαγωγή ζωοτροφών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει εξίσου μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, τη Μέρκοσούρ που θα επιδεινώσει την κατάσταση. Η Αμαζόνια επί δύο εβδομάδε καίγεται. Τέτοια έκταση σε βαθμό που την έβλεπε κανεί από το διάστημα να καίγεται. Έχουμε και εμεί ευθύνε. Α είμαστε συνεκτικοί να μην χρησιμοποιούμε τα προϊόντα που προέρχονται από την αποδάσωση και να μην εθαρρύνουμε τον Πολσονάρο να θυσιάζει τα δάση του Αμαζονίου και τους κατοίκου για τον αγροτροφημικό τομέα, για τη βιομηχανική παραγωγή τροφίμων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μέτς. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Σπυράκη για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, όλοι εδώ σε αυτή την αίθουσα ζητάμε επιγόντω μέτρα για τη βιώσιμη διαχείριση του Αμαζονίου, διότι αν η καταστροφή ξεπεράσει το 30%, η κατάσταση δεν θα είναι αναστρέψιμη η κυβέρνηση μπολσονάρο αντί να συνεχίσει το σχέδιο για τη βιώσιμη διαχείριση που υπάρχει από το 2014, ενθάρρυνε την υπερεκμετάλλευση της γης και κλείνει τα μάτια μπροστά στην καταστροφή σε αυτό το πλαίσιο η συμφωνία ευρωπαϊκής ένωσης μερκοσουρ μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την προστασία των δασών του αμαζονίου. είναι μια συμφωνία δίκαιου εμπορίου είναι μια συμφωνία συνδεδεμένη με τη συμφωνία του παρισιού και στην πραγματικότητα νουθετεί τη βραζιλία να αναδασώσει δώδεκα εκατομμύρια εκτάρια. πυρκαγιές δυστυχώς στον αμαζόνιο είχαμε πολλά χρόνια τώρα όμως τώρα τουλάχιστον έχουμε ένα μέσο πίεσης και όποιος παραβιάζει τη συμφωνία του παρισιού πρέπει να παραβιάζει και τη συμφωνία μερκοσουρ. μέτρα πίεσης δεν έχουμε όμως ούτε για τη σιβηρία ούτε για την αφρική ούτε για την ινδονησία. χρειαζόμαστε μια συνολική πρόταση βιώσιμης διαχείρισης των δασών και εργαλεία για να την προωθήσουμε εκτός ευρωπαϊκής ένωσης. αντί να εξαντλούν συνάδελφοι της Γκουε την ευαισθησία τους Πρόεδρος Διακόπτη, ευχαριστώ κυρία Σπυράκη. Για ένα λεπτό κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι τελευταίε εβδομάδε ο κόσμο παρατηρούσε με φρίκι τεράστιε πυρκαγιέ ε, που έκαψαν πάρα πολύ μεγάλε εκτάσει ε, τη Αλάσκα, τη Ελλάδα, ε, του Αμαζονίου κλπ. Με το ιστορικό ανευπροηγουμένου αλλαγή του κλίματο και αποδάσωση σε επίπεδα που δεν έχουμε δει προηγουμένω, Λοιπόν, τελικά οι πνεύμονες της γης γεμίζουν με καπνό. Δηλαδή, από η ανάγκη για το κλίμα προχωρούν μια καταστροφή του κλίματος και χρειάζεται καλύτερη ανταπόντηση από φτηνά πολιτικά παιχνίδια στο Twitter ο κόσμος. Δηλαδή, το όλο σύστημα είναι λαθασμένο. Ε, ο τρόπος που ζούμε, οι λαϊκιστικές πολιτικές που ακολουθούνται έχουν φρικτές συνέπειες για τη ζωή και την υγεία των παιδιών και των παιδιών μας και των παιδιών αυτών. Ο τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε φυσικού πόρου στον πλανήτη είναι κάτι που δεν είναι βιώσιμο. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρο ε, να πάρουμε σκληρέ αποφάσει που απαιτούνται. Το κάναμε με τα πλαστικά, καταφέραμε να περάσουμε απαγόρευση για μερικά από τα χειρότερα προϊόντα, προχωρήσουμε πιο πέρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ηγηθεί αυτού. Όταν η Κρέτα Αντών Μπερκέ είχε τη φωνή τη γωνιά τη ε, και, και μα ζήτησε να πανικοβληθούμε, και τώρα εξαρτάται από εμά αν θα πανικοβληθούμε πέφτοντα πάνω στον τοίχο ή θα πανικοβληθούμε αναλαμβάνοντα δράση. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ κύριε Μετσόλα. Για ένα μισό λεπτό η κυρία Ευγέν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Αμαστονία είναι ολέθρια. Η μάστιγα της αποψήλωσης όμως είναι παγκόσμια. Δεν αφορά μόνο την Αμαζονία. Για παράδειγμα από τον Ιούλιο η Ινδονησία φλέγεται επίσης ε, σε μια αφόρητη σιωπή μέσα και δεν μπορούμε να τα πολεμήσουμε αυτά μόνο με εμπορικές συμφωνίες, αυτή τη μαζική αποψήλωση. Και ακόμα λιγότερο αν δεν έχουν δεσμευτικά μέτρα οι συμφωνίες, όπως το Μερκοσούρ. Ας διευρύνουμε τη συζήτηση. Χρειάζονται χρόνια για να καταλήξουμε σε μια εμπορική συμφωνία που να εφαρμοστεί. Τώρα όμως χρειάζεται πήγουσα δράση. αναπτυξιακή βοήθεια είναι πιο αποτελεσματικός μοχλός βράχη πρόθεσμα και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα ως μέτρο πίεσης προς τα κράτη που εθελοτυφλούν ε, στην αποψήλωση. Τέλος, θα ήθελα να έχω μια σκέψη για τους αγρότες που δεν έχουν ε, άλλη επιλογή δυστυχώς παρά να επεκτείνουν τις καλλιέργειές τους στο δάσος. Θα πρέπει οι ενάρετες πρακτικές να αμείβουν σωστά τους ε, αγρότες. Ευχαριστώ κύριε Εύγαν. Και τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Βάρμπορν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πέρσι το καλοκαίρι είδαμε ε, τεράστιες πυρκαγιές στην Σουηδία και η ε, υποστήριξη των κρατών μελών ήταν πολύτιμη. 139 πυροσβέστες έστειλε η Πολωνία όπως ε, και οι δασικέ πυρκαγιέ σε όλο τον κόσμο ήταν μεγάλο πρόβλημα και για τους ανθρώπους και για τα ζώα και για, τα, και για τη φύση. Και γι' αυτό συμπάσχω με τους ε, Βραζιλιάνους. Αλλά ε, δεν βλέπω να υπάρχει ε, καμία κίνηση για να σταματήσει το εμπόριο με την Σουηδία επειδή είχαμε πυρκαγιές. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι λάθος, όπως ζητάει η αριστερά, να εκμεταλλευτούν ε, αυτή την τραγική καταστροφή για να σταματήσει το ε, ελεύθερο εμπόριο με τη Βραζιλία και το Μερκοσούρ. Να το πω σαφώς ότι μπλοκάρισμα της συμφωνίας Μερκοσούρ δεν θα σβήσει τις φωτιές στον Αμαζόνιο ούτε θα βελτιώσει το κλίμα. Αντιθέτως, η συμφωνία αυτή δεσμεύει τη Βραζιλία και τις άλλες χώρες ε, να εφαρμόσουν τους στόχους του Παρισιού και να έχουν βιώσιμη γεωργία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την, ε, το εμπόριο ως κίνητρο. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε ευημερία, ανάπτυξη ε, και να έχουμε πιο φθηνές υπηρεσίες και αγαθά. Γι' αυτό καλώ τα, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και όλους τους συναδέλφους εδώ πέρα να ε, συμβάλλουν σε μια όσο γίνεται πιο γρήγορη επικύρωση της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ε, ε, συνάδελφε. Ε, περνάμε στην στην διαδικασία Catch the Eye. Όπως είπε η Αντιπρόεδρος Χάουταλα, έχουμε τρεις φορές περισσότερες επανεβάσεις από ό,τι προβλέπουμε. Παρακαλώ. Άρια Σετσαβερία. Πρόεδρε, Επίτροπε Βέλα, θα αρχίσω με κάποια απλά γεγονότα. Το δάσος του Αμαζονίου παράγει 20% του παγκόσμιου εξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Πάνω από εκατομμύριο αυτόχθονες κινδυνεύουν. Ε, δεκαετίες και φωτιές εκεί που αποψηλώνουν. Έχουν αυξηθεί κατά 85% οι πυρκαγιές, είπε ο Μπολσονάρο. Ο Αμαζόνιος δεν είναι η μόνη περιφέρεια που καταστρέφεται δεν υπάρχουν ε, κανονικές φωτιές απλές. Ε, θα αυξηθεί γρήγορα η παγκόσμια θερμοκρασία του πλανήτη, θα καταστραφεί η βιοπικιλότητα και η ζωή των αυτοχθόνων μέσα στο δάσος. Και εμείς τι κάνουμε όσο φλέγεται και καταστρέφεται εκ βάθρων. Καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και βλέπουμε έντρομοι τον πλανήτη να φλέγεται. Όχι, θα πρέπει να δράσουμε. Χτες κιόλας. Ε, ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η στρατηγική που έχετε τώρα εδώ, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύει τα δάση και να αντιμετωπίζει τις δασικές πυρκαγιές, τι κάνετε, πώς μπορούμε να δράσουμε και με χρήματα για να βοηθήσουμε να ελεγχθούν αυτές οι πυρκαγιές και τελικά να κατασβεστούν. Ευχαριστώ, συνάδελφε Άγγιου Σαλίμπα. Έγινε μια μικρή παρεξήγηση. Θα σα είχα δώσει το λόγο, αλλά αργότερα έλεγα ότι ο συνάδελφο Άρια Ετσιβερία είχε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ, χωρίς καμιά αφιβολία είναι το καλύτερο εργαλείο που έχουμε για την προστασία των δασών του Αμαζονίου. Αν θέλει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ηγέτης παγκοσμίω στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκρίνει τη Συμφωνία με το Μερκοσούρ. Η προστασία του δάσου στον Αμαζόνιο είναι κάτι που οφείλουμε να κάνουμε όλοι. Όπω και σε άλλα δάση, στην Αφρική, ε, Αμερική και στην Ασία. Έχουμε διάφορου στόχου, ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, του ΟΗΕ. Θέλω να εξάρω τη συμφωνία στην πόλη Λετήσια στην Κολομβία μεταξύ 7 κρατών. Κολομβία, Περού, ε, η σημερινός Βολιβία και Βραζιλία ε, και άλλες δύο. Ο πρόεδρος Μακρόν όμως δεν είχε την κατάλληλη στάση στο τελευταίο G7 για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. 20 ε, χρόνια ε, σκληρών διαπραγματεύσεων μεσολάβησαν για το Μερκοσούρ. Είναι ευκαιρία η συμφωνία αυτή, όχι μόνο εμπορική, αλλά και περιβαλλοντική. Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Άρια Σετσεβερία και τώρα η κυρία ε, Ιώβεβα. Sorry. Ευχαριστώ. Εδώ ακούμε να λέγεται ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει το παράδειγμα στην καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο. Και ότι είμαστε βασικό παράγον πάνω σε αυτό. Εντάξει, μπορεί να ισχύει αυτό. Εξίσου αληθεύει όμω ότι από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κινείται μόνη τη. Η αλλαγή του κλίματο είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε για την επίλυσή του. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητούμε μεν, αλλά να δραστηριοποιηθούμε δε. Τώρα, τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να ακυρώσουν τη συμφωνία του Μερκοσούρ, δεν θα πρέπει απλώς να βλέπουμε την καταστροφή στην περιοχή του Αμαζονίου, αλλά πρέπει να δράσουμε, να μην παρατηρούμε. Να μην λέμε απλώ λόγια. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η φύση. Και ήρθε η ώρα να αλλάξουμε κι εμεί. Σαν λαοί. Αν δεν αλλάξουμε, ε, θα είναι επικίνδυνο για όλου. Ευχαριστώ κυρία Γιώβεβα. Η κυρία Τζόνς. Ευχαριστώ. Καμιά φορά ένα θέμα την χάνει τη δημόσια προσοχή, διότι αποκρισταλώνει ένα περιπλοκότατο ζήτημα με έναν τρόπο που όλοι το αισθανόμαστε και το κατανοούμε. Και οι πυρκαγιέ στον Αμαζόνιο είναι τέτοιο παράδειγμα. Δεν είναι οι μόνε πυρκαγιέ πράγματι. Χρειάζεται να βάλουμε περισσότερα δέντρα, να φυτέψουμε στην Ευρώπη. Αλλά η επικέντρωση στι πυρκαγιέ του Αμαζονίου πραγματικά στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα. Βλέπουμε τα προβλήματα. Οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται για τη μοίρα του Αμαζονίου. Μας ενδιαφέρει η κρίση, μας ενδιαφέρει αυτή η ποικιλότητα και η ζωή των αυτοχθόνων πληθυσμών που απειλούνται. Κανείς δεν είναι νησί, είμαστε όλοι αλληλένδετοι. Οι επιλογές μας εδώ στην Ευρώπη, η κατανάλωση, η εμπορική πολιτική έχουν μια επιρροή και αλλού στον κόσμο. Όπω και πολλοί άλλοι, και εγώ φοβούμαι τι συνέπειε που θα έχει η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ. Ανησυχώ ότι στενά οικονομικά ωφέλη τελικά θα αφήσουν εκτό τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντο. Θα τα γνωρίσουν αυτά. Δεν με διαβεβαιώνουν καθόλου οι σχετισμοί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάποιο τρόπο θα έχει περισσότερη ισχύ τώρα και πίεση όσον αφορά το περιβάλλον, την προστασία του και τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά την υπογραφή τη Εμπορική Συμφωνία Μερκοσούρ. Κοιτάξτε το ιστορικό μέχρι τώρα. Οχτώ χρόνια μα πήρε να ξεκινήσουμε την επιβολή των μέτρων στην Κορέα. Όσοι έχει η Συμφωνία του Μερκοσούρ είναι μόνο καρό και εδώ ξαναδιακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσόνς. Η κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ας μην το παίζουμε αθώοι. Συζητούμε την αποψήλωση των δασών από το 2017 όταν εδώ υπέβαλα την έκθεσή μου για το θέμα και θετήθηκε η έκθεσή μου από το Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος Μπολσονάρο σημαίνει καταστροφή για τα δάση. Το ξέρουμε εδώ και ένα χρόνο αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της εμπορικής της πολιτικής αποτελεί τμήμα του προβλήματος. Μην υποκρινόμεθα ότι συγκλονιστήκαμε. Έπρεπε να διερωτηθούμε γιατί περιμέναμε τόσο καιρό για ένα σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποψήρωσης των δασών. Και γιατί δεν υπήρξε ψήφισμα που είναι απόρρια αυτή τη συζήτηση που διεξάγεται τώρα. Απλώ κάνουμε ότι ενδιαφερόμαστε. Και αυτό είναι όλο. Ας αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα τα δάση καταστρέφονται. Και δάσο σημαίνει ζωή. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστροφή. Α σταματήσουμε τώρα τη ρητορική, να σταματήσουμε την αποδάσωση, α ας στηρίξουμε τα δάση και α γίνουμε ένα μέρο τη λύση. Σα ευχαριστώ, κυρία Κονέτσνα. Η κυρία Βάγκ, παρακαλώ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, είμαστε εδώ σήμερα ενωμένοι από αριστερά προς τα δεξιά για να καταδικάσουμε τι δραματικέ πυρκαγιέ στον Αμαζόνιο. Ας σταματήσουμε ε, τους λιγούς και τα κλάματα και α δράσουμε. Μπορεί να κάνει κάτι συγκεκριμένο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εμπορικά μέσα για να ασκήσουμε πίεση και πάντα χρησιμοποιήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη συμφωνία του Μερκοσούρ και επιμένει ότι δεν μειώνει οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές αυτή η συμφωνία και ότι η αρχή της πρόληψης εξασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες Μερκοσούρ μπορούν να συνεχίσουν να προστατεύουν το περιβάλλον. Τώρα μπορούμε να δούμε πόσο ο Μπολσονάρο τηρεί τις υποσχέσεις του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι είναι νομικά δεσμευμένος να σέβεται τη βιοπικιλότητα και το περιβάλλον. Λοιπόν, ας αναστείλουμε την ισχύ της, της συμφωνίας αυτής μέχρι σταματήσουν οι πυρκαγιές και μέχρι ότου έχουν διαρευνηθεί τα αίτια ε, των πυρκαγιών. Αν αυτό το κάψιμο του μεγαλύτερου δάσου στην περιοχή αυτή του κόσμου δεν είναι αρκετά σοβαρό, τι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στείλει αυτή την εμπορική συμφωνία και άμα δεν γίνεται σεβαστό το κεφάλαιο περιβιωσιμότητα. Σα ευχαριστώ, κύριε Άβραμ. Τέλος, Κύριο Κέρερ, παρακαλώ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι ε, η συζήτηση αυτή δεν θα πρέπει να γίνει ιδεολογική συζήτηση αριστερά-δεξιά. Ε, ναι, είναι ε, δεξιό ο Μπολσονάρο, είναι όμω αριστερό ο, ο Μοράλε. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε με ηθικού όρου πώ εμπορευόμαστε και πώ προστατεύουμε τον πλανήτη. Και αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται να είναι κερδοφόρο το να καίει κανείς ε, τα δάση στον Αμαζόνιο ή αλλού στον κόσμο για να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση στις αγορές. Συνεχίζουμε να εισάγουμε σόγια και καφέ ε, από τα μέρη αυτά του κόσμου ε, και αν συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό θα συνεχίσουν να καίνε τα δάση του Αμαζονίου η συμφωνία ε, Μερκοσούρ αν ε, επικυρωθεί σημαίνει ότι η Ευρώπη θα καταστρέψει την συμφωνία του Παρισιού και όχι η άλλη πλευρά. Θα πρέπει να επιμείνουμε ε, σε κάποια ελάχιστα πρότυπα προτού υπογράψουμε οποιαδήποτε συμφωνία Μερκοσούρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κέλεχερ. Ολοκληρώθηκε έτσι η διαδικασία Catch the Eye. Ο Επίτροπος ο κύριος Βέλα, παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι Συμφωνούμε ότι τα τροπικά δάση είναι πολύ σημαντικός πόρος του πλανήτη και η συζήτηση έδειξε ότι είναι πολύ ανησυχητικές οι πυρκαγιές ε, στον Αμαζόνιο ε, και όλα αυτά ε, ενώ βλέπουμε καταστροφικές πυρκαγιές και σε άλλα μέρη του κόσμου. Πολλοί είπαν και συμφωνώ απολύτω ότι πρέπει να ανησυχούμε και να αντιμετωπίσουμε όλε τι δασικέ πυρκαγιέ ε, οπουδήποτε, είτε στην Αγγόλα, την ε, Σιβηρία, την Αρκτική, την Ανταρκτική, την Ευρώπη, την ε, Αμερική. Οι φωτιές αυτές δείχνουν πόσο επίγονοι είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ε, προστατεύσουμε το κλίμα. Τα δάση είναι απαραίτητα στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος. Ε, η προστασία των δασών αποτελεί σημαντικό ε, στοιχείο της ευθύνης μας να τηρήσουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι περισσότεροι ομιλητές μίλησαν για τη Συμφωνία Μερκοσούρ στο κεφάλαιο ε, εμπόριο και ανάπτυξη της συμφωνίας αυτής και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες Μερκοσούρ συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας δέχτηκαν μια ρητή δέσμευση να εφαρμόσουν τους στόχους του Παρισιού. Και η δέσμευση της Βραζιλίας ε, περιλαμβάνει δεσμεύσεις ε, για αναδάσωση και προστασία των δασών. Επίσης ε, θα πρέπει οι ε, έμποροι κρέατος από τη Βραζιλία να μην ε, πολλούν κρέας από τις περιοχές όπου έχουν καταστραφεί τα δάση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί τμήμα μιας γενικής συμφωνίας σύνδεσης που περιλαμβάνει κεφάλαιο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ρήτρες σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος και του κλίματος. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει έτσι επιπλέον εργαλεία στη διάθεσή του, ε, ώστε ε, να μπορέσουμε να φέρουμε πιο κοντά τους πολίτες και τις αγορές μας. Πολλοί ανέφεραν ότι οι δεσμεύσεις υπάρχουν ήδη, θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ περιλαμβάνει εκτενές κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιέχει δεσμευτικές ε, ρήτρες ε, για την προστασία του περιβάλλοντος, ε, την αλλαγή του κλίματος συμπεριλαμβανομένης και της δέσμευτης να τηρηθούν οι στόχοι του Παρισιού. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις αυτές. Εάν η μία πλευρά δεν ε, τηρήσει την ε, συμφωνία, μπορούμε να προσφύγουμε ε, στον μηχανισμό, στο σχετικό μηχανισμό και πιστεύουμε και περιμένουμε θα φροντίσουμε κυρίως η Βραζιλία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού που συμπεριλαμβάνει δέσμευση από τη Βραζιλία μέχρι το 2025 να μειώσει τις εκπομπές της ε, κατά 37% ε, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005. Συμπεριλαμβάνει επίσης ένα σχέδιο δράσης να σταματήσει η παράνομη αποψήλωση των δασών ε, στην Βραζιλία. Επίσης υπάρχει δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουμε κατά τουλάχιστον 40% τις εκπομπές μας μέχρι το 2030. Κάποιοι ευρωβουλευτέ ε, είπαν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τη ζήτηση ε, όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που σχετίζονται με την καταστροφή των δασών. Ένα νομοθετικό πλαίσιο για τέτοια προϊόντα αποτελεί στοιχείο κλειδί. Είναι απαραίτητο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει εσωτερικές ρυθμίσεις ε, που απαγορεύουν, για παράδειγμα, την ε, χρήση παράνομης εξηλία. Στόχος ε, της οδηγίας αυτής είναι να σταματήσει η παράνομη αποψήλωση των δασών και να ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές για τα προϊόντα που αγοράζουν όσον αφορά οποιαδήποτε μελλοντικά μέτρα που να σχετίζονται με προϊόντα ε, από περιοχές που έχουν καταστραφεί τα δάση, θα ήθελα να σας ε, παραπέμψω στα μέτρα που έχουμε ήδη ανακοινώσει, ε, όπως είναι η ενίσχυση προτύπων και προγραμμάτων πιστοποίησης, ώστε να ε, εντοπίζονται και να προωθούνται ε, προϊόντα που δεν, περιέχονται, που δεν προέρχονται από ε, παράνομα αποψηλωμένες περιοχές. Επίσης θέλουμε να αυξήσουμε την διαφάνεια και να μειώσουμε τον κίνδυνο εισαγωγής προϊόντων που σχετίζονται με την υποβάθμιση ή καταστροφή των δασών. Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε ε, την προστασία των δασών ε, και στην ε, εταιρική ευθύνη. Θέλουμε να προωθήσουμε την υπεύθυνη συμπεριφορά στις επιχειρήσεις και θέλουμε να έχουμε και συνομιλίες ανάμεσα στις κυβερνήσεις, τις ΜΚΟ, λιανοπολιτές κλπ. Θα ήθελα τέλος να θυμίσω σε όλους ότι το τελικό νομικό κείμενο της Συμφωνίας Σύνδεσης και οι εμπορικές πτυχές του θα υποβληθούν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έγκριση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Βέλα και τώρα για να κλείσει τη συζήτηση το λόγο έχει εξ ονόματος του Συμβουλίου Υπουργός του Πουράινεν. Mr. President, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κυρίε και κύριοι. Για να κλείσουμε, θέλω να σα ευχαριστήσω. Ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση. Είναι κατεπήγον το θέμα που μα αφορά όλου. Όλοι πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τα δάση μα. Πρέπει να βελτιώσουμε τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω επ' αυτού και να συνεχίσουμε την προσπάθεια ούτω ώστε να τιμήσουμε τι διεθνεί μα υποχρεώσει. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε στη συμφωνία την εμπορική του Μερκοσούρ. Η εμπορική συμφωνία με τις χώρες των Μερκοσούρ έχει ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη που ανταποκρίνεται σε ύψιστες προδιαγραφές συγκρίσιμες με αυτές σε άλλες σύγχρονες συμφωνίες. Βασική υπόθεση ποια είναι ότι η αύξηση του εμπορίου δεν θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα εις βάρος του περιβάλλοντος ή των συνθήκων εργασίας. Αντιθέτως μάλιστα, θα πρέπει να προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη. Η Συμφωνία Μερκοσούρ περιέχει συγκεκριμένο άρθρο περί αλλαγής του κλίματος και δεσμεύονται συμβαλόμενα μέρη να εφαρμόσουν τη Συμφωνία των Παρισίων πράγματι και αποτελεσματικά. Υπάρχουν και προβλέψεις για την καταπολέμηση της αποδάσωσης τη απερίμωση των δασών. Όπω συμβαίνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συζητή στο Συμβούλιο όσον αφορά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Μερκοσούρ είναι σε μια πρώιμη φάση ακόμα. Επαρκή χρόνο απαιτείται για μια πλήρη διεξοδική ανάλυση τη συμφωνία αυτή θα είναι σημαντικό και για τα δύο θεσμικά όργανα να διεξαχθεί ειλικρινή συζήτηση επί της συμφωνίας βάσει στοιχείων. Επίσης θα ήθελα να σημειώσω ότι αν... ανοιχτή εμπορική πολιτική με βάση κανόνες και αξίες που θα βασίζεται στη βιωσιμότητα και στην κάλυψη όλων αποτελεί προτεραιότητα για τη Φιλανδική Προεδρία. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε στην κατεπίγουσα ανάγκη για δράση για το κλίμα. Η ώρα για να δράσουμε είναι τώρα για το κλίμα και όχι αργότερα. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επηρεάσει άλλους μέσω παραδείγματος. Γι' αυτό είναι κρισίμου σημασία να συμφωνήσουμε επί φιλοδόξου στόχου για την ουδετερότητα την κλιματολογική στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2050 και να συμφωνήσουμε το ταχύτερο δυνατόν επ' αυτού. Κυρίε και κύριοι, πρέπει να διαφυλάξουμε τα δάση του Αμαζονίου για τι επόμενε γενιέ. Τεράστια ζημιά έχει γίνει μέχρι τώρα και ε, την καταγγέλλω αυτή. Αλλά θα πρέπει να προλάβουμε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δάση μας και στον Αμαζόνιο και αλλού. Διότι πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές μας. Η αποψήλωση των δασών είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Με πολλές περιπλοκες πτυχές. Γι' αυτό το λόγο, συνεργασία εντός του Συμβουλίου είναι βασικό τμήμα επιτυχούς εργασίας. Κάτι έτσι σημαντικότερο είναι η συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών ε, θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό το λόγο είμαστε όλοι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ νέου για την ενεργό συμμετοχή σας και για την ε, προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. πολύ, ε, κυρία Υπουργέ. Έτσι κλείνει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Λίγα λεπτά διάλειμμα.